I wish you all good afternoon and please be seated as soon as... Καλησπέρα σας, παρακαλώ καθίστε το συντομότερο δυνατόν. Έχει περάσει η ώρα και θα ήθελα να αρχίσουμε παρότι λείπουν αρκετά μέλη της Επιτροπής. Όμως οι αναφέροντες είναι εδώ και είναι έτοιμοι να λάβουν το λόγο, ας αρχίσουμε λοιπόν. Επίσης να πω πως χαίρομαι ότι η κυρία Μαγκίνες, η αντιπρόεδρος του Κοινοβουλίου, βρίσκεται εδώ οι αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου έχουν λάβει πρόσκληση και έχουν απαντήσει με επιστολή που περιλαμβάνει πάρα πολλές λεπτομέρειες. Σας συστήνω να τη διαβάσετε. Ας αρχίσουμε λοιπόν. Θα δώσω το λόγο στη Μαρή Καπόποβα και την Ελίσα Μπέτα Πόποβα και την Σαμπίνα Κοριό Μακνίου. Νομίζω είστε όλες εδώ. Πολύ ωραία. Καλώς ήρθατε. Με χαρά μου σας δίνω λοιπόν το λόγο. Παρακαλώ. Good afternoon. Uh, Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Ελίσσα Πέτα Ποπόβα. Καταρχάς θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία αυτή. Για την ευκαιρία που μου δίνετε. Πραγματικά σημαίνει πολλά για μένα το ότι βρίσκομαι εδώ. Καταρχάς, θα ήθελα να αναφερθώ στην κόρη μου, την Μέγαν, η οποία υιοθετήθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο, χωρίς τη συγκατάθεσή μου. Δεν έχω δει την κόρη μου από τις 8 Αυγούστου του 2013. Πήραν την κόρη μου από μένα με λόγους πιθανή μελλοντική συναισθηματική κακοποίηση και επίσης με έκριναν ως ακατάλληλο γονέα. λόγω ανάρμοστης σεξουαλικής συμπεριφοράς. Το άτομο που έκανε τη διάγνωση αυτή δεν είχε τα κατάλληλα προσόντα για να το πράξει. Μισό λεπτό, λέει η πρόεδρος. Υπάρχει πρόβλημα με τη μετάφραση γιατί έχετε σταματήσει και σταματάτε συχνά. Όχι, λέει αναφέρουσα, ακούω τα ακουστικά. Να τα βγάλετε τότε, λέει η πρόεδρος. Θα είστε πολύ πιο άνετα έτσι. Προσπαθήστε λοιπόν ξανά. Πάρτε όσο χρόνο χρειάζεστε. Εμείς είμαστε εδώ για να σας ακούσουμε. Δικιά σας είναι η μέρα σήμερα. Οι διερμηνείς βρίσκονται εδώ για να μεταδώσουν το μήνυμά σας σε όλες τις γλώσσες. Ζητώ συγγνώμη. Τελευταία λοιπόν επαφή με την κόρη μου είχα το 2013. Λίγο πριν υιοθετηθεί. Κατέβαλα κάθε προσπάθεια για να αποδείξω στις ε, υπηρεσίες ότι είμαι κατάλληλος γονέας κατάλληλος δεμόνας έκανα ό,τι χρειαζόταν, όλα τα σεμινάρια που χρειαζόταν έτσι ώστε να είμαι ασφαλής γονέας. Όμως τίποτα από όλα αυτά δεν έλαβε υπόψη το δικαστήριο. Ήταν σαν να μην έκανα τίποτα απολύτως. Δεν νομίζω πως η μεταχείρισή μου ήταν δίκαιη από τις αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου και πραγματικά αναγνωρίζω ότι σε όλη αυτή τη διαδικασία έκανα λάθη, όμως δεν πιστεύω πως μου αξίζει μια τέτοια ισόβια ποινή εξαιτία ενός λάθους. Πιστεύω πως μου αξίζει μια ευκαιρία να είμαι με την κόρη μου, θέλω να είμαι με την κόρη μου. Και θα ήθελα επίσης να πω ότι κατά την άποψή μου οι Βρετανικές αρχές έχουν κίνητρα στο να παίρνουν αλλοδαπά παιδιά έτσι και δεν είμαι η μόνη που το σκέφτεται αυτό διότι οι αλλοδαποί ξέρουν πώς λειτουργεί ο Βρετανικός νόμος και είναι πολύ εύκολο στόχος λοιπόν κάποιος ξένος εκεί. Το δικαστήριο χρησιμοποίησε όλα όσα είπα εναντίον μου. Αυτή την αίσθηση έχω. Παρά το γεγονό ότι είπα και θετικά πράγματα, ότι του έδειξα πω αγαπώ την κόρη μου, θέλω την κόρη μου. Όλα αυτά δεν τα έλαβε υπόψη του το δικαστήριο. Και σήμερα βρίσκομαι ενώπιόν σα διότι ξέρω πως αξίζει στην κόρη μου να βρίσκεται μαζί μου με τη βιολογική τη μητέρα. Αυτό είναι το καλύτερο για εκείνη και δεν χρειάζεται, δεν πρέπει να βρίσκεται με ξένους ανθρώπους. Την τελευταία φορά που την είδα ήταν πάρα πολύ ταραγμένη και δεν την έχω δει ποτέ έτσι. Και όλε οι φωτογραφίε που έχω από την κόρη μου τη δείχνουν χαμογελαστή και ποτέ πραγματικά δεν την έχω δει τόσο ταραγμένη. Δεν πιστεύω ότι μου δόθη ποτέ το δικαίωμα σε μια δίκαιη δίκη. Το δικαίωμά μου στην οικογενειακή ζωή. Μου έχουν κλείσει όλες τις πόρτες στο να βιώσω το ρόλο του γονέα. Και υπάρχει και ένα πόρισμα σύμφωνα με το οποίο αποτελώ κίνδυνο και στο χώρο εργασίας μόνο και μόνο επειδή μου πήραν την κόρη μου και αυτό πιστεύω πως είναι άδικο. Επίσης, μου αφαιρέθηκε και η γονική συγκατάθεση από τον δικαστή Πλάμστεντ σε ένα δικαστήριο της κομιτείας στην οποία ζούσα. Δεν μου ανέφεραν κανένα λόγο παρά μόνο το ότι στη Μέγαν αξίζει μια καλύτερη ζωή χωρίς κίνδυνο ψυχικής βλάβης. Αποφάσισαν λοιπόν στο δικαστήριο ότι είναι καλό να μου αφαιρέσουν τη γονική συγκατάθεση. Και ποτέ δεν έλαβαν υπόψη του τα δικαιώματα του παιδιού. Και τίποτα από όλα όσα έκαναν η κοινωνική λειτουργία και οι κοινωνικές υπηρεσίες δεν ήταν δίκαιο. Δεν θέλω να επαναλαμβάνομαι, αλλά πραγματικά αυτό περιγράφει αυτό που αισθάνομαι. Και ως Ευρωπαία πιστεύω πως ε, πραγματικά δεν με μεταχειρίστηκαν ως τέτοια. Πού είναι τα δικαιώματά μου, πού είναι τα δικαιώματα του παιδιού μου. Δεν έχω επαφή με το παιδί μου και πραγματικά έχει δικαίωμα να ξέρει ποια είναι, ποια είναι η ταυτότητά της. Δεν ξέρει ποια είναι η μητέρα της ποιοι είναι οι παππούδες της, οι γιαγιάδες της, οι συγγενείς της. Δεν ξέρει τίποτα από όλα αυτά. Γιατί λοιπόν να διαγράψουν έτσι την ταυτότητά της με μία μονοκοπηλιά. Σήμερα αυτό που ζητώ από εσάς είναι να μου πείτε τι μπορώ να κάνω, ποιες είναι οι εναλλακτικέ λύσεις που έχω έτσι ώστε να είμαι ξανά μαζί με την κόρη μου. Ποιο θα πρέπει να είναι το επόμενό μου βήμα. Ε, το μόνο που θέλω να ξέρω είναι ότι είναι ζωντανή και είναι καλά Πήγα στα Βρετανικά δικαστήρια, στα πρωτοδικεία, τα εφετεία. Έκανα έφεση, άσκησε έφεση σε όλες τις δικαστικές αποφάσεις, όμως τίποτα δεν έλαβαν υπόψη από όλα όσα έκανα. Και πραγματικά πιστεύω πως εθελοτυφλούσαν. Και πράγματι, στη ζωή γίνονται λάθη, όμως οι άνθρωποι αλλάζουν και τους αξίζει να έχουν μια ευκαιρία. Ζητώ συγγνώμη γιατί μου είναι δύσκολο να μιλήσω. Μου λείπει τόσο πολύ η Μέγαν και το μόνο που θέλω είναι να είμαι μαζί της. Γι' αυτό ήρθα εδώ σήμερα. Και εάν το επόμενο μου βήμα είναι το δικαστήριο, τότε εκεί θα πάω. Όμως δεν θα το βάλω κάτω μέχρι να είμαι πάλι με την κόρη μου. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ που έχετε το θάρρος να ε, ταξιδέψετε από τόσο μακριά και να έρθετε εδώ να μοιραστείτε τη ζωή, τη ιστορία σας μαζί μας και είναι πραγματικά πάρα πολύ συγκινητική ε, και φαντάζομαι όλοι οι συνάδελφοι θα έχουν συγκινηθεί το ίδιο. Σας ευχαριστώ και πάλι για το θάρρος σας. Στρέφομαι προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τη Μάργα Τσιούτ. Έχετε το λόγο. Thank you, Chair. Good afternoon, everyone. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Πόποβα που μοιράστηκε μαζί μας την ιστορία της. Κατανοούμε πόσο ταραγμένοι είστε. Είναι πραγματικά σπαραξικάρδια και η υπόθεση είναι πάρα πολύ περίπλοκο το θέμα και πιστεύω πως κανένας δεν μπορεί να βγει κερδισμένο σε τέτοιες περιπτώσεις. Τώρα, ας μην ξεχνάμε ότι στα πλαίσια των δικαιωμάτων του παιδιού οι εθνικές αρχές, στην περίπτωση αυτή οι αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου, έχουν καθήκον τους στην προστασία των παιδιών και έχουν καθήκον να αναλάβουν δράση όταν υπάρχει κίνδυνος προς το παιδί αυτό. Γι' αυτό λοιπόν να το έχουμε αυτό υπόψη. Δεν ήμασταν στα δικαστήρια για τη συγκεκριμένη υπόθεση και δεν είμαστε εδώ για να συζητήσουμε τι έκαναν τα δικαστήρια του Ηνωμένου Βασιλείου. Κοιτάξαμε όμως πολύ προσεκτικά όλο το υλικό που μας εστάλει και σας ακούσαμε με πολύ μεγάλη προσοχή. Θα δώσω το λόγο σε λίγο στην συνάδελφό μου, Γιωχανά Σουντίνσκα, από την Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας της Γενικής Διεύθυνσης Justice, η οποία θα μας εξηγήσει τον κανονισμό Βρυξέλλες 2 όσον αφορά την γονική ευθύνη. Από όλα όσα ακούσαμε για την υπόθεση αυτή, αλλά και από άλλες υποθέσεις επιμέλειας, και υιοθεσία χωρί γονική συνένεση και έχοντα λάβει υπόψη το γεγονό ότι υπάρχει υιοθεσία με γονική συνένεση και υιοθεσία όπου η γονική συνένεση έχει αφαιρεθεί, Έχουμε λάβει λοιπόν όλα αυτά υπόψη και έχουμε συντάξει ένα έγγραφο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την προστασία των παιδιών και τη ε, συναφή υπηρεσία ιδιαίτερα σε συνοριακέ περιπτώσει προσπαθώντας να βρούμε δυνατότητες για διασυνοριακή συνεργασία. Επίσης, τα τελευταία δύο χρόνια εργαζόμαστε στον χώρο της δικαιοσύνης και στην ανάπτυξη δυνατοτήτων, κατάρτιση δικαστικών και άλλων λειτουργών, ιδιαίτερα για τα δικαιώματα του παιδιού και τα δικαιώματα του παιδιού να κάνει τη φωνή του ακουστή. Έχουμε λοιπόν πολλούς τομείς στους οποίους εργαζόμαστε. Θα δώσω τώρα το λόγο στην ε, Ιωάννα, η οποία θα σας ενημερώσει σχετικά. Σας ευχαριστώ πολύ. Επιτρέψτε μου να πω δύο λόγια για την υπόθεση αυτή ε, σε σχέση με τον κανονισμό Βρυξέλλες 2. Έχουμε ακούσει και άλλες φορές στην Επιτροπή παρόμοιες υποθέσεις και όπως είπε και η συνάδελφός μου, οι συνθήκες είναι πραγματικά ε, κάτι που μας ε, θλίβει. Προσπαθήσαμε να δούμε πόσο μπορούμε να το συνδέσουμε με τον κανονισμό για την ε, γονική ευθύνη στα πλαίσια του Βρυξέλλες 2. Η ίδια η απόφαση της υιοθεσία δεν καλύπτεται από τον κανονισμό Βρυξέλλες 2. Είναι ευθύνη των κρατών μελών να ασχολούνται με περιπτώσεις υιοθεσία τέκνων. Όμως, ο κανονισμός θα έπρεπε να διευκολύνει τη συνολική συνεργασία, ιδιαίτερα τη δικαστική διασυνοριακή συνεργασία. Κοιτάξαμε τον φάκελο που κατέθεσε η αναφέρουσα, αναλύσαμε τα στοιχεία και όπως είπα η απόφαση για υιοθεσία ήταν μία απόφαση στα πλαίσια του ουσιαστικού οικογενειακού δικαίου, κάτι το οποίο δεν καλύπτει ο κανονισμός Βρυξέλλες 2. Δεν μπορέσαμε λοιπόν να βρούμε κάποια σύνδεση έτσι ώστε να διερευνήσουμε το θέμα περαιτέρω. Και πιστεύω πως η αναφέρουσα έχει μια πολύ σωστή θέση. Δεν διαφωνεί. Και είπατε ότι παραβιάστηκε το θεμελιώδες δικαίωμα του παιδιού σας και αναφέρετε επίσης ότι προσφύγατε στο δικαστήριο του Στρασβούργου. Πολύ καλά κάνατε, διότι περιπτώσεις όπως η δική σας δεν καλύπτονται από τον κανονισμό, όμως καλύπτονται από τον ε, χάρτη των ε, θεμελιωδών δικαιωμάτων και χρειάζεται να εξεταστούν από το δικαστήριο του Στρασβούργου. Για περίπτωση πιθανής παραβίασης των θεμελιωδών δικαιωμάτων του παιδιού σας. Το δεύτερο που ήθελα να πω είναι ότι διάβασα με μεγάλη προσοχή την όλη διαδικασία στην οποία υποβληθήκατε τους τελευταίους μήνες, τα τελευταία χρόνια. Και πρέπει να πω ότι το έχουμε λάβει σοβαρά υπόψη αυτό, διότι διαπιστώσαμε ότι οι εθνικές αρχές δεν ακολουθούν τους ε, μηχανισμούς συνεργασίας που προβλέπονται από τον κανονισμό. Υπάρχουν κάποια κενά και ένα από αυτά τα κενά το ε, υπογραμμίζεται στην αναφορά σας όταν αναφέρεστε στην ε, διαδικασία λήψης αποδεικτικών στοιχείων στη Βουλγαρία. Οφείλω να πω όμως ότι αυτό αυτά δεν καλύπτονται από τον κανονισμό Βρυξέλλες 2. Δεν καταφέραμε λοιπόν να εντοπίσουμε ε, και να διαπιστώσουμε όντως μια παράβαση. Όμως, σημειώσαμε τη διαδικασία που ακολουθήθηκε από το δικαστήριο στις αποφάσεις του. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να ρωτήσω αν παρίσταται κάποιο από τη βουλγαρική πρεσβεία. Όχι. Ναι. Εδώ, ακριβώ. Θέλετε να λάβετε το λόγο από αυτού. Όχι, Δυστυχώ δεν είμαι σε θέση να σχολιάσω, αλλά θα διαβιβάσω όλες τι πληροφορίε ε, στους ε, μου. Άκουσα ότι είναι εδώ και η γιαγιά, η κυρία Μαρίκα Πόποβα, επίσης αναφέρουσα Θέλετε να λάβετε το λόγο για μια σύντομη παρουσίαση. Σχόλιο. Έχετε τίποτα να προσθέσετε στα όσα μόλις είπε η κόρη σας. Παρακαλώ, μην διστάσετε. I think you are more comfortable to sit down. Καθίστε, αν θέλετε καθίστε, δεν χρειάζεται να είστε όρθια. Μία στιγμή, περιμένω. Ακούτε, σας ακούω, αλλά καλύτερα να κάθεστε, γιατί θα λειτουργεί και καλύτερα το μικρόφωνο για να ακούγεται καλύτερα ο ήχος για τους διερμηνείς. Αλλιώς δεν ακούμε τίποτα. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ που με καλέσατε και μου δίνετε την ευκαιρία να μιλήσω. Θα Να σας παρουσιάσω τις απόψεις μου. Και ε, όπως είπατε εγώ είμαι η γιαγιά της Μέγκαν. Και εγώ έχω κάποια θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα όπως το δικαίωμα στο να μπορώ να προσφέρω τη φροντίδα μου στην Μεγκάν. Ουδέποτε η, η οικογένειά μας συνεφώνησε να υιοθετηθεί από αγνώστους η Μεγκάν. Τελείως αγνώστους ούτε από που κρατάει σκούφια τους δεν ξέρουμε. Και αυτό το οποίο θέλουμε είναι η Μέγκαν να μην χάσει την της. Είναι βουλγάρα, αυτό είναι αδιαμφισβήτητο. Είναι θεμελιώδες δικαίωμα το οποίο και παραβιάστηκε διότι ε, ε, μας, μας απέρριψαν λόγω κάποιας αξιολόγησης από κάποια κοινωνική λειτουργό. Ουδέποτε ενημερώθηκαν οι βουλγαρικές αρμόδιες αρχές. Δεν μάθανε ότι πήγε εκεί αυτή η κοινωνική λειτουργός και συνέταξε τη σχετική αναφορά ή έκθεση. Ούτε υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας ενημερώθηκαν σε σχέση με την προστασία του παιδιού, ούτε ενημερώθηκε ούτε η δημοτική αρχή τη γενετηρά μα. Δεν υπήρξε ποτέ συνεργασία των δύο κρατών μελών. Επομένω, εδώ υπάρχει ένα στοιχείο υπερ-εθνικό, διασυνοριακό. Ε, υπάρχουν, ε, είναι δύο οι άδικοι πάντοτε σε αυτέ τι διαφορέ. Ε, θα πρέπει επομένω εδώ να αναχωρεί η περίπτωση εφαρμογή του διεθνού δικαίου. Социален доклад, който тя състави от 200 страници, имам преведени 23 страници. Κοινωνική προνοία, κοινωνική αρρωγή, έκανε και εκείνη μια αξιολόγηση. 23 σελίδες μόνο από όλη την έκθεση μεταφραστηκαν και οι δικαστικές αρχές του Κέιμπριτζ μας αγνόησαν, μας αγνόησαν γιατί δεν είχαμε διερμηνέα και εμεί αγνοούμε ακόμα και την ε, Βρετανική νομοθεσία και σε αυτές τις ε, μεταφρασμένες 23 σελίδες διάβασα ότι εγώ και ο σύζυγός μου δεν μπορούμε να φροντίσουμε την εγγονή μας. Οι δε ε, αρμόδιες βουλευτικές αρχές έχουν συντάξει δύο εκθέσεις και εκεί λέει ότι εγώ, η γιαγιά και ο σύζυγός μου, ο παππούς μπορούμε να φροντίσουμε την εγγονή. Και κάθε φορά ενώπιον παντός δικαστηρίου προσπαθώ να ακουστώ για να υποβάλω τις παρατηρήσεις μου. Στο Λονδίνο δεν με άφησαν να παραστώ και να ακουστώ. Ούτε υπάρχει κάποιο ρύθμιση άμεσης επαφής, προσωπικής επαφής με την ε, εγγονή. Δεν δικαιούμαι να την δω. Θα ήθελα πολλά να σας πω, αλλά ξέρω ότι πιέζει ο χρόνος. Και αυτό το που ήθελα να σας πω είναι ότι και εγώ και ο σύζυγος, δηλαδή ε, ο παππούς και η γιαγιά της Μεγκάν, έχουμε παράσχει ενώπιον του Βρετανικού Δικαστηρίου. Έχουμε εγγυηθεί ότι μπορούμε να φροντίσουμε την εγγονή μας. Τα πάντα να κάνουμε για αυτήν. Οικογενειακό περιβάλλον, προστασία, όλα αναφέρονται σε αυτό το έγγραφο, αυτήν την εγγύηση, εγγύηση όπως ονομάζεται στο Βρετανικό Δίκαιο. Έχουμε προσαράγει επομένω όλα τα στοιχεία σε κάθε βαθμό δικαιοδοσίας και στο εφετείο. Αλλά μας αγνόησαν. Δεν ακουστήκαμε. Παραβιάστηκαν θεμελιώδη δικαιώματα. Δεν μπορώ να δω την εγγονή μου και θεωρήθηκε ότι αυτό είναι ένα επιχείρημα το εξή, ότι δεν μπορώ να φροντίσω την εγγονή. Εγώ θέλω να γυρίσει στη Βουλγαρία, να μας γνωρίσει η εγγονή μου, να γνωρίσει την πατρίδα της, τη μητρική της γλώσσα να μάθει. Δεν μπορώ να πούμε ότι είναι Βρετανή, γιατί η μητέρα της είναι Βουλγάρα. Έτσι είναι με τα παιδιά. Θα πρέπει κανείς να συνυπολογίσει τα δικαιώματα και του πατέρα και της μητέρας του παιδιού. Ούτε μπορεί να γνωρίσει κανείς τον παππού και τη γιαγιά. Δεν είναι δυνατόν όλοι αυτοί να πάνε στην άκρη και να παραδίδεται το παιδί σε αγνώστους. Ευχαριστούμε που μας διαθέσετε εδώ το χρόνο για να, μιλήσουμε και έχω το εξή ερώτημα. Πού να πάμε, σε ποιον απευθυνθούμε για να μπορέσει να έρθει σπίτι η Μέγκαν. Δεν γνωρίζω τον κόσμο, το, τους ανθρώπους αυτούς τους οποίους κατέληξε. Μου λένε ότι είναι Άγγλοι. Μα τι, τι Άγγλοι είναι, ποιοι είναι αυτοί οι Άγγλοι. Ζω και ο σύζυγός μου και εγώ ζούμε. Αν μπορούμε να τη φροντίσουμε και οπότε θα ε, μπορούμε να παράσχουμε και φορολογική δήλωση για τα εισοδήματά μας. Έχω ένα γιο 10, μια ε, κόρη 17. Είμαστε υπεύθυνοι. Ήδη έχω μεγαλώσει τρία παιδιά. Ε, δεν καταλαβαίνω. Δεν καταλαβαίνω, σας λέω. Και άλλη μία ερώτηση, παρακαλώ. Γνωρίζετε τα πραγματικά περιστατικά και διαβάσατε τα σχετικά έγγραφα. Οπότε θα ήθελα να μου πείτε ποιος, ποιος θα μας επιστρέψει την Μέγκαν. Υπάρχει ε, κάποιο όργανο, κάποιος φορέας που να προστατεύει τα δικαιώματα των βιολογικών γονέων. Ποιος, ποιος δικαιούται να λάβει μια δικαστική απόφαση και να ακυρώσει την απόφαση του Βρετανικού Δικαστηρίου. Τώρα το τελευταίο που θέλω να σας πω είναι ότι ο γιος πριν από λίγες μέρες με ρώτησε «Μαμά, γιατί δεν φέρνουμε εδώ την Μέγκα, δεν την έχω δει ποτέ, θέλω να τη δω, να παίξω μαζί της, θέλω να απολαύσω τη ζωή μαζί της». Τι να το απαντήσω? Τι να του πω, τι μπορώ να του πω, μα πραγματικά να του πω ότι το, το, διάφορα δικαστήρια τα Βρετανικά δεν θέλησαν να μας δώσουν την ε, Μέγαν γιατί δεν μας εμπιστεύονται μα έχουμε σπίτι έχουμε ήδη φτιάξει ένα δωμάτιο για την Μέγαν έχουμε ανακαινήσει το σπίτι έχουμε κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να μπορέσει να έρθει η εγγονή μας είναι Βουλγάρα κανείς δεν μπορεί να το αμφισβητήσει αυτό είναι μισή Βουλγάρα μισή Βρετανίδα. Δεν είναι δυνατόν να μας παίρνουν, μας ε, απαγάγουν έτσι την, ε, την εγγονία και να τη δίνουν σε άγνωστους. Ποιος μπορεί, πέστε μου, να ακυρώσει την απόφαση του Βρετανικού Δικαστηρίου. Δεν ξέρω αν είναι ευχαριστημένοι, δεν ξέρω εάν μεγαλώνει σωστά, συναισθηματικά, ψυχολογικά. Μα τι να κάνω, παρατηθώ. Έχω εγγονή, αλλά δεν ξέρω τι γίνεται. Αυτό είναι φυσιολογικό, μα αυτό το οποίο ξέρουν ότι όλα αυτά τα μέτρα σε σχέση με την υιοθεσία τη εγγονή από αγνώστους δεν είναι προ το συμφέρον τη. Ούτε προ το δικό μα συμφέρον. Θα πρέπει να μας γνωρίσει η εγγονή τις ρίζες, τις, ε, τους παππούδες, γιαγιάδες, τη, τη γλώσσα. Μα ποιος πρόκειται να την ε, παρηγορήσει όταν συνειδητοποιήσει ότι έγινε υποκείμενο ή αντικείμενο τέλο πάντων υιοθεσία. Μα ε, έχει μητέρα και πατέρα. Και ότι υιοθετήθηκε από κάποιου ξένου. Αλλοδαπού. Ποιο θα την παρηγορήσει. Και σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Απόποβα για την παρέμβασή σας. Όπως είπα προηγουμένως, είναι πραγματικά πολύ συγκινητικό, είναι σπαραξικάρδια αυτό που μας λέτε. Αλλά κοιτάξτε, εμείς δεν είμαστε δικαστήριο, ούτε πρόκειται να δικάσουμε κανένα. Βρισκόμαστε εδώ για να προσπαθήσουμε να εξετάσουμε την αναφορά και την κατάσταση. Γι' αυτό θα ανοίξει τώρα η συζήτηση, θα μπορέσουν να μιλήσουν οι συνάδελφοι και να δούμε αν υπάρχει τρόπος να βρεθεί μια ε, εξοδικαστική ε, λύση για την κατάσταση αυτή. Θα ήθελα να δώσω πρώτα το λόγο στον κύριο ε, Ζάντεφ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Πολλές φορές επικρίνεται η Βουλγαρία ε, επί τη βάση του δικαϊκού της συστήματος, αλλά μένα με εξέπληξε το βρετανικό σύστημα, βρετανική δικαιοσύνη από ε, την υπόθεση αυτή της Μέγκαν. Είπαμε ότι πρέπει να υπάρχει δικαστική συνεργασία, αναβαθμισμένη, αμοιβή αρρωγή κλπ. κλπ. Όμω, εν προκειμένου, ο δικαστή δεν ετήρησε αυτά τα οποία προβλέπει ο κανονισμό, η συμφωνία υπαριθμών 2 των Βρυξελών τέλο πάντων, δεν ήρθε σε επαφή με τι αρμόδιε δικέ μα αρχέ. Και ήρθε η ο για να περισυλλέξει στοιχεία για την υπόθεση. Ήρθε, αλλά δεν ενημέρωσε τις αρμόδιες βουλγαρικές αρχές, δηλαδή το Υπουργείο Δικαιοσύνης της Βουλγαρίας. Το μέλλον του παιδιού αγνοήθηκε. Επομένως δεν τηρήθηκε το κοινωτικό δίκαιο, το οποίο κατησχύει της εθνικής νομοθεσίας. Εμείς εδώ νομοθετούμε κάθε μέρα. Και βέβαια το πιο πολύτιμο πράγμα είναι τα παιδιά. Άρα θα πρέπει εδώ να κατησχύσει και να εφαρμοστεί το κοινωτικό δίκαιο και έτσι να μπορούμε να καλύψουμε τα αιτήματα αυτή τη βουλγαρική οικογένεια. Ευχαριστώ πολύ, με κυρία Γκαμπρίελ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω εγώ ότι αφού άκουσα ε, τις αναφέρουσες και τη συγκεκριμένη περίπτωση και ε, πρέπει να πω ότι ως μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν μπορούμε να μείνουμε απαθείς και ψυχροί απέναντι σε αυτή την ανθρώπινη τραγωδία. Θα πρέπει όμως να αναρωτηθούμε, όπως έκανε μόλις ο συνάδελφος Ράντεφ, εμείς ως Ευρωπαίοι νομοθέτες θα πρέπει να φροντίσουμε κυρίως να γίνεται σεβαστό και να ε, εφαρμόζεται το ευρωπαϊκό δίκαιο. Γι' αυτό θα πρέπει να επιμείνουμε για να ε, ε, εφαρμόζεται από τα ε, Βρετανικά δικαστήρια ο κανονισμός Βρυξέλλες 2.1. Υπάρχουν υπηρεσίες κοινωνικές αρμόδιες στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά δεν μπορώ να παραβλέψω αυτά που μας ανέφεραν οι κυρίες. Θα πρέπει να προβληματιστούμε και να αναρωτηθούμε. Είναι άραγε δίκαιο να αφαιρεί κανείς ε, την κυδαιμονία, την επιμέλεια από μία μητέρα που ε, μιλάει ε, καλά αγγλικά, που έχει εκπαίδευση, μόρφωση αντίστοιχη, ώστε να μπορεί να φροντίζει σωστά το παιδί της. Σε ό,τι αφορά τη γιαγιά επίσης και το παππού της. Δεν μπορούμε να παραβλέψουμε το γεγονός ότι υπάρχει διακριτική μεταρρύθμιση. Και βασίζονται όλα αυτά σε μία και μόνη ε, συνάντηση με τη γιαγιά, η οποία πάντα υποστηρίζει την κόρη της, η οποία είναι πάρα πολύ αξιοπρεπής, ε, ε, χέρι υψηλού κύρου ε, στην κοινότητά τη, Έχει και άλλα δύο παιδιά που είναι καλοί μαθητέ και τα πάνε πολύ καλά. Το προξενείο στο Λονδίνο ε, ασχολείται και φροντίζει τα ε, δικαιώματα των Βουλγάρων πολιτών στην Αλοδαπή. Δυστυχώ σήμερα δεν μπόρεσε να παρευρεθεί κανεί, αλλά καλό θα ήταν να γνωρίζει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι οι εκπρόσωποι του, προξενείου, του βουλγαρικού προξενείου στο Λονδίνο απευθύνθηκαν στο δικαστήριο και στον ε, λόγο δικαστή Βλουμστέτ για να του θέσουν υπόψη τις ισχύουσες ε, διατάξεις του κανονισμού Βρυξέλλες 2. Οι κοινωνικές υπηρεσίες τα γνωρίζουν αυτά στο Ηνωμένο Βασίλειο και πώς ε, προέβησαν στις αποφάσεις αυτές που έλαβαν χωρίς να ενημερώσουν τις αρμόδιες αρχές του βουλγαρικού προκειμένου Υπουργείου Δικαιοσύνης το δικαστήριο στο Κέμπριτζ πώς μπορεί να αποφασίσει για μια έρευνα ε, σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς να ζητήσει δικαστική συνδρομή ή χωρίς να ενημερώσει τις ερμόδιες αρχές. Ε, θα πρέπει ε, λοιπόν όλες οι αρμόδιες αρχές σε κάθε κράτος μέλος να σέβονται την κοινοτική νομοθεσία. Θέλω να ακούσω όμως την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τι μέσα ε, έχουμε για να μπορέσουμε να ελέγξουμε και να παρακολουθούμε την κατάσταση αυτή και να γίνεται σεβαστή πάντα η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Θα ήθελα επίσης να καλέσω και να παρακαλέσω τους συναδέλφους της Επιτροπής Αναφορών να ε, βοηθήσουν. Ξέρουμε ότι έσχατη λύση είναι ε, το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Στρασβούργο. Εμείς έχουμε κάποια δυνατότητα να επηρεάσουμε τα πράγματα ώστε να επιταχυνθεί η εκδίκαση εκεί. Η κυρία Πρόεδρος και η κυρία Μαγκίνες ενδεχομένως θα μπορούσατε από κοινού να στείλετε μία επιστολή στο δικαστήριο επισυνάπτοντας το αποτέλεσμα της σημερινής συνεδρίασης για την αναφορά αυτή. Χρειάζεται γραπτή υποστήριξη όλων όσοι σήμερα βρισκόμαστε εδώ. Υποστηρίζουμε όλη αυτή την αναφορά που τόσο πολύ μας συνεκίνησε. Και πάλι, πέρα από τα συναισθηματικά και το θυμικό, θα πρέπει πάνω απ' όλα να επικεντρωθούμε στο πιο σημαντικό που είναι ο σεβασμός της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. Ευχαριστώ. Thank you very much, Mr. Malinov. Ευχαριστώ κύριε Μάλενοφ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Σας ευχαριστώ. Τι να σας πω, ε, είναι πολύ σημαντικά φορτισμένη η περίπτωση. Βέβαια ούτε εμείς μπορούμε να κάνουμε τον νομικό γιατί είμαστε πολιτικοί, είμαστε μέλη της Επιτροπής των Αναφορών, αλλά θεωρώ ότι ε, δικαίως, δικαίως το μας πληρώνει η συγκίνηση γιατί δεν μπορούμε να παραμείνουμε αδιάφοροι. Δεν είναι δυνατόν. Θα πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν ε, ούτως ώστε να βοηθήσουμε σε την υπόθεση με τέτοιες υιοθεσίες. Θα πρέπει να είμαστε ειλικρινείς και τώρα δεν πρόκειται για υιοθεσία. Πρόκειται για υιοθεσία δια της βίας. Δεν πρόκειται μόνο για αυτή την περίπτωση, γιατί υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις που θα πρέπει να τις έχουμε υπόψη, οι οποίες είναι δυνατόν να ε, ξανασυμβούν. Εδώ πέρα έχουμε απέναντί μας ε, μια πρακτική του Ηνωμένου Βασιλείου. Είναι πάρα πολύ επιλήψιμη, αμφισβητήσιμη. Το θέμα δεν είναι ε, εάν είναι σύνομη ή όχι. Πρόκειται για μια πρακτική η οποία σοβεί εκεί, συνηθίζεται εκεί και στην συγκεκριμένη περίπτωση θύμα είναι ένα, ένας ανήλικος βούλγαρος ένα παιδί από τη Βουλγαρία. Οπότε θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με τα δικαιώματα των ανηλίκων. Γιατί υπάρχει η Διεθνή Σύμβαση και δεν είναι δυνατόν να επιτρέπουμε ε, να, να αρπάζεται το παιδί δια της βίας από τους γονείς του εκτός εάν έχουμε περίπτωση άσκησης βίας από πλευράς των ε, γονείων. Εάν δεν βρίσκονται εις διάσταση οι γονείς τότε θα πρέπει να σκεφτούμε για τον τόπο κατοικίας του παιδιού. Ε, αυτά όλα αναφέρονται στη Διεθνή Σύμβαση για τους Ανηλίκους οπότε δεν υπάρχει εδώ πρόβλημα για την επιμέλεια και για την κυδαιμονία. Έχουμε και τους δύο γονείς. Το πατέρας δεν έχει καμία διεκδίκηση επί του ανηλίκου, οπότε μπορούμε να παραδώσουμε τον ανήλικο, το παιδί, στην μητέρα και το παιδί να επιστρέψει στην Βουλγαρία. Γι' αυτό μας πλημμυρίζουν, ε, ε, μας πλημμυρίζει η συγκίνηση. Οι Βρετανικές αρχές ε, πέδειξαν μια συμπεριφορά απαράδεκτη διάβασα και διάβασα όλα τα στοιχεία και ξανά και ξανά και δεν κατάλαβα γιατί δεν δικαιούνται οι παππούδες να αναλάβουν το εγγόνι τους. Σε ένα σωρό μέρη στην ε, Βουλγαρία υπάρχει αγανάκτηση για αυτό το θέμα. Δεν, όμως, δεν πρόκειται εδώ για μεμονωμένη περίπτωση. Είναι μια περίπτωση που αποδεικνύει ότι υπάρχει δυσμενής διάκριση και δεν είναι δυνατόν ε, εδώ να υπάρχει τέτοια αντιμετώπιση. Τέλος πάντων θα πρέπει να αποφανθεί το Ευρωπαϊκό Διαστήριο ξεκάθαρα, ε, θα πρέπει ένα θεσμικό όργανο να αποφασίσει και να αποφασίσει ολομόντια και σας προτείνω το εξή. να μείνει ανοιχτή η αναφορά και επίσης θεωρώ ότι οφείλουμε να ζητήσουμε γνωμοδότηση από την Νομική Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτή έχει την ε, αρμοδιότητα όσον αφορά την ε, γονική μέρημνα, την επιμέλεια από πλευρά των γονέων. Έτσι, να επιταχύνουμε τη διαδικασία ενώπιον της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Στρασβούργο. Για μένα ήταν πάρα πολύ δύσκολο να φουγκραστώ αυτήν την τόσο στεναχωρημένη μητέρα. που προσπαθεί να εξηγήσει για το κατά πόσο εμπίπτη στο πεδίο εφαρμογή του κανονισμού Βρυξέλλες 2. Ε, αυτό είναι θλιβερό. Ναι, είμαι καινούριο εδώ σε αυτή την επιτροπή, αλλά ξέρω ότι υπάρχει κανονισμό ο οποίο πρέπει να εφαρμοστεί. Υπάρχουν πήγοντε υποθέσει και κατεπίγουσε υποθέσει. Και πιέζει ο χρόνο. Σήμερα η Μέγαν ζει μαζί με την οικογένεια που την υιοθέτησε. Είναι καλή οικογένεια, αλλά το θέμα είναι τι θα γίνει με τη μητέρα της, τι θα γίνει με τους παππούδες της. Είναι πολύ θλιβερή αυτή η υπόθεση. Θα πρέπει κάτι να κάνουμε για να βοηθήσουμε την οικογένεια. Και θα πρέπει να το πράξουμε με τρόπο αντικειμενικό. Δεν είναι εδώ απλή περίπτωση της μενούς διάκρισης. Είναι κάτι πολύ χειρότερο. Γι' αυτό και ε, οδήγησε σε τόση αγράγηση από πλευράς ε, τόσων Βουλγαρών. Αλλά κάτι θα πρέπει να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Χιλιάδες, χιλιάδες Βουλγάρων. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να δώσω τώρα το λόγο στην κυρία Μαρκίνη. Thank you very much. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Βρίσκομαι εδώ με το ρόλο της διαμεσολαβήτριας για τα παιδιά και όχι της Αντιπροέδρου του Κοινοβουλίου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή Αναφορών για την άψογη συνεργασία που έχει με το γραφείο μου. Πιστεύω πως ε, μπορούμε να κάνουμε καλύτερη δουλειά όταν συνεργαζόμαστε και καλά. Σας ευχαριστώ λοιπόν. Τώρα, μερικά γενικότερα σχόλια προτού να στη συγκεκριμένη περίπτωση. Καταρχάς, θα ήθελα να ευχαριστήσω τις αναφέρουσε, διότι πραγματικά ήρθαν εδώ για να μας παρουσιάσουν κάτι το οποίο ματήρα πολύ δύσκολε συνθήκες. Να σας πω ότι δεν είμαστε δικαστήριο, όπως πολύ σωστά είπατε. Ήμουν και εγώ στην Επιτροπή Αναφοράς και ξέρω αυτό που κάνουμε είναι να δίνουμε ένα βήμα στους ανθρώπους για να εκφράσουν τα προβλήματά τους και να προσπαθούμε να τους βοηθήσουμε. Έπειτα, θα ήθελα να αναφερθώ στις ε, ε, συναισθηματικές στοιχείες της περίπτωσης αυτής, διότι είμαι και εγώ μητέρα και πραγματικά μπορώ να φανταστώ πώς θα αισθανόμουν αν κάποιος μου έπαιρνε το παιδί και το έδινε για υιοθεσία. Καταλαβαίνω, θα ρω, και την ε, μητέρα του παιδιού και τη γιαγιά του παιδιού που είναι μαζί μας σήμερα. Ωστόσο, Κάθε κράτος μέλος έχει το δικό του σύστημα προστασίας των παιδιών. Και δεν μπορούμε εδώ να αποφασίσουμε για τις ε, επιμέρους συνθήκες, τις συγκεκριμένες συνθήκες αυτής της περίπτωσης, διότι δεν έχουμε όλα τα στοιχεία και δεν είμαστε κοινωνική λειτουργή. Δεν μπορούμε επομένω να κρίνουμε. Ας φύγουμε λοιπόν από τις επιμέρους λεπτομέρειες και ας επικεντρωθούμε στα γενικότερα στοιχεία αυτό που χρειάζεται να καταλάβουμε είναι το ότι πρέπει να αναζητήσουμε αν τα κράτη-μέλη πραγματικά ασχολούνται με το συμφέρον του παιδιού και αν το παιδί απολαμβάνει τα θεμελιώδη δικαιώματά του. Είναι ουσιαστικό σε όλα αυτά να δούμε ότι το οικογενειακό δίκαιο σε πολλά κράτη-μέλη δεν είναι κάτι το πολύ γνωστό, είναι κάπως μυστικό. Στη δική μου χώρα, για παράδειγμα, οι πληροφορίες που λαμβάνουμε δεν είναι για τις συγκεκριμένες υποθέσεις, αλλά για τις τάσεις που επικρατούν στο οικογενειακό δίκαιο. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να λάβουν υπόψη τους όσοι ασχολούνται με τη χάραξη πολιτικής. Θα ήθελα από προσωπικό ενδιαφέρον να παρακολουθήσω το θέμα και να συνεργαστώ και με εσάς και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με το δίκτυο των Ευρωπαίων Διαμεσολαβητών, διότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό που προτείνω βέβαια είναι αρκετά μακροπρόθεσμο και δεν θα λύσει το συγκεκριμένο πρόβλημα αμέσως. Ας έρθω όμως σε αυτό. Πιστεύω πως όποια οικογένεια αναγκάζεται να φτάσει μέχρι το σημείο του να φτάσει μπροστά σε μια κοινοβουλευτική επιτροπή θέλει πραγματικά να επανασυνδεθεί με το παιδί της. Αυτό λοιπόν που θα πρότεινα, όπως πρότεινε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι κάτι που θεωρώ την καλύτερη λύση και η συνάδελφος κυρία Μαρία Γκάμπριελ έκανε και αυτή αναφορά στο ίδιο πράγμα. Είναι η προσφυγή στο δικαστήριο του Στρασβούργου. Δεν ξέρω τι θα γίνει με το χρονοδιάγραμμα και αν θα μπορέσει να ακουστεί η υπόθεση αυτή. Όμως πιστεύω πως είναι η σωστή λύση. Αυτό που μας δυσκολεύει εμάς ως ευρωβουλευτές είναι ότι οι αρχές, όπως είπα, δεν ασχολούνται με συγκεκριμένες υποθέσεις. Δεν θα μας ενημερώσουν για τη συγκεκριμένη υπόθεση. Η συγκεκριμένη όμως υπόθεση δεν φέρνει στο φως αυτό το θέμα των υιοθεσιών χωρίς την γονική συνένεση. Αλλά, και εδώ είναι η δυσκολία, εκτός από τη συγκεκριμένη υπόθεση και τις συγκεκριμένες συνθήκες που την διέπουν, πρέπει να δούμε την ευρωπαϊκή διάσταση, να δούμε τι γίνεται στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση στον συγκεκριμένο τομέα και πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Σας υπόσχομαι λοιπόν ότι θα μελετήσω πάρα πολύ προσεκτικά τη συγκεκριμένη περίπτωση και πιστεύω πραγματικά πως ε, η οικογένεια Απόποβα έχει κάνει κάτι που θα ωφελήσει πάρα πολύ τις οικογένειες στην Ευρωπή που βρίσκονται σε παρόμοια θέση. Θα διερευνήσουμε λοιπόν τι μπορούμε να κάνουμε σε παρόμοιες περιπτώσεις στην Ένωση. Και όπως είπα, δεν πιστεύω πως η απάντηση είναι η Βρυξέλλες 2. Δυστυχώς, διότι εδώ πρόκειται για θέμα υιοθεσία. Και Μάλιστα, εφόσον οι επαφές με τις βουλγαρικές αρχές δεν ήταν αυτές που επιθυμούσαμε. Όμως, επαναλαμβάνω, πραγματικά συμπονώ του, τις αναφέρουσες και τις ε, καταλαβαίνω. Είναι μια περίπτωση μιας οικογένειας που υιοθέτησε τώρα ένα παιδί. Σίγουρα θα έχει κάποια σχέση μαζί του, αλλά από την άλλη έχουμε και μια οικογένεια που έχασε ένα παιδί. Δεν ξέρω τι θα γίνει στο μέλλον, αλλά ελπίζω το παιδί να είναι καλά και να απολαμβάνει τη φροντίδα που του αξίζει. Και επίσης να πω ότι το θέμα δεν είναι βουλγαρικό ή βρετανικό, είναι ευρωπαϊκό. Και σίγουρα η δική μου αρμοδιότητα είναι να ασχολούμαι με τέτοια ζητήματα. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που μου δώσατε τη δυνατότητα να μιλήσω και συγγνώμη αν μακρηγόρησα. Προτίθεμαι να έχω πολύ στενές επαφές και συνεργασία με εσάς και να σας ενημερώνω για οποιαδήποτε εξέλιξη και άλλα σχετικά ζητήματα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Πραγματικά είναι πολύ ενδιαφέρουσα η συγκεκριμένη περίπτωση και είναι πολύ ενδιαφέρον το ζήτημα και διασυνοριακά. Και δεν είναι η μόνη αναφορά αυτή. Υπάρχουν πάρα πολλές αναφορές από πολλά κράτη-μέλη που έχουν παρόμοιο θέμα. Όμως, όπως είπατε και εσείς πολύ σωστά, αυτό που κάνει η οικογένεια εδώ είναι να μας επιστήσει την προσοχή σε κάτι που συμβαίνει συστηματικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό λοιπόν φυσικά και θα ωφελήσει η υπόθεση αυτή και πολλές άλλες οικογένειες στην Ευρώπη. Εγώ προσωπικά πιστεύω πως εδώ υπάρχει σοβαρότατο θέμα διακρίσεων και Συμφωνώ με τον συνάδελφο Μάλινοβ. Τώρα έχουν ζητήσει πολύ το λόγο. Πάβελ, αρχίζεις. Ευχαριστώ πολύ. Θα είμαι σύντομος. Έχω δύο παρατηρήσεις να κάνω. Δεν είναι η πρώτη φορά που έρχεται κάποιος εδώ για να συζητήσει ένα τέτοιο θέμα που αφορά κάτι δεν πάει καλά εδώ με τις Βρετανικές αρχές. Κάτι βρωμάει στη Μεγάλη Βρετανία και νομίζω πως υπάρχει κάποιο λάθος στο όλο σύστημα εκεί. Γι' αυτό λοιπόν συμφωνώ με όλους τους συναδέλφους που είπαν ότι πρέπει να παραμείνει αναφορά ανοιχτή και προτείνω να στείλουμε μια επιστολή στις Βρετανικές αρχές όπου θα τους παρακαλούμε να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα το συντομότερο δυνατόν μαζί με τις βουλγαρικές αρχές. Και προτείνω τους ε, βούλγαρους, στους βούλγαρους συναδέλφους να είναι πιο ενεργοί στο θέμα αυτό. Πραγματικά πιστεύω πως είναι ενθαρρυντικό το ότι βρίσκονται πολλοί συνάδελφοι από τη Βουλγαρία εδώ, συνάδελφοι που δεν είναι συνέχεια παρόντες στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Αναφορών. Αντίθετα, με σοκάρει το γεγονός ότι δεν υπάρχει ούτε ένας Βρετανός Ευρωβουλευτής. Και είχαν ενημερωθεί όλοι. Πίτερ, έχει το λόγο. Ο Πέτερ Γιάρε, ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Μια συμπλήρωση μόνο ακούστηκε επανειλημμένα, το είπατε και εσείς, ότι είναι σπάραξη κάρδια. Όποιος έχει παιδιά είναι και παππούς και όλα τα καταλαβαίνει όλα αυτά και τα νιώθει. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους, ιδιαίτερα εσάς, ε, που ε, δεχτήκατε την αναφορά αυτή και με την ταχεία διαδικασία, την επίγουσα. Σωστά είπε ο προλαλή Το θέμα είναι τι γίνεται με το δικαίωμα του παιδιού. Όταν λένε ότι ε, ε, τηρήθηκαν όλα σε πλήρη νομιμότητα και οι διαδικασίες ήταν εντάξει, αλλά έχει και το παιδί δικαιώματα και θα πρέπει να τα λαμβάνουμε υπόψη. Και σωστά υπόθηκε ότι δεν είναι η μοναδική τώρα αναφορά με τη Μεγάλη ε, Βρετανία. Έχουμε μια ολόκληρη σειρά τέτοια θέματα και τέτοιες αναφορές. Κάποιο πρόβλημα υπάρχει στη Μεγάλη Βρετανία με το δίκαιο υιοθεσία και θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ακούσει και αυτό λέτε ότι είναι αρμόδια τα κράτη-μέλη. Υπάρχει όμως ο κανονισμός ε, Βρυξέλλε 2 και τουλάχιστον εκεί προσφέρεται συνεργασία. Αλλά συνεργασία όταν πρόκειται για παιδιά τι σημαίνει. Ότι θα πρέπει να συμμετέχουν τα ε, αρμόδια κράτη-μέλη ή τα ενεχόμενα κράτη-μέλη των γονέων και να αγωνίζονται να βρούνε την καλύτερη λύση. Όχι το ένα κράτος να κοινοποιεί στο άλλο ότι αποφάσισε και το τρίτο να κανονίζει την πορεία του. Συνεννόηση ή συνεργασία σημαίνει καθόμαστε όλοι μαζί και ε, πρότεινε και η βουλγαρική ε, πρεσβεία στο δικαστήριο να ληφθούν υπόψη και οι γονείς ε, και οι ε, παππούδες, γιατί η μητέρα είναι Βουλγάρα και οι παππούδες είναι Βουλγαροί. Και εγώ είμαι πολιτικός, το λέω ως πολιτικός αυτά, όχι ως νομικός. Ε, το ελάχιστο ε, που θα μπορούσε να κάνει κανείς είναι να μην χρησιμοποιήσει κατευθείαν πυρηνική βόμβα, ας πούμε, υιοθεσία. Υπάρχουν και ενδιάμεσες λύσεις. Υπάρχουν και πιο ελαφρά όπλα από αυτό. Αλλά ε, αποφάσισαν τα Βρετανικά δικαστήρια ε, και κοινοποίησαν στη Βουλγαρία την απόφαση την οποία θα πρέπει να δεχτεί κιόλας. Δεν είναι τρόπος αυτός ε, θα πρέπει να στείλουμε και επιστολές, να το ψάξουμε περισσότερο. Ε, δεν ξέρω οι συνάδελφοι πώς το βλέπουν, αλλά για μένα συνεργασία σημαίνει ότι συνεργάζομαι και όχι απλώς κοινοποιώ αποφάσεις ηλυμένε και τελεσίδικες. Και το γράφει ο νομοθέτης. Πρέπει να συνεργάζεστε. Δεν εννοεί αυτό ο νομοθέτης λοιπόν κοινοποίηση, αλλά συνεργασία και προς όφελος του παιδιού να βρούμε την καλύτερη λύση και όχι να αποφασίσουμε και να το κοινοποιήσουμε στην άλλη χώρα. Φυσικά θα ανοίξει, θα παραμείνει ανοιχτή αυτή η αναφορά. Να στείλουμε τα γράμματα που είπαμε και προς τους Βρετανούς και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να το κοιτάξει λίγο περισσότερο, ε, να δει ποια συνεργασία υπήρξε ή δεν υπήρξε και αυτό που με εξοργίζει εμένα και με ενοχλεί είναι ακριβώς ότι δεν ξέρω αν είναι βρετανική ε, σπεσιαλιτέ, αλλά η υιοθεσία σημαίνει και απόφαση. Το είπε και πολύ σωστά ε, κάποιος προηγουμένως. Έχουμε ένα παιδί σε μια νέα οικογένεια. Δηλαδή, ό,τι και να κάνουμε, πάλι θα το ε, αποσπάσουν από την οικογένεια και θα είναι σπαραξικάρδι αυτό για τη νέα οικογένεια. Τι σημαίνει λοιπόν συνεργασία, το Ιβρυξέλη 2 και σε εμάς τους πολιτικούς γενικά λέμε ότι η πολιτική είναι η τέχνη του εφικτού και αρχίζει από την παρατήρηση της ε, πραγματικότητας. Και αν δεν σ' αρέσει η πραγματικότητα που δεν μας αρέσει σε κανένα, σημαίνει ότι αρχίζει να συζητάς πώς θα την αλλάξεις. Ε, βέβαια αυτό είναι ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και προς το Συμβούλιο. Εμείς θέλουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, θέλουμε την Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια, αλλά όταν πρόκειται για τα δικαιώματα των παιδιών, θα πρέπει να τα λαμβάνουμε και αυτά υπόψη, γιατί εδώ έχουν τελείως ε, γίνει στην άκρη και παραμεληθεί. Thank you, Mrs. Kuneva. Ευχαριστώ, κυρία Κούνεβα, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα μιλήσω βουλγαρικά αυτή τη φορά, ακόμα και αν ε, προσωπώ την Ελλάδα ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα ήθελα να δώσω και εγώ τη γνώμη μου και την υποστήριξή μου σε αυτή τη βουλγαρική οικογένεια η οποία ήρθε να μας εξηγήσει την περίπτωσή της. Αυτή η περίπτωση αφορά όλη την Ευρώπη. Όπως υπόθηκε, δεν είναι μεμονωμένη περίπτωση, είναι συνήθως πρακτική. Έχω διαβάσει μια στατιστική όπου λέγεται ότι η πρακτική αυτή για πρώτη φορά παρατηρήθηκε με τους Τούρκους που ε, ήρθαν μετανάστες στην Ευρώπη για να δουλέψουν. Και μετά ε, αυτό επεκτάθηκε και σε άλλες εθνικότητες και σε άλλους πολίτες. Και λένε οι στατιστικές ότι το 2% των παιδιών που ε, αποσπώνται, που απαγάγονται κυριολεκτικά από τους γονείς τους, δίνονται για υιοθεσία. Ξέρουμε ότι υπάρχει σχετική ευρωπαϊκή νομοθεσία, αλλά Κατά την άποψή μου, αν αυτή είναι ευρωπαϊκή πολιτική θα πρέπει να δούμε τι πάει στραβά. Γιατί κάτι πάει στραβά, έτσι δεν είναι. Αν μπορούν ακόμα τέτοιες πρακτικές να ε, υφίστανται και να εφαρμόζονται στην Ευρώπη. Και επαναλαμβάνω, και ε, ε, είναι αρκετά διαδεδομένη και στις Ηνωμένε Πολιτείε ε, και στην Αυστραλία, αλλά και στην Ευρώπη, στην Νορβηγία, στη Γαλλία και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Πρέπει να δούμε τι λάθος γίνεται για να μην επαναληφθούν τέτοιες ε, περιπτώσεις. Και επίση θα πρέπει να αναβάνουμε υπόψη και τις άλλες καταχρήσεις που έχουμε στη Βουλγαρία. Διότι στη Βουλγαρία παγάγουν παιδιά από τις μανάδες τους και τα δίνουν σε ανάδοχες οικογένειες, οι οποίες ανάδοχες οικογένειες ούτε τα ταΐζουν, ούτε τα αλλάζουν και τα αφήνουν να μεγαλώνουν στους δρόμους. Οι πατεράδες μάλιστα αυτών των οικογενειών των αναδόχων υποτίθεται είναι ε, μεθύστακες που δένουν και τη γυναίκα τους και τα ε, ε, παιδιά αυτά τα καημένα, τα φουκαριάρικα ζουν μέσα στη μιζέρια και στη φτώχεια και στην απόλυτη ένδυα. Αυτό υπάρχει στη Βουλγαρία και ο κόσμος ε, δεν μπορεί να μεγαλώνει σωστά τα παιδιά του. Πολύ, σωστά, πολύ συχνά οι μητέρες πριν ακόμα γεννήσουν ξέρουν ότι δεν θα είναι σε θέση να μεγαλώσει το παιδί τους. 600 λέβα ή 300 ευρώ δίνουν στις μητέρες ως επίδομα τέκνου. Δεν φτάνει αυτό για να μεγαλώσεις ένα παιδί στη Βουλγαρία. Άρα κάτι πάει λάθος, κάτι λάθος έχουμε κάνει στην Ευρώπη, στην ευρωπαϊκή πολιτική για την προστασία των παιδιών. Ε, έριξα μια ματιά στην αλληλογραφία μεταξύ των διαφόρων αρχών ε, στις αναφορές αυτές και απεκόμισα την εντύπωση ότι η γιαγιά είναι μια γυναίκα πάρα πολύ έξυπνη και αξίζει την εμπιστοσύνη μας. Έχει μεγαλώσει τρία παιδιά και αποδεικνύει την ικανότητά της αυτό. Αυτά. Ευχαριστώ για την ε, προσοχή σας. Εγώ ευχαριστώ. Η κυρία Πιτέρα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας σε μια διαφορετική οπτική γωνία του προβλήματος αυτού. Να σας επιστήσω λοιπόν την προσοχή στο ότι εδώ ασχολούμαστε με παραβιάσεις του κανονισμού για τη δικαστική συνεργασία όπου ο πελάτης αναφέρει ότι ορισμένα έγγραφα δεν μεταφράστηκαν στη γλώσσα του. Πιστεύω λοιπόν ότι ανεξάρτητα από όλε αυτέ τι πραγματικά δραματικέ περιγραφέ που ακούμε κάθε φορά που έχουμε τέτοια περίπτωση εδώ, διαφαίνεται και ένα άλλο πρόβλημα. Ότι τα δικαστήρια στη Μεγάλη Βρετανία, γιατί δεν σέβονται τα δικαιώματα των αντιδίκων στις ε, δίκες αυτές. Ίσως θα έπρεπε λοιπόν να ελέγξουμε πώς γίνονται αυτές οι διαδικασίες στα Βρετανικά δικαστήρια. Εάν υπάρχει νομική αρρωγή, διότι εάν δεν έχουν τα οικονομικά μέσα θα πρέπει να έχουν νομική αγαρογή, εάν θα έχουν δυνατότητα μετάφρασης ή διερμηνίας, όπως θα έπρεπε να δικαιούνται όλοι οι πολίτες ενός δημοκρατικού κράτους. Και πιστεύω πως αν κοιτούσαμε εκεί θα μπορούσαμε να καταλάβουμε όλα αυτά που συζητούμε εδώ, διότι Πραγματικά, πολλές φορές οι αποφάσει αυτέ έχω την αίσθηση ότι λαμβάνονται μονόπλευρα. Σας ευχαριστώ πολύ. Πιστεύω πως είχαμε πολύ γόνιμη συζήτηση. Και πραγματικά νομίζω πως διαφαίνεται ένα μοτίβο εδώ. Διότι η μία μετά την άλλη υπόθεση έχει παρόμοια στοιχεία. Τώρα, θα... παρακαλώ, ναι, πάρτε το λόγο, αλλά πολύ σύντομα. Ονομάζομαι Σαμπίν Μακνίλ και εγώ εντόπισα αυτή τη, την περίπτωση, αυτό το σύστημα, το μοτίβο με τις συστηματικές ε, ξαναγκαστικές υιοθεσίες στη Μεγάλη Βρετανία. Να σας πω ότι 4% μόνο των παιδιών που ε, μπαίνουν στο σύστημα αυτό υιοθετούνται και σας διαβεβαιώνω ότι όσα παιδιά καταλήγουν να υιοθετούνται δεν καταλήγουν απαραίτητα σε ωραίες και ευτυχισμένες οικογένειες. Την περασμένη εβδομάδα και αυτή τη εβδομάδα βρέθηκα σε δύο βρετανικά δικαστήρια και πραγματικά ήταν αποκρουστικό αυτό που είδα. Αυτές οι αποφάσεις είναι απαράδεκτες και πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω αυτή τη συμπεριφορά και ιδιαίτερα όταν οι αντίδικοι είναι όπως οι γυναίκα που βρίσκεται δίπλα μου. Έχουν συλλεγεί υπογραφές, πολλές υπογραφές. 5.500 υπογραφές για την περίπτωση αυτή και πραγματικά δεν μπορείτε να φανταστείτε τι γίνεται στη Μεγάλη Βρετανία με αυτές τις υιοθεσίες. Σας ευχαριστώ λοιπόν πολύ που μας ακούσατε. Σας ευχαριστώ και εγώ. Μου είναι πολύ δύσκολο να συνοψίσω τα όσα είπαμε. Σίγουρο όμως είναι ότι η αναφορά αυτή θα παραμείνει ανοιχτή. Και εγώ προσωπικά θα ήθελα να ρωτήσω την Επιτροπή εάν θα μπορούσα σε συνεργασία με την κυρία Μαγκίνες που είναι αντιπρόεδρος για θέματα δικαιωμάτων των παιδιών να αναλάβουμε το θέμα και να έρθουμε σε επαφή με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έτσι ώστε να δούμε πώς θα προχωρήσουμε. Και μετά να σας αναφέρουμε τα όσα θα γίνουν. Ας δούμε λοιπόν τι μέσα διαθέτουμε και πώς θα τα χρησιμοποιήσουμε με τον καλύτερο τρόπο. Θα συμφωνούσατε με αυτό. Υπέροχα. Έτσι θα πράξουμε λοιπόν αφήνουμε την αναφορά ανοιχτή και συνεχίζουμε. Συμφωνείτε? Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ. Αυτό λοιπόν θα κάνουμε και να είστε έτοιμοι εσείς στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα σας τηλεφωνήσουμε. Σας ευχαριστώ και εσάς για τη συνεισφορά σας. Λοιπόν, αυτό δεν σημαίνει ότι λύνεται το πρόβλημα. Σε καμία περίπτωση τουλάχιστον προσπαθούμε να δούμε ε, πώς θα κάνουμε το επόμενο βήμα αφού κάναμε αυτό το βήμα τώρα. Σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε και νομίζω ότι έχουμε καθυστερήσει πάρα πολύ και θα πρέπει να περάσουμε αμέσως στην επόμενη αναφορά που είναι από τη Γαλλία εξ ονόματος της Ένωσης Διαμάν σχετικά με τα δικαιώματα των ατόμων που πάσχουν από αυτισμό στη Γαλλία. Εδώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρευρίσκεται ο κύριος Λαβρέντζος και του δίνω μέσω στο λόγο. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. La Η αναφέρουσα ισχυρίζεται ε, ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα και το δικαίωμα ε, η μη διάκριση ε, στην εκπαίδευση είναι κάτι το δεδομένο, αλλά στη Γαλλία τα άτομα που πάσχουν από αυτισμό δεν πρέπει τα δικαιώματά τους να γίνονται σεβαστά και ζητά από το Κοινοβούλιο να ε, ληφθούν μέτρα για να μην είναι σε ψυχιατρικά ιδρύματα. Στη Γαλλία όμως θεωρείται ψυχιατρική ασθένεια αυτισμός και όχι νευροβιολογική ασθένεια. Η αναφέρουσα ισχυρίζεται ότι στη Γαλλία τα άτομα που πάσχουν από αυτισμό δεν απολαμβάνουν ίση μεταχείριση, ούτε υφίστανται μεταχείριση με βάση τι ικανότητε και τα δικαιώματά τους. Και ζητάει να βρεθεί ένας τρόπος που να ενθαρρύνει την ανάπτυξή του στο έπακρο. Το 2003 Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κοινωνικών Δικαιωμάτων, ένα σώμα του Συμβουλίου της Ευρώπης, εξέδωσε μία απόφαση επί καταγγελίας της Ένωσης ε, κατά της Γαλλίας. Η απόφαση αναφέρει ότι η κατάσταση των ατόμων που πάσχουν από αυτισμό στη Γαλλία λόγω χάρη εκπαιδευτική τους κατάσταση παραβιάζει τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη. Αυτός ο χάρτης έχει σχέση επίσης με το Συμβούλιο της Ευρώπης. Το 1961 υιοθετήθηκε και αναθεωρήθηκε το 1996. Θα έρθω στη συνέχεια ε, στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, η οποία κυρώθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και προστατεύει τα δικαιώματα των παιδιών με αναπηρία και το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία στην εκπαίδευση, άνευ διακρίσεων και επί τη βάση της ισότητας των ευκαιριών. Είναι τα άθρεπτα και 24 της ελόγου σύμβασης. Η γαλλική νομοθεσία σχετικά με την ισότητα των ευκαιριών για τα άτομα με αναπηρία έχει τεθεί σε ισχύ από το 2005. Είναι ο νόμος 102 κάθετος 2005 της 11 Φεβρουαρίου του 5 και προβλέπει την υποχρέωση ένταξης των παιδιών με αναπηρία στο κανονικό εκπαιδευτικό σύστημα. Επιπλέον η Γαλλία εφήρμοσε το σχέδιο για τον αυτισμό 2008-2010, το οποίο επέβλεπε σε τρεις σκοπούς. Τη βελτίωση της επιστημονικής γνώσης σχετικά με τον αυτισμό, καθώς και της επαγγελματικής κατάρτισης. Την καλύτερη αναγνώριση των ατόμων που πάσχουν από αυτισμό με σκοπό την ενίσχυση της βοήθειας προς τα άτομα αυτά και τις οικογένειές τους και τη διαφοροποίηση των προσεγγίσεων με παράλληλο σεβασμό των ατομικών θεμελιωδών δικαιωμάτων. Περισσότερα από 170 εκατομμύρια ευρώ έχουν διατεθεί για τη σύσταση 4.100 περίπου επιπλέον θέσεων για άτομα που πάσχουν από αυτισμό μέχρι το τέλος του 2012. Αυτά παρατηρεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν για την παρούσα αναφορά. Η Επιτροπή δεσμεύεται πλήρω ω προ την προστασία και την προώθηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων καθώ και τη βελτίωση τη κατάσταση των ατόμων με αναπηρία στην Ευρώπη. Δύο είναι τα άρθρα του Χάρτη Θεμελιδών Δικαιωμάτων που αναφέρονται σχετικά. Το άρθρο 24 που προβλέπει ότι τα παιδιά έχουν δικαίωμα στην προστασία και τη φροντίδα που απαιτούνται για την καλή διαφύωσή τους και το άρθρο 26 επίσης του χάρτη που αναγνωρίζει και σέβεται το δικαίωμα των ατόμων με ειδικέ ανάγκες να υποφελούνται μέτρων που θα τους εξασφαλίζουν την αυτονομία, την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή τους στον κοινωνικό βίο. Ωστόσο, υπάρχει και ένα άρθρο 51.1 του χάρτη που ορίζει ότι οι διατάξεις απευθύνονται στα κράτη-μέλη μόνο όταν εφαρμόζουν το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει και το άρθρο 6 τη Συνθήκη για τη Λειτουργία τη Ευρωπαϊκή Ένωση που λέει ότι οι διατάξει του χάρτη δεν συνεπάγονται καμία επέκταση των αρμοδιοτήτων τη Ένωση όπω αυτέ ορίζονται στι συνθήκε. Και τέλο θέλω να σα αναφέρω και το άρθρο 165 τη Συνθήκη σύμφωνα με το οποίο η οργάνωση του εκπαιδευτικού συστήματος και το περιεχόμενο της εκπαίδευσης είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών και όχι των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Επί τη βάση λοιπόν όλων αυτών η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έρχεται να διαπιστώσει ότι δεν παραβιάζεται το κοινοτικό δίκαιο και δεν μπορεί να επέμβει Βεβαίως ε, ενδιαφέρει τα κράτη-μέλη να σέβονται πλήρως τα δικαιώματα των παιδιών αλλά θεωρεί ότι σε αυτό το κεφάλαιο της εκπαίδευσης και της παιδείας δεν μπορεί να διαπιστώσει ότι έχει παραβιαστεί το κοινοτικό δίκαιο και θεωρεί ότι η αναφορά αυτή πρέπει να κλείσει. Ε, Ευχαριστώ πολύ. Συζήτηση τώρα. Rosa, the Η Ρώσα Sí, muchas gracias. Ε, Ευχαριστώ πολύ. Όπως τα είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι αρμοδιότητε για την ε, παιδεία είναι κάτι το οποίο υπάγεται στην αρχή τη χωρικότητα, άρα είναι θέμα κρατών μελών, αλλά κάποια κρατημέλη έχουν ε, μετακυλήσει αρμοδιότητα στι ε, περιφερειακέ αρχέ. Οπότε η Ένωση προσυπέγραψε τη σύμβαση του ΟΗΕ για του αναπήρου, στην οποία σύμβαση μιλούν και για την παιδεία. Και λέει ότι όλοι θα πρέπει να υπαγόμεθα σε μια τέτοια ρύθμιση για την παιδεία και έχουμε αυτά τα ειδικά σχολεία όταν η αναπηρία είναι πάρα πολύ βαριά και αυτό αποτελεί μια εξαίρεση ούτω ώστε να είναι δυνατόν να πετύχουμε ε, το στόχο αυτό της παιδείας που θα τους αγκαλιάσει όλους, της παιδείας για όλους. Και οι καθηγητές δεν θα είναι ο ένας οποιοδήποτε καθηγητής, θα είναι ένας καθηγητής για όλη την τάξη και θα πρέπει να σεβαστεί την ισότητα των ευκαιριών. Και αυτό είναι μια νομική υποχρέωση. Προσυπογράψαμε τη σύμβαση, αλλά θα πρέπει να δούμε το ότι δεν εφαρμόζεται πουθενά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και η παιδεία για όλους είναι η εξαίρεση και ο κανόνας είναι η ειδική ε, εκπαίδευση. Κάτι το οποίο θα είναι το αντίστροφο το τι έπρεπε να ισχύει. Θα έπρεπε επομένω να αναγνωρίζεται διαφορετικότητα και ένα παιδί μέσα σε άλλα και αν το παιδί αυτό έχει αναπηρία δεν έχει τις με τους άλλους. Άρα είναι αρμοδιότητα κοινοτική να εποπτεύει για την εφαρμογή της ε, διεθνούς αυτής συμβάσεως του ΟΗΕ για την αναπηρία. Για, την, ε, για τον αυτισμό, ένα αυτοκίνητο κατέφυγε στη Γαλλία, τότε τα πράγματα πάνε στραβά κάπου, γιατί ε, αυτή η περίπτωση δεν καλύπτεται από αυτή την ρύθμιση, αυτή τη σύμβαση, σύμβαση ε, ακριβώς όπως υπάρχει η ρύθμιση για την συμπεριληψή στην αγορά εργασία. Έχουμε επομένω τώρα μια τέτοια αναφορά από μια χώρα σαν τη Γαλλία και ο αυτισμό φύσταται αυτού του είδου την, ε, την αντιμετώπιση. Έχουμε εδώ ένα σωρό διαφορετικές περιπτώσεις σε σχέση με τα άτομα ειδικών αναγκών. Θα πρέπει όμως να λάβουμε υπόψη ότι έχουμε εδώ και τα ανθρώπινα δικαιώματα τα θεμελιώδη, αλλά και έχουμε και αυτή τη σύμβαση του ΟΗΕ. Η πολιτική απασχόληση, η πολιτική πολιτικών ελευθεριών και η δική μας εδώ επιτροπή θα πρέπει να εξετάσουμε το πώς έχει υλοποιηθεί, πώς εφαρμόστηκε αυτή η σύμβαση για τους ε, αναπήρους. Και θα πρέπει τώρα να κάτσουμε και να δούμε ότι στα πρώτα σχέδια κειμένου, όπως προέκυψαν και από το φόρουμ για τους αναπήρους, ε, είχαν αυτά τα κείμενα λέγω πάρα πολλές ελλείψεις. Άρα, η μεγάλη επιτυχία που προήλθε από αυτή τη Διεθνή Σύμβαση, ε, όπως κάθε περίπτωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ε, έχουμε εδώ το θέμα του να είναι όλα καλά και στρογγυλά στο γράμμα, αλλά να μην έχει εφαρμοστεί το γράμμα του νόμου. Άρα θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουμε το Ευρωπαϊκό Σχολείο εδώ των Βρυξελών. Δεν είναι ένα σχολείο που τους καλύπτει όλους. Υπάρχουν πάρα πολλά παράπονα που έχουν έτσι στην ε, Επιτροπή των Αναφορών. Όμως θα πρέπει να απασχίσουμε να πετύχουμε τον επιθυμητό μας στόχο. Ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ. Άρα, δεν θα συνεχίσουμε τη συζήτηση. Και διαπιστώνουμε ότι δεν έχουμε τώρα παραβίαση διάταξης ε, του κοινωτικού δικαίου. Αυτό που θα πρέπει να κάνουμε είναι να κάνουμε κάτι. Προτείνω να διαβάσουμε μια επιστολή σε αυτό το φόρουμ για την αναπηρία εδώ στις ε, Βρυξέλλες και στην, στον φορέα Save Our Children και να τους επισημάνουμε το πρόβλημα. Έχετε να προτείνετε κάτι άλλο. Ε, εντάξει, ξέρω, είμαστε λίγο πεσμένοι τέτοια ώρα, αλλά τέλος πάντων ε, είμαστε αναγκασμένοι κάτι να σκαρφιστούμε εδώ επί τόπου. Επομένως, περιμένω τη γνώμη σας. Ναι, είναι καλή ιδέα, ωραία. Θα κάνουμε αυτό επομένως. Καλώς. Οπότε τώρα προχωρούμε. είδαμε το θέμα το προσωπικό γίνεται τόσο δύσκολο και τώρα πάμε στον ανταγωνισμό και πάμε ε, όσον αφορά αυτού του είδους την εξαίρεση αυτών των παραχωρήσεων από το τελικό κράτο και έχουμε εδώ πέρα του αναφέροντε τον Λορέντζο και τον ε, Σεβανο Τζοβάνι και έχουμε επίση ο κύριο Λαβάτζη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οπότε πρώτα πρώτα δώσουμε το λόγο στους ε, αναφέροντες. Παρακαλώ. Δεν έχουμε χρόνο. Προσέξτε, προσπαθήστε να είστε συγκεκριμένοι. Bene, grazie Σας ευχαριστούμε τόσο πολύ για το ότι εδώ μας ε, ακούτε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για την μα Ονομάζομαι Παπάνη και είμαι πρόεδρος ε, αυτής της Ομοσπονδίας ΦΕΔΕ. Φέντερ Μπάιν, δηλαδή που εκπροσωπούμε πάρα πολλέ επιχειρήσει που ενδιαφέρονται για την εκμετάλλευση ε, παρακτήων ζωνών και ε, είναι κάτι που αφορά τι μικρομεσαίε επιχειρήσει και οπότε θεωρούμε ότι φροντίζουν αυτό το τόσο πολύτιμο ιταλικό προϊόν ε, το οποίο αφορά τα, τα, την, το τουρισμό στην Ιταλία, Ιταλία είναι ιταλικό προϊόν Τώρα, γιατί κάνουμε αυτήν την ε, αναφορά. Πάνω από 10 χρόνια οι Ιταλικές αρχές δεν μπόρεσαν να μας καλύψουν όσον αφορά το Ιταλικό δίκαιο το οποίο ρυθμίζει ε, το πώς, το ε, οι παραχωρήσεις των παρτίων ζωνών και από το 2006 δεν έγινε τίποτα μετά το νόμο αυτό το 296. και οπότε με αυτή μας την αναφορά θέλουμε να καταφέρουμε το να προκύψει μια μέθοδος, ένα κριτήριο, μια διάταξη που να εφαρμόζει τον σχετικό νόμο. Πάρα πολύ ικανοποιητική ήταν η υποδοχή της αναφοράς μας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σήμερα πρέπει να σας πούμε ότι ε, συνεννοούμαστε με τις Ιταλικές Αρχές για να κλείσει το θέμα μέσα στην φετινή χρονιά. Και πρέπει να σας πούμε ότι μιλούμε για κτές 8.000 χιλιόμετρων. 4.000 είναι πλάζ που μπορούν να διατεθούν. Και το περίφημο κριτήριο της ελευθερίας εγκατάστασης που προβλέπεται στην οδηγία Βόλκεστάιν θεωρούμε ότι δεν συντρέχει στη δική μας περίπτωση. Οπότε το θέμα είναι κατά πόσον διατίθενται αυτές οι πράκτικες ζώνες από το κράτος. Εμείς θέλουμε να υπάρχει μια ε, προστασία στις 30.000 οικογενικές ε, επιχειρήσεις που είναι μικρές επιχειρήσεις. Και οπότε εδώ ε, από το 2016 θα αρχίσουν να τρέχουν καινούργιες παραχωρήσεις και θα υπάρχει ένα κριτήριο για τις ε, επενδύσεις αλλά επίσης αυτό θα αφορά και την ε, απασχόληση ε, το οποίο θα προέρχεται από αυτές τις αρχές που παραχωρούν οπότε θα έχουμε κάποιο είδους εκμισθώσεις 5 έως 30 ετών ανάλογα βέβαια με τις επενδύσεις που τελικά θα υλοποιηθούν τώρα να δώσω το λόγο στον Τανίλο Λορέντζο Είναι νομικός, ο οποίος θα σας πει συγκεκριμένα ε, τι γίνεται με τον νομικό που ισχύει. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Όπως είπε ο κύριος ε, Παπάνη, να σας πω από πλευράς τεχνικής το τι ισχύει. Μια από αυτήν η δουλειά μου. Όσον αφορά την αναφορά μας, καταγγέλνουμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό το ότι ήδη υπάρχει μια νομοθεσία ο, ο νόμος του 93 του 44, που δεν ε, ε, επιτρέπει παραχώρηση να ισχύσει μέχρι 20 χρόνια όσον αφορά συγκεκριμένες επενδύσεις που οι επιχειρήσεις θέλουν να ανακάνουν όσον αφορά αυτού του είδους ε, την γη του δημοσίου και να την βελτιώσουν αυτή την επένδυση. Οπότε είπαμε η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει ε, αυτόν τον νόμο επί τη βάση της ε, οδηγίας Πόλκισταν, κατά τη γνώμη μας. Δεν συγκρούεται η Ιταλική νομοθεσία με την οδηγία Μπόλτεστάιν. Τον Αύγουστο του 2014 η Επιτροπή ε, γνωμοδότησε και διαπιστώθηκε επίσης ότι η διάρκεια αυτής της παραχώρησης είναι μια δραστηριότητα που είναι αρμοδιότητα του κράτους μέλους. Και ε, αφορά τους διάφορους τρόπους αξιοποίησης ή παραχώρησης περιουσίας του δημοσίου. Θέμα τώρα αν υπάγεται στην οδηγία Μπόλκεσταν αυτή η δραστηριότητα. Υπάρχει τώρα κάτι πάρα πολύ σημαντικό το οποίο διαπιστώθηκε, ότι δηλαδή αυτού του παραχωρήσει δημοσίου χώρου ήδη υπάγονται σε κάποια οδηγία που συνάδει προς την οδηγία Μπόλκεστάιν. Αλλά δεν υπάρχει κάποιος Ιταλικός νόμος. Έχουμε όμως το άρθρο 18 του κώδικα που ρυθμίζει αυτές τις παραχωρήσεις και λέει ότι θα πρέπει αυτές οι παραχωρήσεις να γίνονται ε, και να γίνεται και δημοσίευση της παραχώρησης. Οπότε, μπορεί κάποιος να υποβάλει ένσταση όσον αφορά την παραχώρηση αυτού του δημοσίου αγαθού. Και στην περίπτωση κατά την οποία έχουμε πιο πολλές τέτοιου είδους ε, ε, αιτήσει τότε παραχωρείται το δημόσιο αγαθό σε αυτόν παρέχει περισσότερε εγγύσει για την αξιοποίησή του. Οπότε αυτέ οι παραχωρήσει του δημοσίου αγαθού τώρα έχουν υπαχθεί σε αυτή τη διαδικασία. Κατά τη γνώμη μα, πρόκειται για μια διαδικασία η οποία είναι σύντομη με την οδηγία για τι ε, υπηρεσίε. Υπάρχει διαφάνεια, όλοι μπορούν να συμμετάσχουν και υπάρχει αυτή η δημοσίευση τη οδηγία. Ε, και έτσι υπάρχει εγγύηση για όλους ότι έχουν το δικαίωμα να ασκήσουν ε, αυτού του είδους ε, την, την επένδυση, να κάνουν αυτή την επένδυση για το δημόσιο αγαθό. Και αυτή η διαδικασία επομένω δεν έρχεται σε αντίθεση με τον οδηγία για τις υπηρεσίες. Οπότε η Φέντερ Μπαλνεάρη θέλει αυτές οι παραγωγές που ήδη έχουν γίνει να θεωρηθούν ότι δεν αντιβαίνουν στο κοινοτικό δίκαιο το οποίο ρυθμίζει ε, την χρήση, την απόλαυση το, του δημοσίου αγαθού. Η Πρόεδρος, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν τόσο ε, σύντομος για να μας περιγράψετε το πρόβλημα. Και τώρα, όποιος θέλει μπορεί κάτι να ρωτήσει, να παρατηρήσει. Συνάδελφε, κόμι. Ναι. ένα πρόβλημα που σχετίζεται με την οδηγία Μπόλκεστάιν ε, είναι πρόβλημα ευρωπαϊκών διαστάσεων και το εντοπίσαμε και κατά την προηγουμένη κοινοβουλευτική θητεία. Αυτό το οποίο τώρα είπαμε ακολουθεί την ανάλυση αυτή που έχει γίνει από πλευρά τη Ιταλίας και υπάρχει ένα πρόβλημα. Έχουμε 30.000 οικογένειες που πλήσονται από την ανεργία. Και πρόκειται επομένω εδώ για ε, τι επιχειρήσει του, οι οποίε είναι οικογενειακέ επιχειρήσει. Έχουμε και το Small Business Act και τις οδηγίες της αγοράς, ούτως ώστε να υποστηριχθούν αυτές οι οικογενειακές μικροεπιχειρήσεις. Θεωρούμε ότι η Ευρώπη μπορεί να βοηθήσει, να κρατηθεί ανοιχτή αυτή η αναφορά. Γιατί η Ιταλική κυβέρνηση ακριβώ όπω ελέγχθη δεν μπόρεσε να προχωρήσει προ κάποια επίλυση του προβλήματο. Είπαμε ότι δεν υπάρχει αυτόματη ρύθμιση και για τις νέες παρακτίες περιοχές, νέε πλάζ, δεν θα πρέπει να ισχύσει η αρχή της ελευθερία αγοράς και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεώρησε ότι ήταν θέμα διαπραγμάτευσης της κυβέρνησης με τους παγιωμίδες του κλάδου. Αυτοί που έχουν επενδύσει και έχουν επενδύσει σημαντικά χρήματα για αυτές τις δραστηριότητες οι οποίοι θα μπορούν να ασκούν αυτή τη δραστηριότητα για τον χρόνο στον οποίο θα καταλήξουν σε συμφωνία με την κυβέρνηση. Και είχαμε ε, ε, από πλευρά Φόρτσα Ιτάλια ή όπως είπε και ο Αλμπέρτο, προσπαθήκαμε, φτάσαμε να ε, προωθήσουμε το θέμα στα πλαίσια της εθνικής αρμοδιότητας, γιατί εδώ πέρα πρόκειται για παραχώρηση δημοσίας περιουσίας. Μπορεί να αποφασίσει η κυβέρνηση, αλλά σε σχέση με όλα όσα ήδη τώρα ισχύουν θα πρέπει να δοθεί μια συνέχεια, αν όχι παρά, παράταση αυτής της δραστηριότητας. Γιατί τώρα υπάρχει μια βεβαιότητα για το τι θα ισχύσει τον Ιούνιο, τι θα ισχύσει τον Ιούλιο, οπότε κανένας δεν μπαίνει στην αγορά. Και άρα εδώ υπάρχει πρόβλημα, επαγγελματικό πρόβλημα απασχόλησης. Άρα και αυτό λέμε θα πρέπει να βοηθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση αν θέλουμε μια ένωση ευρωπαϊκή που να είναι πολιτική, να, τι μπορεί να κάνει. Πάντως η Ιταλική κυβέρνηση ακόμα δεν έκανε τίποτα. Και τελευταία φορά μιλήσαμε το Δεκέμβριο. Ε, κατόπιν είχαμε την καινούργια θητεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και γι' αυτό και εκπροσωπώντα τους πολίτες προσπαθούμε να βρούμε κάποια βοήθεια, κάποια υποστήριξη και θέλουμε να μην ανοιχτεί η αναφορά και να συνεχίσουμε για την προσπάθεια εξέβρεση λύση. Η πρόεδρος, σας ευχαριστώ, αλλά έκαναν λάθο. Ε, ξέχασα ότι εδώ πέρα ε, έχουμε και τον αναφέρον της αναφοράς 15-17, τον τρίτο. Για να δούμε. Προσπαθούμε τώρα να δούμε τι θα γίνει. Πώ μπορούμε να, να κατά πόσο αυτή η Επιτροπή τη Οδική Αγορά έκανε κάποιο λάθο. Και με λίγα λόγια θεώρησε ότι αυτή η εκχώρηση είναι μια απλή αδειοδότηση για υπηρεσίε, αλλά τελικά δεν έγινε καμία τέτοια δραστηριότητα. Απλώ ε, έτσι δίνει την δυνατότητα στον, ε, ε, στον ανάδοχο να μπορεί να ασκήσει μια τέτοια δραστηριότητα σε, δημόσιο, σε δημόσιο χώρο. Και πρόκειται για κάτι που είναι δημοδιωτική υπόθεση, γίνεται, δίνεται μια, ένα ετήσιο μίσθωμα, άρα είναι σαν κάτι, ε, ε, κάτι σαν εκμίσθωση. Πρόκειται μέσα εδώ πέρα για κάποιες δραστηριότητες επικερδής, παροχή ε, υπηρεσιών, αλλά αυτό ε, δεν είναι πάντα, πάντα έτσι. Διότι υπάρχουν και ε, κάποιο είδου έτσι εκχωρήσει απλώ για να χρησιμοποιηθεί, για να μείνει κάποιο. Και έχουμε επομένω το άρθρο 12 που λέει ότι όταν υπάρχουν αυτέ όλε οι, οι αδειοδοτήσει για συγκεκριμένη δραστηριότητα, τότε μπορούμε ε, να ρυθμίσουμε να έχει αυτόματη ανανέωση και άρα θα πρέπει να υπάρχει κάποια λύση της σύμβασης μέσω μιας επιλογής των υποψηφίων. Όμως εδώ πέρα όσον αφορά αυτή την ε, δραστηριότητα έχουμε διάφορες δραστηριότητες και αυτή η δραστηριότητα αφορά πολλαπλής χρήσης και δεν εξαρτάται από την άδεια που θα δοθεί. Αλλά όσον αφορά και τη χωροταξία και τις τοπικές αρχές, ε, έχουμε πολλές φορές παροχή υπηρεσιών όπως εστιατόρια, ε, κέντρα διασκέδασης, δισκοτέκ κλπ. Ne Επομένως θα πρέπει να υπάρχει κάποιο είδους ρύθμιση για την λήξη αυτών των ε, παραχωρήσεων. Κάτι το οποίο οδηγεί στη λύση της αυτόματης ανανέωσης. Και έτσι να σε κάποια δραστηριότητα, οποιαδήποτε είναι αυτή, που δεν έρχεται σε σύγκρουση με την οδηγία στο άρθρο 12. Εκεί που αναφέρονται οι φυσικοί πόροι που αφορούν όχι ε, την ιδιωτική χρήση, αλλά την ε, κρατική περιουσία. Στην περίπτωση αυτών των χώρων που έχουν παραχωρηθεί, ε, έχουμε τις ρυθμίσεις από πλευράς των τοπικών αρχών και έχουμε κάποιο είδους ε, προγράμματα χωροταξικά, εθνείς χωροταξικές, για να υπάρχει η εκμετάλλευση των χώρων ε, και πρόκειται για φυσικές πηγές, ε, φυσικού πόρους που καλύπτει το άρθρο 12. Πρόεδρος, νομίζω ότι επαναλαμβάνεται όλα όσα έχει διλεχθεί. Παρακαλούμε, μπορείτε να είστε συντομότερος γιατί πιέζει ο χρόνος. Μάλιστα, λέω να θέλω. Εν κατακλείδη, θα μπορούσαμε να δούμε κατά άλλο τρόπο. Έχουμε την οδηγία του 2014, του 23, που αφορά ε, κάποιες συμβάσεις εκχώρησης που αφορούν ε, υπηρεσίες και παροχή ε, άλλων ε, εργασιών οπότε αφορά αυτούς τους πόρους, τους φυσικούς πόρους και δεν θα πρέπει να θεωρηθούν εκχωρήσεις εν τη ενία της παρούσης οδηγίας. Οπότε φαίνεται ότι είναι παράλογο το ότι αυτού του είδους οι παραχωρήσεις δεν θεωρούνται ότι είναι παραχωρήσεις για παροχή υπηρεσιών. Οπότε θα ήθελα να σας τονίσω τις συνέπειες από αυτή, από αυτή τη λαθασμένη ερμηνεία. Και δεν είναι αδύνατο να μεταφραστεί ο μιλητή γιατί διαβάζει πάρα πολύ γρήγορα. Il domicilio e la sede l'impresa sono le stesse, quindi spesso nella concessione anche l'abitazione. Οπότε, πάρα πολλέ οικογένειε διακινδυνεύουν όλε του τι επενδύσει. Και η ζημία είναι τεράστια. Και θα ήθελα να ζητήσω εν τέλει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει υπόψη το εφαρμόσιμο αυτής της οδηγίας για αυτού του είδους της παραχωρήσεις και ότι ε, θα πρέπει να υπάρχει μια συγκεκριμένη οδηγία για τέτοιου είδους παραχωρήσεις που να εφαρμόζεται σε όλες τις χώρες και να μην υπάρχουν δυσμενείς διακρίσεις και έτσι να παραβλάπτεται ο ανταγωνισμός ιδίω όσον αφορά τον τουρισμό. Θα πρέπει να θεωρηθεί σωστή η εφαρμογή της οδηγίας και ζητώ να υπάρχει μια παράταση, να υπάρχει μια μεταβατική περίοδος, όπως γίνεται στην Ισπανία. Και αυτό να είναι το ελάχιστο όριο, η παράταση 30 ετών έως 75. The Commission... Ευχαριστώ πολύ. Τώρα θα δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον κύριο Τιέντιε. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομο διότι οι αναφορέ αυτέ έχουν ήδη συζητηθεί εκτενώ. Θα σα ενημερώσω για τι νεότερες εξελίξεις. Καταρχάς, αυτή τη στιγμή συζητούμε πώς να εφαρμόσουμε την εφιστάμενη νομοθεσία στις συγκεκριμένες περιπτώσεις. Ε, έχει διατυπωθεί το επιχείρημα του αν μπορούμε να εφαρμόσουμε την οδηγία για τις υπηρεσίες ή όχι. Και καταλήξαμε πώς μπορούμε. Βέβαια, οι, συνθήκη, οι συνθήκες εγγυώνται διάφορα δικαιώματα, όπως το δικαίωμα εγκατάσταση, για παράδειγμα, και φυσικά το δικαίωμα της ε, διαφάνειας όσον αφορά την πρόσβαση σε μια συγκεκριμένη αγορά. Όταν λοιπόν κάποιος θέλει μια έγκριση για μια παραχώρηση, πρέπει κατά καιρού να γίνεται προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού. Και αυτό με φέρνει στο επόμενο που θα ήθελα να πω. Πολύ συχνά Πρόκειται για οικογενειακές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις περιοχές αυτές. Λοιπόν, παίζονται πάρα πολλά για εκείνους. Επίσης, νομίζω πως δεν μπορούμε να λάβουμε μια απόφαση σήμερα, διότι εκκρεμεί μια απόφαση ενώπιον του δικαστηρίου στο Λουξεμβούργο από τον Οκτώβριο του 2014. Είναι η 158 κάθετος 14, 458 κάθετος 14, για την διοικητική κατάσταση στη Λομβαρδία και το περιεχόμενό της είναι αντίστοιχο. Η υπόθεση λοιπόν αναφέρεται, που αναφέρεται στη Λίμνη Γκάρτα ασχολείται με το ίδιο θέμα. Έχει λοιπόν γίνει αυτή η προσφυγή στο δικαστήριο του Λουξεμβούργου και επομένως υπάρχει νομοθεσία γι' αυτό. Γι' αυτό πιστεύω πως δεν είναι θέση της Επιτροπής Αναφορών να αποφανθεί αυτή τη στιγμή, αλλά του δικαστηρίου στο Λουξεμβούργο. Γι' αυτό πρέπει να περιμένουμε και να δούμε τι θα γίνει εκεί. Κατά τα άλλα, συνεχίζουμε τις ε, συζητήσεις για τεχνικά ζητήματα με τις Ιταλικές αρχές και φυσικά πρέπει να βρούμε μια ισορροπία, να υπάρχουν μεν οικονομικές ελευθερίες, να υπάρχει κάποιος ανταγωνισμός, από την άλλη όμως να προσπαθήσουμε να ισορροπήσουμε αυτόν τον ανταγωνισμό με τις οικογενειακές αυτές υπηρεσίες και την προστασία τους. Σας ευχαριστώ πολύ. Ήσασταν σύντομος και περιεκτικότατος και έτσι θα έπρεπε να είναι όλοι. Και πραγματικά σας άκουσα με μεγάλη χαρά. Τώρα, κανονικά, πρέπει να δώσω το λόγο σε εσάς, όμως, όχι ακόμα στους αναφέροντες, διότι μιλήσατε πάρα πολύ ώρα πιο πριν. Θα ήθελα να ακούσω τώρα τα μέλη της Επιτροπής. Σύντομα παρακαλώ. Κύριε Ακόμη. Όχι, μια διευκρίνηση κύριε Πρόεδρε. Το λόγο λόγω άρθρο αποκλειστικά αφορά τις ε, παραχωρήσεις σε σχέση με, τις, με τους θαλάσσιους χώρους. Γι' αυτό η αναφορά αφορά αυτού του είδους τις ε, παράκτιες περιοχές. Πάρα πολύ ωραία η λίμνη, αλλά είναι άλλη υπόθεση. η λίμνη της Γκάρντα, απλώς διευκρινιστικά. Κύριε Τσίριο, πολύ σύντομα, απλώς γιατί νομίζω ότι κατόπιν των όσων είπαν και ό,τι είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, μας οδηγεί στο ότι θα πρέπει να μείνει ανοιχτή η αναφορά εν ώψη της γνωμοδότησης ε, των ενεργειών των της Ιταλικής κυβέρνησης οπότε να συνεχιστεί αυτή η διαδικασία ούτω ώστε να μπορέσουμε να παρακολουθήσουμε τι γίνεται, τι θα κάνει η κυβέρνηση και να μην ε, ξεχνούμε ότι αυτό το οποίο διακυβεύεται δεν είναι ναι, μόνο όλες αυτές οι θέσει εργασίας σε επιχειρήσεις, αλλά και όλος ο, όλη η υποδομή τουριστική, γιατί πρόκειται για αυτές όλες τις, ε, τις ακτές, παρακτίες ζώνες, που, όπου γίνεται η μετάλλευση τουριστική και είναι πάρα πολύ σημαντικό για τη χώρα. Πρόεδρος. Ευχαριστώ. Άλλος θέλει το λόγο. Αν τώρα σας ξαναδώσω σε εσά τους αναφέροντες ε, το λόγο, νομίζω θα κάτσουμε εδώ κοβιδιάζουμε μέχρι αύριο. Μήπω ένας, ένας από όλου θα μπορούσε να μα τα πει. Τι θα το ότι πριν, πριν ήμασταν τόσο, τόσο σύντομοι. Θέλω να σας διευνήσω ότι αυτές οι αναφορές ε, δεν είναι η ίδια περίπτωση. Γιατί αν δεν ζητούμε να, να εφαρμοστεί αυτός ο νόμος. Πρόκειται για την ελευθερία της εγκατάστασης. Όμως, στην άλλη αναφορά, αυτό το οποίο θέλουμε και προβάλλουμε τα επιχειρήματα είναι όλος ε, διαφορετικά. Δεν το έχω καταλάβει πάρα πολύ καλά, αλλά νομίζω ότι η δική μας ε, αναφορά έχει μία διαδρομή, μία κατεύθυνση, ένα στόχο. Δεν ξέρουμε και δεν ξέρουμε τι γίνεται με την άλλη αναφορά. Ωραία. Ακούστε. Τι θα μπορούσαμε να κάνουμε από αυτού τώρα όπως λέει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πρώτη αναφορά. Να ενθαρρύνουμε τους αναφέροντες που βεβαίως έχει το δικαίωμα να προσφύγει, να προσπαθήσει να βρει το δίκαιο του σε εθνικό επίπεδο για να αποζημιωθεί. Δεν έχει εξαντληθεί η δικαστική οδό σε εθνικό επίπεδο. Στο μεταξύ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύτηκε να ε, αρχίσει ένα διάλογο με τις αρμόδιες Ιταλικές αρχές έτσι ώστε η οδηγία για τις υπηρεσίες να εφαρμόζεται πλήρως. Να το διασταυρώσουμε αυτό δηλαδή και σύμφωνα με το υλικό που μας έχει δοθεί, διαβάζω, έχετε δεσμευτεί να το κάνετε. Να φροντίσετε να εφαρμόζεται και για τις εγχωρήσεις για παραλίες ε, αυτή η οδηγία. Το ξέρω ότι είναι πάρα πολύ ε, περίπλοκο αυτό το θέμα, εκρεμεί και στο δικαστήριο στο Λουξεμβούργο. Θα μπορούσαμε ακόμα και να κλείσουμε αυτές τις αναφορές και να περιμένουμε την απόφαση του δικαστηρίου. Στο Λουξεμβούργο ή μπορούμε και ανοιχτή να την αφήσουμε και τη μία και την άλλη. Σε εμάς είναι απόκειτο αυτό. Open, ανοιχτή. Συμφωνείτε οι άλλοι συνάδελφοι. Ωραία. Δεν κλείνουμε λοιπόν τις αναφορέ αυτές. Ευχαριστώ πολύ. Προχωρούμε και ελπίζω να είναι ικανοποιημένοι και οι αναφέροντες. Αλλά σας εθαρρύνω να ε, κρατήσετε ανοιχτό το διάλογο με τις αρμόδιες ιταλικές αρχές, όχι μόνο με εμά, για να βεβαιωθείτε ότι η οδηγία θα εφαρμόζεται σωστά και απολύτως. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι δεν εφαρμόζεται απολύτως. Εν Πάμε στι μεταφορέ τώρα. Έχουμε μια αναφορά από την Πολωνία. Στην πόλη Πλοκ που είναι στην κεντρική Πολωνία σχετικά με προβλήματα μεταφορικών υποδομών. Παραμελημένοι δρόμοι, και υποδομές μεταφορών. Θα δώσω αμέσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αφού δεν παρευρίσκονται οι αναφέροντες. Η κυρία Καρολίνα Ντιμπόφσκα έχει το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η αναφορά αφορά μια πολωνική πόλη και δράτω με τις ευκαιρίες για να μιλήσω τη μητρική μου γλώσσα που είναι τα πολωνικά. Λοιπόν, η αναφορά αυτή αφορά μια κοινωνική εκστρατεία που γίνεται για να διορθωθεί η υποδομή μεταφορών στην πόλη Πλοκ που είναι και μια ε, πόλη, ένα εξαιρετικά σημαντικό κέντρο παραγωγής καυσίμων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τα όσα προτείνει ε, ο αναφέρον να σας πω τι άποψη έχει. Ε, θέλω να αναφέρω δύο ζητήματα. Το ένα έχει να κάνει με την πολιτική συνοχή και τη ε, συνδιαχείριση, τη συνυπευθυνότητα, που ε, είναι μια εταιρική σχέση και διαχείριση κοινή μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των κρατών μελών. Είναι στη συνυπευθυνότητα δηλαδή. Έχω την έννοια αυτή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκεί δεν αναμειγνύεται στην επιλογή του έργου, εκτός από τα βασικά μεγάλα έργα υποδομών που γίνονται. Δηλαδή για πολύ μεγάλα έργα από ένα επίπεδο και πάνω. Το, το 2007-2013 ήταν 50 εκατομμύρια, μέχρι το 2012 ήταν 75 εκατομμύρια. Πάντα για τις μεταφορές μιλούμε και τις αντίστοιχες υποδομές το νέο πλαίσιο και τη νέα προγραμματική περίοδο ε, είναι πλέον πιο ανεπτυγμένη η περιφέρεια, το πλοκ, και είναι περιορισμένη η δυνατότητα χρηματοδότησης από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες. Είναι τέσσερις οι θεματικές ενότητες. Τώρα, τι σημαίνει αυτό για τη συγκεκριμένη αναφορά. Στην τρίτη αναφορά, όπως αναφέρεται εδώ, γίνεται μία πρόταση για νέα νομοθεσία η οποία θα αναγκάζει τα κράτη-μέλη να προβαίνουν σε κάποιες ενέργειες έτσι ώστε να εξασφαλίζουν πάντα τη σωστή λειτουργία ε, σε κρίσιμες περιφέρειες για την οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Γενική Διεύθυνση Ρίτζιο για τα περιφερειακά ζητήματα δεν έχει γνώμη για το νομοθέτημα, αλλά έχει γνώμη για τη βελτίωση του δικτύου υποδομών και του δικτύου μεταφορών στην περιφέρεια. Παρά το γεγονός ότι η ε, συγκεκριμένη περιφέρεια δεν είναι από τις πιο μειονεκτούσες, ε, γίνονται διαπραγματεύσεις και για το στρατηγικό αναπτυξιακό πρόγραμμα, το πολωνικό ΕΣΠΑ δηλαδή, για την περίοδο 2014-2020, η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα ληφθεί τέλη του μηνός. Έχουν δρομολογηθεί αυτές οι εξελίξεις. Και σε ένα ε, προσωρινό κατάλογο προβλέπεται αυτό το έργο, προβλέπεται αναζωγόνηση του σιδηροδρόμου στην περιφέρεια εκεί και άλλα έργα υποδομής που θα λάβουν συγχρηματοδότηση και από εθνικούς πόρους. Υπάρχει και ένα έργο που αφορά μια νέα σύνδεση Πλότσκ ε, και MODELING που θα συνδέσει το δηληστήριο ε, του Πλότσκ με τους ευρωπαϊκούς διαδρόμους ε, για την κυκλοφορία της ενέργειας. Θέλω να πω ότι για να κατασκευαστούν νέοι αυτοκινητόδρομοι, αυτό χρειάζεται και κρατική συγχρηματοδότηση. Χρειάζονται εθνικοί πόροι. Αλλά η διαχειριστική αρχή δεν έχει προβλέψει νέα έργα αυτοκινητοδρόμους κλειστούς ας πούμε, πολύ ψηλής ταχύτητας ή όχι. Υπάρχει δυνατότητα όμως επισκευής μικρότερων εθνικών οδών ας πούμε και μικρότερου δικτύου. Τέτοιοι δρόμοι μπορούν να κατασκευάζονται ε, εντός των εθνικών προτεραιοτήτων και εφόσον πρόκειται για χαμηλής εμβέλειας και ε, χαμηλών εκπομπών. Ε, προγράμματα. Αυτά τα έργα δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα ούτε καν ως πρόταση γιατί έχουν να κάνουν με την ολοκληρωμένη περιφερειακή στρατηγική και την ολοκληρωμένη χρηματοδότηση στην Πολωνία. Ε, όλα θα εξαρτηθούν λοιπόν από τα περιφερειακά προγράμματα για τη μαζωρία. Ευχαριστώ πολύ. Ερωτήσεις έχετε? Πιτέρα. Κυρία Πιτέρα. Είναι δύσκολο θέμα αυτό και αφορά την εκλογική μου περιφέρεια και εδώ και παλαιότερα στις εθνικές εκλογές. Είναι κάποιες μικρές, είναι μια μικρή πόλη 130.000 κατοίκων, είναι κοντά στη Βαρσοβία, έχει ένα μεγάλο δηληστήριο είναι πάνω από 100 χρόνια εκεί. Υπάρχουν διάφορα προβλήματα λοιπόν με την εταιρεία και με τις μεταφορές, διότι το πετρέλαιο φεύγει από το πλός προς όλες τις δυνατές κατευθύνσεις στην Πολωνία και υπάρχει λοιπόν θέμα. Δεν νομίζω πως μπορούμε να ισχυριστούμε ότι δεν κάνει επενδύσεις το πολωνικό κράτος. Αυτό δεν ισχύει. Έχουν υπάρξει διάφορες πρωτοβουλίες. Για παράδειγμα, έχουν γίνει ανακαινήσεις στο σιδηροδρομικό δίκτυο, στις γέφυρες. Υπάρχουν όμως προβλήματα που έχουν να κάνουν με τη διαχείριση του δικού δικτύου. Γι' αυτό η απόφαση έχει να κάνει και με το ποιος ξοδεύει τα χρήματα. Η κοινότητα, η περιφέρεια, η κυβέρνηση, το κράτος. Υπάρχουν λοιπόν αυτές οι διαφορές και δυστυχώς υπάρχουν αυτά τα προβλήματα, όμως να σας πω ότι μέχρι τώρα δεν έχει σημειωθεί κάποιο μεγάλο ατύχημα, όμως η περίπτωση που συνέβαινε φυσικά και θα ήταν καταστροφικές οι συνέπειες. Τώρα, να σας πω επίσης ότι αυτές οι επενδύσεις που έχουν γίνει έχουν κοστίσει πάρα πολύ και φυσικά δεν θα γίνουν όλες αμέσως και όλες μαζί. Οι επενδύσεις αυτές θα εφαρμοστούν σταδιακά, σε βάθος χρόνου και χρειάζονται πολλά. Χρειάζονται δρόμοι, χρειάζονται συνδέσεις μεταξύ του, ε, των ε, δρόμων, χρειάζονται δυνατότητες παράκαμψης και όλα αυτά θα χρειαστούν χρόνο, διότι υπάρχουν οικονομικοί περιορισμοί. Θα ήθελα λοιπόν να προτείνω να αφήσουμε ανοιχτή την αναφορά και να ζητήσουμε από την διοίκηση της περιοχής αυτής στην Πολωνία τι γίνεται με το θέμα της ασφάλειας εκεί. διότι μέχρι το 2020 θα συνεχίσουν να γίνονται επενδύσεις και να υλοποιούνται. Και από όσο ξέρω, υπάρχουν εγγύσεις για την ασφάλεια, υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες που διέπουν όλο αυτό το σύστημα και υπάρχει αυτό το σύστημα εκεί έτοιμο να χρησιμοποιηθεί σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύω πως καταρχάς θα πρέπει να δούμε τι γίνεται εκεί. Καταρχάς να απευθυνθούμε στην Επιτροπή Περιβάλλοντος και να τους ζητήσουμε την άποψή τους και πώς θα προσέγγιζαν εκείνη το ζήτημα. Έτσι ώστε να δούμε πώς μπορεί να βλάψει πιθανά το περιβάλλον αυτή η εγκατάσταση και ταυτόχρονα φυσικά να απευθυνθούμε στις πολωνικές αρχές έτσι ώστε να έχουμε ακριβέστερες πληροφορίες. Όμως, από ό,τι καταλαβαίνω, η κυβέρνηση της Πολωνίας κάνει ό,τι μπορεί για να διασφαλίσει την ασφάλεια στην περιοχή. Σας ευχαριστώ πολύ. Υπάρχει κάποιος άλλος που θα ήθελε να προσθέσει κάτι. Η κυρία Πιτέρα πρότεινε λοιπόν να αφήσουμε την αναφορά ανοιχτή. Εγώ θα πρότεινα να στέλναμε μια επιστολή στην κυβέρνηση της Πολωνίας και να αναφέρουμε όλα αυτά που έχουμε κάνει και τις αναφορές που υπάρχουν και αφόσον μας ενημέρωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι δεν υπάρχει καμία παράβαση να κλείσουμε την αναφορά. Όμως πρέπει να επιστήσουμε την προσοχή στο θέμα αυτό και να τους ενημερώσουμε ότι αυτό το θέμα συζητιέται. Και πραγματικά δεν πιστεύω πως θα έπρεπε να παραμείνουν οι αναφορές αυτές ανοιχτές. Δεν έχουμε κάτι άλλο να προσθέσουμε και είναι από το 2013 αυτές οι αναφορές. Αλλά παρακαλώ, ζητήσατε το λόγο. Κυρία Άουγκεν. Χωρίς μικρόφωνο, δυστυχώς. Ευχαριστώ. Καμιά φορά θα πρέπει να είμαστε αρκετά θαραλέοι ώστε να κλείνουμε και κάποιες αναφορές. Καλή ιδέα θα ήταν, όπως είπατε, να στείλουμε μια επιστολή στους αναφέροντες, αλλά να έχουμε και το θάρρος καμιά φορά να κλείνουμε τις αναφορές όταν δεν χρειάζεται να παραμένουν ανοιχτές. Δεν ξέρω. Δεν θέλω να αναγκάσω κανένα, κάνει τίποτα, αλλά δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο και να παραμείνουν ανοιχτές. Ωραία. Κανονικά, εγώ δεν κάνω προσωπική πρόταση μέχρι να ακούσω όλους τους συναδέλφους, αλλά είδα ότι ήσουν οι μόνοι που ήθελες να ε, ε, μιλήσεις. Βλέπω και η Μάργαρε τώρα θέλει να κλείσει η κάθε αναφορά αυτή. να στείλουμε μια καλή επιστολή στην κυβέρνηση και κάποια στιγμή να κλείσουμε τις αναφορές μετά από αυτό. Αφού γράψουμε και στους αναφέροντες, είπαμε, και στην κυβέρνηση. Πώς θα το έβλεπες. Ευχαριστώ. Ναι, θέλω ακριβώς αυτό να προτείνω και εγώ. Να δούμε ποια θα είναι η αντίδραση της πολωνικής κυβέρνησης, τι στάση θα τηρήσει. Μπορεί να καταθέσει ένα πρόγραμμα, γιατί υπάρχει αυτό το πρόγραμμα και έχουμε μια πολύ καλή βάση για να κλείσουμε τις αναφορές αυτές. Αλλά να, μην το αποφασίσουμε τώρα αυτό. Ναι, έτσι λοιπόν θα κάνουμε. Ωραία. Ας προχωρήσουμε τώρα. Και τώρα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα αναφορά. Ο κύριος Μικρόπουλος, καλώς ορίσατε στα ελληνικά η πρόεδρος, για το ρόλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε σχέση με τη χρηματοδοτική βοήθεια που παρέχεται στην Ελλάδα και την εικαζόμενη παράβαση του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σε σχέση με την Ελλάδα. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει προσκληθεί, πρέπει να σας το πω. Τους καλέσαμε να έρθουν εδώ στην Επιτροπή να συμμετάσχουν, αλλά αρνήθηκαν την πρόσκληση. Οπότε είστε εδώ, αναφέρον, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Πρόεδρε, για τον μου δίνετε το λόγο και τη δυνατότητα να βρίσκομαι σήμερα εδώ μπροστά σας. θα ήθελα να εκφράσω την α, έκπληξή μου, τη λύπη μου και την οργή μου για την απουσία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και τι έχουν προσκληθεί. Πραγματικά α, δεν μπορεί να εξηγηθεί. σε κάθε περίπτωση, η υποσυζήτηση αναφορά συντάχθηκε το Μάρτιο του 2012. Οι διαπιστώσεις της υιοθετήθηκαν στο σύνολό τους δύο χρόνια αργότερα με τη μορφή δύο ψηφισμάτων του προηγούμενου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με την προηγούμενη σύνθεση. Παράλληλα υπήρξαν και άλλες εξελίξεις ως προς το περιεχόμενο της αναφοράς όπως η απόφαση του, του ΔΕΚ για την υπόθεση Τόμας Σπρίγκλ κατά κυβέρνηση της Ιρλανδίας αλλά και πολλές εκθέσεις διεθνών φορέων και ανεξάρτητων οργανισμών σχετικά με την καταπάτηση, παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ελλάδα, που και αυτέ επιβεβαίωσαν και συμπλήρωσαν πολλά από τα περιεχόμενα τη αναφορά. Ενδεικτικά αναφέρω την έκθεση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, συντάκτη ο Σέφα Λουμίνα Μάιο 14, για την καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ελλάδα. Η έκθεση Βουλίου τη Ευρώπη, Safeguarding Human Rights in Times of Economic Crisis, Νοέμβριο 2013. Report on Austerity Measures and Economic and Social Rights, Αύγουστος 2013 από United Nations Human Rights Office of the High Commissioner. Επίσης, η έκθεση της Διεθνούς Ομοσπονδίας για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, Δεκέμβριο του 2014 και περιοδικές εκθέσεις του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας. Α, υπό το φως αυτών των, αναφορών, των διαπιστώσεων και των συμπερασμάτων από τους ανεξάρτητους διεθνούς οργανισμούς και φορείς, οι οποίοι είναι και επίσημοι συνομιλητές Ευρωπαϊκής Ένωσης, και πολλοί καταλήγουν σε κοινέ διαπιστώσει και συμπεράσματα ότι η κατάσταση στην Ελλάδα έχει λάβει χαρακτήρα ανθρωπιστική κρίση και υπάρχουν σωρία παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων τα οποία εγγυάται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Βάζω μια ανωτελεία. Η πρώτη απάντηση που έλαβα από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στις 15 Ιουνίου του 2012 μεταξύ άλλων λέει ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν γνωρίζει κανένα μέτρο που έχει ληφθεί από την ελληνική κυβέρνηση στο πλαίσιο του προγράμματο οικονομική προσαρμογή, το οποίο να προσβάλλει θεμελιώδη δικαιώματα ή τι συνθήκε Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απάντησε μερικέ εβδομάδε αργότερα και μεταξύ άλλων συνοψίζει και επιθυμεί να με διαβεβαιώσει ότι ω θεματοφύλακα των συνθήκων παρακολουθεί κατά πόσο τα μέτρα και οι πολιτικέ του προγράμματο συνάδουν με το κινητικό κεφτημένο και καταλήγει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν παρεκκλίνει από τις συνθήκες, ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κρίνει ότι οι πολιτικές αυτές συνάδουν με το κοινοτικό κεκτημένο. Ε, θεωρώ ότι αυτές οι απαντήσεις δεν είναι απαντήσεις, είναι υπεκφυγή, γιατί οι πραγματικότητες τις οποίες βιώνουμε όλοι στην Ελλάδα και είναι γνωστές σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, και αυτές οι πραγματικότητες διαπιστώνονται από ανεξάρτητους οργανισμούς, λένε αυτό που είπα πριν, ότι υπάρχει σωρία παραβάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ελλάδα. Τώρα καταλαβαίνω ότι αν οι πραγματικότητε δεν συμφωνούν με τι διαπιστώσει τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τόσο το χειρότερο για τι πραγματικότητε. Σε κάθε περίπτωση εκκρεμεί μια απάντηση. Στην απόφαση του ΔΕΚ για την υπόθεση Πρίγκλ, για να επανέλθω, μεταξύ άλλων δέχτηκε ότι δεν αντιβαίνει στι συνθήκε ο Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξη. Και σωστά, είναι ένα διακυβερνητικό οργανισμό γιατί έχει σταθεί εκτό του πλαισίου τη Ένωση. Επομένω, τα κράτη-μέλη έχουν αρμοδιότητα για τη σύναψη μεταξύ του συμφωνία, όπω αυτό προβλέπεται. Εν τούτης, και αυτό είναι σημαντικό, τα κράτη-μέλη δεν μπορούν να απαλλαγούν από την υποχρέωση τήρηση του δικαίου τη Ένωση κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του στον τομέα αυτό και οι δεσμεύσει που αναλαμβάνουν τα κράτη-μέλη στον τομέα αυτό πρέπει να είναι συμβατέ με το δίκαιο τη Ένωση. Γιατί απλά, κύριε Πρόεδρε, το δίκαιο δεν αναστέλλεται σε περίοδους χρηματοπιστική κρίση. Το δίκαιο ή υπάρχει ή δεν υπάρχει. Και θέλω να ρωτήσω επίση και με ποιο τρόπο παρακολουθείτε τη συμμόρφωση των κρατών στο ανωτέρω τη σκεπτικό τη απόφαση του ΔΕΚ μέσω τη συμμετοχή σα στην Τρόικα. Αυτή η ερώτηση είναι προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, Επίση, το 10 αποφάσισε ότι τα κράτη-μέλη μπορούν να αναθέτουν επιπλέον καθήκοντα στα θεσμικά όργανα, εφόσον τα καθήκοντα αυτά δεν αλλοιώνουν τι αρμοδιότητε, τι οποίε συνθήκε αναθέτουν στα ελόγω θεσμικά όργανα. Με τη λογική ότι τα θεσμικά όργανα τη Ένωση δεν πρέπει να επιτρέψουν να γίνουν υποχείρια των εθνικών κυβερνήσεων κατά την χρηματοπιστωτική κρίση. Βάσει των ανωτέρων σκέψεων, η συγκρότηση ενό άτυπου εξωθεσμικού οργάνου με τη μορφή ενό σχήματο συνεργασία Τρόικα ελέγχεται λαμβανωμένο υπόψη του γεγονότο ότι αποτελείται από τρία ανεξάρτητα θεσμικά όργανα, άνεση κατανομή αρμοδιοτήτων σε συνδυασμό με διαφορετική αποστολή, διαφορετικέ δομέ διαπραγμάτευση και λήψη απόφαση, με διαφορετικά επίπεδα λογοδοσία όπου υπάρχουν και γενικά στερούμενη διαφάνεια και δημοκρατική επίβλαψη. Όλα αυτά μπορούν να συνοψιστούν με τον όρο σκόπιμα οργανωμένη ανευθυνότητα. Και θέλω να ρωτήσω έχω κάνει κάποιε ερωτήσει πρωτού έρθω, ότι ποια είναι η διαδικασία σχεδιασμού, λήψη αποφάσεων, όταν κατατίθεται ένα πρόγραμμα, καθώ και η πορεία υλοποίηση μόρφωση. Τι προβλέπετε όταν ένα από τα τρία μέρη έχει αντιρρήσεις. Πού λογοδοτούν οι επικεφαλείς της Τρόικας. Εσωτερικό οργανόγραμμα αντιρρήσει, που λογοδοτουν οι επικεφαλει τη τροϊκα. εσωτερικο οργανογραμμα υπαρχει πώ καταρτιζονται οι αποφάσει που υλοποιουνται γιατι δεν δέχομαι την απάντηση ότι εμεί απλά παρέχουμε τεχνικέ συμβουλέ. Αυτό είναι μια καραμέλα η οποία διατυπώνεται επί σειρά ετών. Αυτό στην πατρίδα μου το λέμε περιπεκτικά, είναι παραμύθι για μικρά παιδιά. Δεν είναι τεχνικέ συμβουλέ. Στην πράξη, αυτοί οι κύριοι, οι οποίοι είναι υπάλληλοι τη Ευρωπαϊκή Ένωση, εκβιάζουν εκλεγμένε κυβερνήσει. Εφόσον οι ευρωπαϊκέ συνθήκε είναι σε ισχύ, ο χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων είναι σε ισχύ, το κράτο δικαίου δεν μπορεί να ανασταλεί από αυτού που λαμβάνουν πολιτικέ και οικονομικέ αποφάσει. Δηλαδή από την τράγκα και όσου κρύβονται από πίσω. Όταν λαμβάνονται αποφάσεις ανεξάρτητα από το δίκαιο, τότε απλά δεν υπάρχει δίκαιο. Επίσης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εσείς, διαπίστωσε στο ψήφισμά του, το θεσμικό όργανα της Ένωσης είναι συνυπεύθυνα για τους όρους που επιβάλλονται στο πλαίσιο των προγραμμάτων δημοσιονομικής προσαρμογής. Ε, όλοι συμφωνούν ότι το δημοσιονομικό πρόβλημα της Ελλάδας ήταν κατά κύριο λόγο πρόβλημα συλλογής φόρων λόγω εκταμένης φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής, καθώς και πρόβλημα βραδίας απονομής δικαιοσύνης. Αντί να επικεντρωθεί ευθύ εξ αρχής σε αυτούς τους τομείς από τα πρώτα μέτρα που έλαβε η Τρόικα και πίεσε την αλάβη την ελληνική κυβέρνηση ήταν η απορρίδηψη των εργασιακών σχέσεων και η κατάργηση στην πράξη της δυνατότητας των συνδικαλιστικών οργανώσεων για τη σύναψη συλλογικών συμβάσεων ποιο ποιοι επέβαλαν την ιεράρχηση αυτών των προτεραιοτήτων αντί τη βελτίωση του μηχανισμού ίσπραξη εσόδων. Ενοχοποιήθηκαν μισθοί, συντάξει, κοινωνικά επιδόματα, δαπάνε υγεία, εκθεμελιώθηκαν κοινωνικά δικαιώματα που κατακτήθηκαν μέσα από δεκαετίε αγώνων. Η πρόταξη αυτών των νεοφιλελεύθερων πολιτικών έχει ταξικό χαρακτήρα. Εξυπηρετεί την πρόθεση νεοφιλελεύθερων μέτρων και μεταρρυθμίσεων στι χώρε που κατέφυγαν σε μνημόνια. Οι επικεφαλεί τη Τρόικα, πρώην και νυν, Σερβά Ντερούζ, Γιούργεν Κρούγκερ, Ματία Μόρ, Ντέγκλαν Κοστέλο, Κλάου Μαζού, καθώ και όσοι υπηρετούν στα τεχνικά κλιμάκια είναι υπάλληλοι τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και υπάλληλοι τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Πρέπει να τηρούν το κοινωνικό κεκτημένο. Και η ερώτηση είναι σαφέστατη. Πόσε μέρε το χρόνο ενεργούν με βάση το δίκαιο τη Ένωση, είναι θεματοφύλακε των συνθήκων και όταν παίρνουν το αεροπλάνο για να πάνε στην πατρίδα μου ή σε άλλε χώρε, δεν το τηρούν και το πίσω του. Εδώ υπάρχει διχασμό προσωπικότητα. Στην, ε, υπάρχει ένας ε, παλαιός θεός των Ρωμαίων, ο Ιανός, με τα δύο πρόσωπα, ο θεός της μετάβασης. Εδώ υπάρχει αυτή η περίπτωση. Τηρούμε το δίκαιο στις Βρυξέλλες και όταν φεύγουμε από τις Βρυξέλλες δεν μας ενδιαφέρει το δίκαιο. Κάνουμε ό,τι θέλουμε. Πλήρης απουσία λογοδοσίας. Δεν αναγνωρίζεται σύγκρουση φορώντων που υπάρχει όταν πέρα από υψηλόβαθμοι υπάλληλοι που υπηρετούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ταυτόχρονα ελεκτέ συμμόρφωση κρατών. Με τι δράσει του παρεμβαίνουν κατά παράβαση των σε τομεί δημοσιονομικού, τομεί υγεία, τομεί παιδεία, κοινωνική πολιτική που δεν του έχουν κορυφθεί από καμία συνθήκη. Με βάση τη μέχρι τώρα δράση του, έχω ζητήσει να, να αυτοαξιολογηθούν. Δεν το έχουν κάνει και περιμένω μια απάντηση. Έχουμε τι παρακάτω πραγματικότητε. Η πατρίδα μου είναι πρώτη στην Ευρώπη στην ανεργία. 20% η επίσημη. Στι γυναίκε 31%. Στου νέου κάτω των 25 ετών 60%. Πραγματικότητα δεύτερη. Πρώτη στην Ευρώπη στην υπογεννητικότητα και μείωση πληθυσμού. Πραγματικότητα τρίτη. Πρώτη στην Ευρώπη στο δημόσιο χρέο. Περίπου 194% του ΑΕΠ. Πραγματικότητα τέταρτη. Πρώτη στην Ευρώπη στη μείωση του ΑΕΠ. Μείον 25% σε καιρό ειρήνη. Στην πατρίδα μου είναι σε εξέλιξη μια λευκή ανέμακτη γενοκτονία. Έχει όνομα μείωση γεννήσεων. Για πρώτη φορά από τη σύσταση του ελληνικού κράτου, πέρα από τη μείωση του ΑΕΠ, τη μείωση των μισθών και των συντάξεων, την υποχώρηση του κοινωνικού κράτου και των κοινωνικών δικαιωμάτων, υπάρχει μείωση πληθυσμού σε επίπεδο 1,34%. Η μείωση του πληθυσμού δεν μπορεί να αναζητηθεί μόνο στη μείωση των γεννήσεων, αλλά και στη μετανάστευση των Ελλήνων πολιτών στο εξωτερικό, σαν αποτέλεσμα τη πρωτοφανού αύξηση ανεργία που ήρθε ω φυσική συνέπεια των μνημονιακών πολιτικών λιτότητα. Παράλληλα και με την βάση την έκθεση τη UNICEF 2013 για την κατάσταση των παιδιών στην Ελλάδα, 700.000 παιδιά υποσυτίζονται. Αυτό που στην πραγματικότητα έχει πετύχει η Τρόικα με τη δράση τη είναι πράγματι πρωτογενέ πλεόνασμα. Αλλά όχι με οικονομικού όρου όπω φαντάζεστε, αλλά με όρου κοινωνικού. Έτσι υπάρχει πρωτογενέ πλεόνασμα απελπισία, αυτοκτονιών, φτώχεια ανεργία και κοινωνικού αποκλεισμού. Ζούμε σε μια χώρα με 1,5 εκατομμύριο ανέργου, 2 εκατομμύρια ημιάνεργους, 40% αύξηση αυτοκτονιών. Το σήμερα είναι καταστροφή, φτώχεια και λιτότητα. Ανύπαρτε κοινωνικέ δαπάνε, φθηνή εργασία. Όλα αυτά κρυμμένα με όμορφε ουδέτερε λέξει. Μεταρρύθμιση, ανταγωνιστικότητα, δημοσιονομική σταθερότητα. Η επιτυχή διακυβέρνηση τη Ευρωπαϊκή Ένωση με βάση τι ανθρώπινε ανάγκε και όχι τι ανάγκε των τραπεζών είναι θέμα προτεραιοτήτων και πολιτική. Αν η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμείνει στα χέρια πολιτικών αμοραλιστών, θα διαλυθεί. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να έχει ω πρότυπο τον τραπεζίτη που εφορμά στην κοινωνία δολοφονώντα την με ούτε τον οικονομικό προτεστατισμό. Η Ευρώπη είναι κουλτούρα, πολιτισμό, ιστορία, αρχέ, διαφωτισμού δεν είναι στην έννοια της ανάθεσης καθηκόντων, όπως ψευδώς ισχυρίζονται, ο σχεδιασμός και επιβολή πολιτικής για θέματα υγείας. Συγγνώμη. Θα παρακαλούσα να σας θυμίσω να είστε λίγο πιο ακριβείς και σύντομος γιατί μας τελειώνει ο χρόνος. Αν θα μπορούσατε να καταλήγετε, ε, θα σας ήμουν ευγνώμων. Σε μια γνήσια δημοκρατική Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι σε αυτή που υπάρχει τώρα με το τεράστιο δημοκρατικό έλλειμμα, οι ενέργειε αυτέ στις οποίε υποπίπτουν κοινοτικοί υπάλληλοι, θα είχαν ονομασίε όπω παράβαση καθήκοντος, κατάχρηση εξουσία, βαριά παραβίαση του κοινοτικού δικαίου. Και κανονικά θα έπρεπε οι υπάλληλοι τη Τρόικα αλλά και όλοι όσοι κρύβονται από πίσω του να ελέγχονται δικαστικά για πράξει και παραλήψει. Και όχι να είναι ελεκτέ και τιμητέ. Ένα από τα πρώτα πράγματα που μαθαίνουν οι φοιτητέ στι οικονομικέ επιστήμε είναι ότι η οικονομική επιστήμη είναι επιστήμη των επιλογών. Εδώ βλέπουμε μια και μοναδική επιλογή. Λιτότητα χωρί τέλο καταλήγω σε ένα κείμενο, θα είμαι πολύ σύντομος κύριε Πρόεδρε, σε ένα κείμενο στις Βρυξέλλες Ευρωπαίοι διπλωμάτες αλλά και εκπρόσωποι του ιδιωτικού τομέα αναφέρουν. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο αλαζονική, η μυστικοπαθή σε σημείο σαδισμού είναι η συμπεριφορά των στελεχών τη Επιτροπή. Ανέφερε χαρακτηριστικά διπλωμάτης μικρή ευρωπαϊκής χώρας, Προσθέτοντα πως λειτουργούν με εσκεμμένα δυσνόητες διαδικασίε, ώστε κανεί από του υπόλοιπου να μην μπορεί να καταλάβει τι συμβαίνει το μοτίφ τη αλαζονία συναντά κανεί όλε τι συζητήσει με ευρωβουλευτέ, ε, δημοσιογράφου που καλύπτουν την Ευρωπαϊκή Ένωση και επισκέπτε εξ Αθηνών. Εξίσου σαφή είναι πάντω και η υπεροψία των εργαζομένων τη Επιτροπή έναντι των μελών του Κοινοβουλίου. Η πλειονότητα των Ευρωβουλευτών τονίζει χαρακτηριστικά ανώτερο αξιωματούχο Επιτροπή είναι πολιτική δεύτερη και τρίτη κλάση. Τα παραπάνω αφορούν την Επιτροπή με τον κύριο Ζακ Σαντέρ. Αλλά μπορούν κάλλιστα να αναφέρονται και στο σήμερα. Άκρινα από τη στάση των γραφειοκρατών υπαλλήλων απέναντι σε κράτη. Έχετε ευρύτερη, έχετε ευρύτερη νομιμοποίηση, αφού είστε εκλεγμένοι σε σχέση με του γραφειοκράτε υπαλλήλου που είναι διορισμένοι. Για να μην μείνουν στα χαρτιά οι διαπιστώσει των ψηφισμάτων σα, αναλάβετε εντονότερη δράση. Παρότι υπάρχει νέα επιτροπή, οι δράσει και ενέργειε τη Τρόικα δεν έχουν αλλάξει το παραμικρό, το οποίο σημαίνει ότι οι πολιτικέ λιτότητα παραμένουν κυρίαρχε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι ατομικέ ελευθερίε και τα κοινωνικά δικαιώματα αποτελούν τι βάσει τη Ένωση. Άρθρο 2 τη Συνθήκη Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε μια ευνομούμενη και με γνήσια δημοκρατική διάρθρωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έπρεπε να ελέγχει την Τρόικα και όχι να συμμετέχει σε αυτήν. Υπάρχει τεράστιο δημοκρατικό έλλειμμα όταν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι σκόπιμα εκτό τη λήψη αποφάσεων για τα θέματα που συζητάμε. Η άποψη ότι τα δικαιώματα κοστίζουν είναι σαφρή η παραβίασή του κοστίζει πολύ περισσότερο γιατί πλήττει το ανθρώπινο αδυναμικό τη χώρα μου. Διαβρώνει το δημοκρατικό χαρακτήρα τη ιδιότητα του πολίτη. Και τέλο, η έννοια τη Ευρωπαϊκή Ένωση του Ευρωπαίου πολίτη καθίσταται ένα ζήτημα αδιάφορο. Ο πολίτη γυρίζει την πλάτη στην Ένωση. Μια Ευρωπαϊκή Ένωση στην οποία οι άνθρωποι δεν έχουν πια κανένα συμφέρον θα καταρρεύσει. Σα ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ήθελα να σα ευχαριστήσω, αλλά δεν έχουμε ώρα τώρα, δεν έχουμε καιρό πρέπει να, να, να συνεχίσουμε να δουλεύουμε. Uh, well, I would like... λοιπόν, θα ήθελα να απευθυνθώ τώρα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Καπριέλη Τζούντιτσε, έχετε το λόγο. Thank you, Um... Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον αναφέροντα θέτει πάρα πολύ σημαντικά ζητήματα στις σχέσεις ε, μιας χώρας με τις άλλες χώρες εταίρους της ε, που κάνουν μια προσπάθεια αλληλεγγύης ε, όταν η Ελλάδα πέρασε από πάρα πολύ μεγάλες δυσκολίες. Πολλά είναι τα επιχειρήματα που προέβαλε ο αναφέρον. Το ένα έχει να κάνει με την νομική ουσία, αλλά υπάρχουν και άλλα ουσιαστικά θέματα που δεν είναι νομικά. Ας αρχίσω από το νομικό για να ξεκαθαρίσουμε πού βρισκόμαστε. Όντως, καταρχάς θα πρέπει να εκτιμήσουμε το ρόλο της δράσης της Ελλάδας και των άλλων κρατών μελών στο πρόγραμμα οικονομικής βοήθειας και ποια νομοθεσία εφαρμόζεται σε αυτή την περίπτωση. Στην περίπτωση του Μνημονίου Συνεννόησης, Memorandum of Understanding, που είναι το προαπαιτούμενο, ε, ως αντάλλαγμα της οικονομικής βοήθειας που παρέχεται στα κράτη-μέλη, υπάρχουν μέτρα που έχουν συμφωνηθεί με τους δανειστές και αυτά είναι εκτός ε, της ε, κοινοτικής νομοθεσίας. Ε, ε, είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών και κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να συμμορφούνται προς τις υποχρεώσεις. Και σύμφωνα με το χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων, αυτό αφορά τα κράτη-μέλη όταν εφαρμόζουν κοινοτικό δίκαιο. Είμαστε σε ένα πλαίσιο εκτός του κοινοτικού δικαίου και την ευθύνη φέρουν ακέραια τα κράτη-μέλη. Αυτό δεν σημαίνει ότι ε, δουλεύουν και σε ένα νομικό κενό ή στον αέρα και δεν πρέπει να εφαρμόζουν καθόλου θεμελιώδη δικαιώματα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι δεσμευμένη να εξασφαλίζει ότι όταν εφαρμόζεται κοινοτική νομοθεσία από τα κράτη-μέλη θα πρέπει αυτά να σέβονται ταυτόχρονα το χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Στα πλαίσια αυτά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαμεσολαβεί μεταξύ των κρατών που παρέχουν τη μακροοικονομική βοήθεια και ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αξιολογήθηκε και στην υπόθεση Pringer, Springer. Ε, είναι αντίστοιχη ε, περίπτωση και ξεκαθαρίζει ε, το ρόλο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν έχουν καμία εξουσία Απλώ ε, απλώς ισχύουν αυτά που σας είπα προηγουμένω. Τώρα, επί τη ουσία, πέρα από το νομικό θέμα, τι λέγει ο Ναφέρον και τι αποδίδει ε, πολλά από τα δεινά ε, τα φλιβερά γεγονότα που έγιναν στην Ελλάδα την τελευταία δεκαετία το, αποδίδει στην Τρόικα και στα θεσμικά όργανα γιατί η Τρόικα δεν υπάρχει ουσιαστικά ως όργανο αλλά θα, θέλαμε να θυμίσουμε ότι η κατάσταση έφτασε ως εδώ μετά από πολλά χρόνια ατυχών πολιτικών και, και ε, πολιτικών εξελίξεων που οδήγησαν σε μεγάλες ανισορροπίες στα φορολογικά, στα δημοσιονομικά, στη σώρευση χρέους, εξωτερικά, ε, ε, ίσως που δεν ήταν σε ισοσκελισμό ε, και δεν υπήρχε καμία δυνατότητα άσκησης κοινωνικής ή άλλης πολιτικής από το κράτος. Γι' αυτό χρειάστηκε η χώρα να υποστεί μια πάρα πολύ μεγάλη προσαρμογή και αυτό διευκολύνθηκε με οικονομική βοήθεια. Γιατί αν δεν υπήρχε αυτή η οικονομική βοήθεια θα ήταν άτακτη χρεοκοπία και ε, τα προβλήματα θα ήταν πολύ μεγαλύτερα και τα κοινωνικά και οι αρνητικές συνέπειες εν γέννη. Βεβαίως έχουμε επίγνωση και γνώση των γεγονότων και ε, Συμμεριζόμαστε τις ανησυχίες για τις δυσκολίες, τις προκλήσεις και τα δεινά που έχει υποστεί ο λαός. Είδαμε να αυξάνεται και η ανεργία και η φτώχεια, αναφέρατε κάποια στοιχεία και κάποια γεγονότα που δυστυχώς είναι αυτά και δείχνουν οι αριθμοί πόσο μεγάλη είναι η δυσκολία που αντιμετωπίζει η χώρα, αλλά δεν σημαίνει ότι η πολιτική ε, ε, που ακολουθεί η Τρόικα ήταν η αιτία, ούτε ότι δεν προσπάθησε να αντιμετωπίσει. Από την ανεργία, ας πούμε, ή το δίκτυο κοινωνικής προστασίας. Μα δεν υπήρχε αυτό στη χώρα, ούτε επιδόματα ανεργίας, ούτε μια ελάχιστη κοινωνική προστασία. Γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μαζί με τα άλλα θεσμικά όργανα και το κράτος μέλος την Ελλάδα προσπάθησε να δημιουργήσει αυτό το δίκτυο κοινωνικής προστασίας, ιδιαίτερα Πρόσφατα, μετά από πολλά έτη συζητήσεων, για πρώτη φορά υπάρχει ε, το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα ως πιλωτικό πρόγραμμα, ε, το οποίο θα αρχίσει να εφαρμόζεται, ελπίζουμε, του έτους. Εάν συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια και θα ε, είναι ευεργετική για όλη την κοινωνία. Επίσης, για την αντιμετώπιση της ανεργίας. Ε, ε, υπάρχουν προγράμματα για την νεολαία, για τους ε, νέους, για τους ανέργους που είναι βραχυχρόνια, μακριχρόνια, άνεργοι. Προσπαθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συντονίζει και να διευκολύνει και τη δουλειά της κυβέρνησης όσο αυτό είναι δυνατό. Υπήρξαν και άλλα στοιχεία στα οποία αναφέρθηκε, αναφέρω, και για θέματα συντάξεων ε, που έπρεπε να λάβει η κυβέρνηση. Είναι ευθύνη της κυβέρνησης ε, που ασκεί τις πολιτικές, τις αποφασίζει, τις φέρνει στο κοινοβούλιο και στη συνέχεια τις εφαρμόζει με τα άλλα θεσμικά όργανα. Χρειαζόταν συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση γιατί ήταν πολύ μεγάλο το, το ποσοστό του ΑΕΠ που πήγαινε στις συντάξεις και το χρέος αυξανόταν με μεγάλους ρυθμούς. Χρειάζεται απλούστευση και διαφάνεια όσο γίνεται στο σύστημα, μεγαλύτερη δικαιοσύνη και στοχευμένα επιδόματα για τους ανθρώπους που χρειάζονται περισσότερο παροχές. Βεβαίως τώρα, έτσι όπως έχει η κατάσταση, χρειάστηκαν να γίνουν πολλές οικονομίες, πολλές περικοπές στις δαπάνες, αλλά έγινε και μια προσπάθεια, μια απόπειρα οι περικοπές αυτές να πλήξουν τα πιο ευάλωτα στρώματα του πληθυσμού, τους πιο φτωχούς και τους πιο στερημένους και για τους συνταξιούχους. Η προσαρμογή στράφηκε προς ε, υψηλοσυνταξιούχους, ας πούμε, ή εκείνους που είχαν πολλαπλές συντάξεις και όχι προς τους χαμηλοσυνταξιούχους. Έτσι και η κατάσταση είναι οδυνηρή για όλο το λαό. Ε, αλλά προσπαθήσαμε όσο γινόταν να ε, κάνουμε έτσι την προσαρμογή. Σας είπα, όλα αυτά ήταν μετά από διαπραγμάτευση και συνεννόηση με τις ελληνικές αρχές. Εκείνες φέρουν την ευθύνη της εφαρμογής και της υλοποίησης. Τα τελευταία χρόνια κάναμε αυτή την προσπάθεια και συνεχίζουμε τώρα να εφαρμόζουμε τις πολιτικές. Η αναφορά αυτή είναι λίγο παλαιότερη Πέρυσι έπλησε το τέλος της ύφεσης και το 2014 κανονικά δημιουργήθηκαν 100.000 θέσεις εργασίας, μειώθηκε σιτά η ανεργία παρόλο που είναι ακόμα γύρω στο 26%. Αυτό είναι ένα θέμα αναδιανομής των πόρων γιατί μεγάλο τμήμα του πληθυσμού ε, απασχολείται σε τομείς που δεν ήταν παραγωγικοί ε, γι' αυτό και τώρα πρέπει να γίνει αυτή η μετατόπιση. Προσπαθούμε να υποστηρίξουμε τη μεταρρύθμιση και τη μετάβαση όσο γίνεται με τα κοινοτικά ε, μέσα και εργαλεία που διαθέτουμε. Και θα έρθουν τα αποτελέσματα και τα ευεργετήματα σύντομα. Θα είναι πιο ορατά. Σε ό,τι αφορά αυτό που ε, είπε ο αναφέρον, με πολλές αναφορές και παραπομπές, εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να ε, συνιστούν παραβίαση του χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων και θεωρούμε ότι αυτό παραμένει. Με μεγάλη προσοχή ε, θα παρακολουθούμε την κατάσταση και είμαστε πρόθυμοι να συζητήσουμε και με τις ελληνικές αρχές και με τα άλλα θεσμικά όργανα για να αντιμετωπίσουμε τέτοια ζητήματα στο βαθμό που θα εμφανιστούν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω το λόγο στους αδέλφου, Ο κύριος Μαριάς πρώτος και μετά η κυρία Άουκεν. sorry. Ε, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Σήμερα πραγματικά μου δίνεται μια ευκαιρία να τοποθετηθώ εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για αυτό το σοβαρό ζήτημα της Τρόικας. Βρέθηκα σαν Ευρωβουλευτής ακριβώς επειδή πήρα μια συγκεκριμένη δέσμευση πολιτική ότι θα έρθω εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αναδείξω τρία ζητήματα. Πρώτον, την ευθύνη που έχει η ίδια η Τρόικα για την καταστροφή στην Ελλάδα. Δεύτερο, ότι πρέπει να υποχρεωθεί να αποζημιώσει και την Ελλάδα αλλά και διάφορους πολίτες για αυτή την καταστροφή. Και τρίτον, ότι δεν πρέπει να ξαναγίνει αυτό που έγινε στην Ελλάδα αλλού. Και στην πολιτική δεν ε, μπήκα επειδή ξεκίνησα ένα αγώνα στην Ελλάδα από το 2010 με πάρα πολύ λίγους την εποχή εκείνη καθηγητές απέναντι στην Τρόικα. Διότι το επάγγελμά μου είναι καθηγητής θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό που είδα ήταν να παραβιάζεται η συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την ίδια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γι' αυτό και από το 2011, κυρία Πρόεδρε, έχω γράψει αυτό εδώ το βιβλίο, το οποίο εξηγεί αναλυτικά πώς έγινε η παραβίαση της συνθήκης στην Ελλάδα. Με απλά πράγματα για τους κυρίους της Κομισιόν που κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν. Πρώτον, με την απόφαση για την δίθεν στήριξη της Ελλάδας εκχωρήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το δικαίωμα να εκπροσωπεί τα κράτη-μέλη ως δανειστές έναντι της χώρας. Επομένως η Επιτροπή ως μέλος της Τρόικας ενεργεί ως εκπρόσωπος των δανειστών. Αυτό να το ξεκαθαρίσουμε. Αυτό δημιουργεί μια τεράστια αντίφαση. Διότι η Επιτροπή υποτίθεται ότι υπάρχει για να υποστηρίζει το κοινό συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα και τα δικαιώματα των πολιτών. Ταυτόχρονα, επειδή πρέπει να ενεργεί ως εκπρόσωπος των δανειστών, αυτό αναφέρεται στο πρώτο μνημόνιο και αυτό αναφέρεται και στην πρώτη δανειακή σύμβαση Ελλάδας χωρών Ευρωζώνης, όσον εκπροσωπεί τους δανειστές πρέπει να πάρει τα λεφτά τους. Δηλαδή να επιβάλλει τις πολιτικές που είναι σκληρές για να μπορέσουν κάποτε οι δανειστές να πάρουν τα λεφτά τους. Δεύτερο, λέει ότι το μνημόνιο είναι μια σύμβαση μεταξύ της Ελλάδας και των δανειστών και δεν ξέρει τίποτα η Επιτροπή. Να σας πω λοιπόν το εξή στους κυρίους. Κάθε μνημόνιο περιλαμβάνει αναλυτικά 50 και 80 και 100 σελίδες τι μέτρα πρέπει να εκτελέσει η Ελλάδα διαφορετικά δεν θα πάρει τα δανεικά από τους δανειστές. Σε αυτά τα μέτρα περιλαμβάνονται αποφάσεις για μισθούς, για συντάξεις, για κοινωνικό κράτος, που είναι εκτός των αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ρωτώ, έχει δικαίωμα η Επιτροπή να παρεμβαίνει σε αυτά. Όχι. Αλλά σου λέει, μα αυτό δεν είναι κοινοτικό δίκαιο. Κύριοι της Επιτροπής να πείτε την αλήθεια. Μετά από κάθε μνημόνιο, κυρία Πρόεδρε και αυτό είναι σημαντικό, η απόφαση του μνημονίου ενσωματώνεται σε απόφαση του ΕΚΟΦΗΝ και δημοσιεύεται στην εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Δηλαδή γίνεται απόφαση του ΕΚΟΦΗΝ, δηλαδή γίνεται κοινοτικό δίκαιο το οποίο αναφέρει αναλυτικά κάθε φορά πόσο θα είναι η μισθή, αν θα μειωθούν οι συντάξεις, αν θα πουληθούν οι εταιρείες για τα ύδατα κλπ. Επομένω, εδώ είναι κοινοτικό δίκαιο και εδώ παρεμβαίνετε με βάση το κοινοτικό δίκαιο. Άρα έχετε ευθύνη διότι αν αποδειχτεί παραβίαση του κοινοτικού δικαίου τότε έχετε ευθύνη τεράστια. Σας λέω λοιπόν και αυτή είναι η πραγματικότητα και θα φέρω και ντοκουμέντα γιατί εγώ δεν θα σταματήσω την υπόθεση αυτή μόνο με αυτή την αναφορά θα συνεχίσω αυτόν τον αγώνα. Δεύτερο θέμα. Ο νόμος, διότι τα έζησα αυτά, ο νόμος ο πρώτος του μνημονίου είναι ο 3845. Αυτός ο νόμος, γιατί λέει το ελληνικό κοινοβούλιο τον ψήφισε. Αυτός ο νόμος έχει τρία άρθρα. Ένα άρθρο που συστήνει τον δίθεν μηχανισμό στήριξης, δεύτερο άρθρο όλο το μνημόνιο και τρίτο άρθρο τους ελληνικούς νόμους που εφαρμόζουν το μνημόνιο. Επομένως το μνημόνιο ενσωματώθηκε στην Ελλάδα διότι είπε η Τρόικα ή θα κάνετε αυτά που θέλουμε ή δεν θα πάρετε χρήματα. Και επειδή επί δύο χρόνια ήμουν βουλευτής στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, κάθε φορά ερχότανε και έλεγαν 19 Δεκεμβρίου του 2012, δύο, τελειώνω, δύο μέρες πριν τα Χριστούγεννα, ή θα ψηφίσετε αυτούς τους νόμους ή αλλιώς η Τρόικα δεν σας δίνει λεφτά. Και έτσι η πλειοψηφία του Ελληνικού Κοινοβουλίου, εγώ διαφωνούσα, πιεζόμενη ψήφιζα αυτά. Δεύτερο θέμα. Πού πήγαν τα λεφτά. Γιατί είπαν για αλληλεγγύη. Ξέρετε ότι η Ελλάδα πήρε μέχρι σήμερα 215 δισεκατομμύρια ευρώ σε πέντε χρόνια. Είναι δυνατόν μια χώρα να πάρει 215 δισεκατομμύρια ευρώ δανεικά και να έχει 1,5 εκατομμύριο ανεργούς. Είναι δυνατόν να έχει χιλιάδες κλειστά μαγαζιά. Ρώτησα τον κύριο Κατάινεν. Πού πήγαν τα λεφτά κύριε Κατάινεν και μου απάντησε εδώ στο κοινοβούλιο, δεν ξέρω. Θα σας πω εγώ, I'm going to finish right now. Και είπε, δεν ξέρει που πήγαν τα λεφτά, θα σας πω εγώ που πήγαν τα λεφτά. Δεν διασώθηκαν οι Έλληνες, φτωχοποιήθηκαν. Απλά 150 δισεκατομμύρια ευρώ από τα 214 πήγαν στα ομόλογα των ξένων τραπεζών και σώθηκαν οι ξένες τράπεζες, οι γερμανικές, οι γαλλικές κλπ. 50 ναι. Madam President, I'm going to finish really. 50 δισεκατομμύρια πήγαν για να σωθούν οι Έλληνες ολιγάρχες. Εκεί πήγαν τα λεφτά. Και τέλος, τέλος. Αυτή είναι ευθύνη μόνο της Ελλάδας. Ήξερε η Ευρωπαϊκή Ένωση τι έκανε. Διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, κύριοι, έχετε μια αρμοδιότητα να ελέγχετε την Ελλάδα. Εφόσον υπερεύει, εφόσον είχε ελλείμματα, τι κάνατε. Θα σας πω εγώ τι είπε ο κύριος Γιούνκερ. Και αυτό το δήλωσε το 2010, αλλά επειδή ήθελα να ήμουν δίκαιος απέναντί του, όταν ήρθε εδώ για να είναι υποψήφιος πρόεδρος και ήρθε στο ECR, τον ρώτησα και του διάβασα αυτή τη δήλωση και την επιβεβαίωση. Ακούστε λοιπόν τι είπε ο κύριος Γιούνκερ. Είπε, οι Ευρωπαίοι γνώριζαν ότι κάποια μέρα η Ελλάδα θα πρέπει να αντιμετωπίσει τη δημοσιονομική κρίση. Και συνέχισε ο κύριος Γιούγκερ. Ήταν φανερό ότι η Ελλάδα θα έπρεπε να αντιμετωπίσει το πρόβλημα και ήξερα, δηλαδή ο κύριος Γιούγκερ ήξερε το πρόβλημα, το συζητούσα, είπε ο κύριος Γιούγκερ, με τους Γερμανούς, τους Γάλλους, τον Τρισέ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και εγώ ίδιος συζητούσαμε λέει για τις προοπτικές αυτές που δεν ήταν γνωστό που αποκαλούμε κρίση. Και λέει ο Γιούγκερ, ήξερα ακόμη ότι η Γαλλία και η Γερμανία κέρδιζαν τεράστια ποσά της τις εξαγωγές στην Ελλάδα. Αλλά εγώ, δηλαδή ο Γιούνκερ, δεν μπορούσα να πω δημόσια τι ήξερα. Επομένως, ο κύριος Γιούνκερ και όλοι σας ξέρατε ότι υπερχρεώνεται η Ελλάδα. Απλά με την υπερχρέωση κέρδιζαν οι γερμανικές, οι γαλλικές και οι άλλες επιχειρήσεις. Αυτή η υπερχρέωση, αυτή η υποχρέωση ονομάζεται odious debt επονίδιστο χρέος και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο πρέπει να διαγραφεί. Can point out that we are dealing... Θα ήθελα να πω ότι ασχολούμαστε με μια συγκεκριμένη αναφορά, όχι γενικά δημόσια συζήτηση εδώ. Αναφορά, άκουσα αυτά που είπε ο αναφέρον, είναι εντός της αναφοράς η οποία είναι 50 σελίδες. So ραγίζει και η καρδιά μου όταν βλέπω πως υποφέρουν οι Έλληνες. Αλλά τώρα έχουμε αυτή τη στιγμή, δεν έχουμε η ώρα για ε, okay. μεγάλο. Well, I am on the specific petition, because this petition is... Τοποθετούμε σε αυτή τη συγκεκριμένη αναφορά. Η αναφορά είναι 50 σελίδε Τη διάβασα λοιπόν και αναφέρομαι ακριβώ σε αυτή την αναφορά. Στα νομικά ζητήματα τα οποία έφυξε η Κομισιόν και σε άλλα ζητήματα. Κύριε Μαριά, διακοπτή πρόεδρος, αναφέρεστε και κατονομάζετε συγκεκριμένα άτομα τα οποία δεν βρίσκονται εδώ. Μπορείτε να τα καλέσετε εδώ, λέει ο κύριος Μαριάς, για να συζητήσουμε. Δεν μπορούμε να τους καλέσουμε και δεν είναι ούτε η ώρα ούτε το μέρος ε, για μια συζήτηση για τον κύριο Γιούμ και την κυρία Μέρκελ για ναι, άλλους. Θα μου δώσετε ένα λεπτό να ολοκληρώσω. Σα δίνω 10 δευτερόλεπτα. Δώστε μου 24 στον μπάσκετ. Πέτρε, τα θέματα είναι έτσι όπως τέθηκαν. Υπάρχει παραβίαση του κοινοτικού δικαίου, υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, γι' αυτό είχα θέσει εδώ τις τροπολογίες για να πάει υπόθεση στον Όμπουτσμαν. Καταγγέλλω την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα που δεν τόλμησε να έρθει και επιφυλάσσομαι να συνεχίσω κι εγώ τον αγώνα μου και εδώ και σε άλλες επιτροπές διότι ήρθε η ώρα οι κύριοι της Επιτροπής να αποζημιώσουν τον ελληνικό πληθυσμό για τη ζημιά που ανέρχεται σε πολλές εκατοντάδες δισεκατομμύρια ευρώ. Thank you very Εγώ σας ευχαριστώ και ήρθε και η ώρα σας τώρα. <laughs> To conclude, wonderful. Now, next, next speaker on my list. Ο επόμενος ομιλητής. Τώρα είναι η κυρία Όχιν. Σύμφωνα με τον κατάλογο των απαραίτητων. Αυτό θα ήταν ε, κάπως επικίνδυνο. Ρισκάραμε αυτό που θα σας πω τώρα. Αλλά πάντως μετά από τις ε, εκλογές ίσως θα μπορούσαμε να θέσουμε κάποια ερωτήματα για την ε, Ελλάδα. Γιατί η πράσινη επικρίναμε την Τρόικα και επικεντρωθήκαμε τόσο πολύ στην λιτότητα και λοιπά και υπάρχει και επίσης ε, όλη αυτή η υπόθεση που έχει τονίσει και ο Δημοσιοδής αλλά το θέμα είναι τώρα να δούμε τι γίνεται με το θύμα στην Ελλάδα γιατί κάποιοι από εμά έχουμε διαπιστώσει πάρα πολύ μεγάλη διαφθορά και καμία καμία θέληση να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο. Να, παράδειγμα πριν από ένα χρόνο ασχολούμουν με την φαρμακοβιομηχανία και οι μεγάλες εταιρείες κατάφεραν να χειραγωγήσουν όλο το δημόσιο τομέα και τους γιατρούς στην Ελλάδα. Οπότε δεν συνταγογραφούν για νόσημα. Άρα ποιος ωφελήθηκε, όχι ο κόσμος, όχι ο κόσμος. Δημοκρατία έχετε. No, you have elected the people τώρα, in the democracy and you should stop being the victim and start to... Και θα πρέπει να σταματήσετε να παίζετε το θύμα και να μπορέσετε να καθαρίσετε αυτό, αυτή, όλο το σκουπιδοντενικέ της διαφθοράς. Listen, I guess... Ακούστε λέει ο Πρόεδρος. Νομίζω ότι όλοι είμαστε κάπως κουρασμένοι τώρα. Δεν έχουν ζητήσει άλλοι το λόγο. Και είμαι πάρα πολύ κουρασμένη κι εγώ. Και να σου πω την αλήθεια, δεν έχω ακούσει και πολλές προτάσεις. Άρα, να κάνουμε το εξής. Να ξαναδώσουμε το λόγο στον αναφέροντα, αλλά παρακαλώ και εσείς να αντιδράσετε στο εξής. Όχι, με τίποτα να μην κλείσουμε αυτήν την αναφορά, μια που έχουμε εδώ Έλληνες συναδέλφους. Επομένως, πρέπει να σας πω ότι υπάρχει μια μελέτη από το Τμήμα Μελετών, η οποία τώρα εκπονείται και αφορά τις επιπτώσεις της κρίσης όσον αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα, όσον αφορά την κοινωνία και βρίσκεται στη διαδικασία της ε, ολοκλήρωσης ε, θα την λάβουν. Είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η μελέτη και επίσης σας επισημαίνω ακριβώς το ότι ολοκληρώνεται. Σε λίγες εβδομάδες θα έχει δημοσιευθεί. Στη συνέχεια μπορούμε να επισηρούμε την προσοχή σε αυτή τη μελέτη και μια που η ΕΚΤ δεν παρέστησε σήμερα εδώ μπορούμε να ρωτήσουμε και την Κεντρική Τράπεζα πώς αντιδρά σε αυτή τη μελέτη, ώστε έτσι να υπάρχει μια ένδειξη σεβασμού στον αναφέροντα. Αυτό μπορούμε να κάνουμε. Ή έχετε κάτι άλλο να προτείνετε, κύριε Μαριά. Α, συμφωνώ, συμφωνώ. Ε, πρώτα απ' όλα να παραμείνει ανοιχτή η αναφορά, όχι επειδή υπάρχουν ελληνικά μέλη, αλλά επειδή είναι πάρα πολύ σοβαρή. Δεύτερο, πράγματι αυτή η έρευνα που αναφέρεστε είναι σημαντική Τρίτον, υπάρχει από ό,τι γνωρίζω μια έκθεση που ξεκινά να γίνεται στη Λίμπε για το θέμα της παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ελλάδα με αφορμή την Τρόικα οπότε και αυτό είναι ένα σοβαρό θέμα έτσι έχω ενημερωθεί ότι υπάρχει μια τέτοια πρόταση τέταρτον να κληθεί κυρία Πρόεδρε η κεντρική τράπεζα να έρθει. Όχι να τους στείλουμε μια επιστολή. Να τους καλέσουμε να έρθουν να τοποθετηθούν για το θέμα αυτό. Διότι πρέπει να δείξουν σεβασμό στην Επιτροπή μας. Ας έρθουν να πούνε αυτά τα οποία αβάσιμα έχει πει μέχρι στιγμής η Κομισιόν, αλλά τουλάχιστον η Κομισιόν ήρθε. Και από εκεί και πέρα να δούμε τι άλλες προτάσεις υπάρχουν για το ζήτημα αυτό. Επομένως ας μείνει ανοιχτή και ίσως μια καλή ιδέα θα ήταν κυρία Πρόεδρε να καλούσατε και τη νέα ελληνική κυβέρνηση να έρθει να μας πει τις απόψεις της εδώ για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ. Thank you very much. Well, um, Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, πιστεύω πως αυτό πάει κάπως μακριά. Η δική μου πρόταση είναι να ζητήσουμε μια γραπτή απάντηση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στην αναφορά αυτή και επίσης να κρατήσουμε την αναφορά ανοιχτή και πιστέψτε με, θα υπάρξουν πολλές ευκαιρίες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να μπορέσουμε να δώσουμε προσοχή και την προσοχή που αρμόζει σε αυτό το θέμα. Τι άποψη έχετε, Πίτερ? Δεν είμαστε πολλοί και οι πράσινοι συμφωνούν υπέροχα. Πιστεύω πως θα έπρεπε να πιέσετε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα να έρθει εδώ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν μπορούν να αγνοούν αυτήν την Επιτροπή. Έχουν κέρδος 4 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο από ελληνικά ομόλογα. Και πρέπει να έρθουν εδώ και να παρουσιαστούν ενώπιόν μας. Δεν είναι υπεράνω του νόμου. Κύριε Μαριά, ξέρετε κάτι. Τους καλέσαμε. Τους καλέσαμε ευγενικά, εγκάρδια και Πιστέψτε με, εφόσον δεν εμφανίστηκαν τώρα, δεν θα εμφανιστούν ούτε στο μέλλον. Γι' αυτό και επιμένω να τους ζητήσουμε μια γραπτή απάντηση. Αλλά ίσως ξέρουν ότι θα είστε εσείς εδώ και δεν τολμούν να έρθουν. Ποιος ξέρει να το κάνουμε έτσι μπορούμε και μετά να προχωρήσουμε. I was trying to be a bit funny. Προσπάθησα να κάνω κάποιο αστείο. Κύριος Μαριάς. Και αυτό επίσης αφορά και τις εταιρείε τις οποίες ο κύριος Γιούνκερ ή ε, είχε στο Λουξεμβούργο και αυτές οι εταιρείες διαχειρίστηκαν ελληνικό φορολόγητο χρήμα. Αυτή είναι η αλήθεια. Κύριε Μαριά, δείξτε σεβασμό στον αναφέροντα, ο οποίος έχει τώρα το λόγο. Απλά θα ήθελα να αναφερθώ ε, ότι ουσιαστικά δεν έλαβα απάντηση από τον ε, εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε ό,τι αφορά τις εκθέσεις των διεθνών οργανισμών το προσπέρασε ε, με μια απάντηση ότι παρακολουθούμε γενικότερα τις εξελίξεις και έχουμε μια ανησυχία για αυτά που γίνονται στην Ελλάδα. Επειδή έχω αναπτύξει και κοινωνική δράση στην Ελλάδα, όταν γυρίσω πίσω θα πω στα 700.000 παιδιά που υποσυτίζονται ότι να συμμεριστούν την ανησυχία του εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής και Μπορεί να μην χορτάσουν, αλλά τουλάχιστον είναι καλό που εκφράζεται μια ανησυχία. Είναι καλό αυτό. Ε, σε ό,τι αφορά το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα που είπε ο, ο εκπρόσωπος, ε, ότι δεν υπήρχε ένα ε, ελάχιστο δίκτυ κοινωνικής προστασίας, πρόκειται περί μιας απάτης. Ε, είναι, ένα, εισόδημα, το, είναι, ένα, είναι επίδομα το οποίο ψηφίστηκε πριν από μερικούς μήνες και έρχεται σαν συμπληρωματικό ε, άλλων παροχών που δίνει το κράτος και ο σκοπός του είναι ουσιαστικά να κόψει κοινωνικές παροχές. Ε, δεν είναι τυχαίο ότι μέσω τη ε, ρύθμιση του ελάχιστου κειμένου εισοδήματο, το οποίο είναι και πιλωτικό σε τρει-τέσσερι Δήμου, ε, περιμένουν να έχουν ε, ωφέλεια στι κοινωνικέ δαπάνε, δηλαδή να μειωθούν οι κοινέ δαπάνε και όχι να αυξήσουν. Γιατί σου λέει, άμα πούμε παίρνει δύο-τρία επιδόματα, θα σου δώσω αυτό που είναι το minimum, οπότε δεν παίρνει τίποτα. Είναι γύρω στα 200 ευρώ το μήνα. Ε, συγγνώμη, 200 ευρώ το μήνα. Ναι, 200 ευρώ το μήνα και πρέπει να είσαι τελείω πέννητα για να πάρει αυτό, αυτό το επίδομα στην πράξη θα το πάρουν ελάχιστοι και μόνο οι φοροφυγάδε. Ε, το μόνο σημείο που θα συμφωνήσω με τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής ε, Επιτροπής είναι ότι αυτή, αυτή η κατάσταση προϋπήρχε. Ουσιαστικά κλήθηκαν, ε, κλήθηκε η ελληνική κυβέρνηση με το διάγγελμα από Ανδρέας στο Καστελόριζο να διαχειριστεί μια καυτή πατάτα ή μια φούσκα θέλετε που έσκασε. Και εδώ θα συμφωνήσω με τον κύριο Μαριά ότι οι ευθύνε των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων, Στατιστική Υπηρεσία, Κεντρική Επιτροπή είναι τεράστιες. Έρχονται δηλαδή μετά από τόσα χρόνια απραξίας που δεν κάναν τίποτα με την ρομφαία ε, του Αρχαγγέλου Γαβρίλ και παίρνουν κεφάλια. Δηλαδή δεν κάναν τίποτα, γνωρίζαν ότι υπήρχε παραβίαση του κοινοτικού δικαίου από την Ελλάδα, γνωρίζαν ότι δεν υπήρχε, το, τα, τα στατιστικά στοιχεία ήταν ψευδή. Δεν υπήρχε τίποτα. Και έρχεται τώρα να παραστάνουν του τιμητέ και να πούνε τώρα θα μαζέψουμε την κατάσταση. Και τι κάνανε τόσα χρόνια. Λοιπόν, και κλείνω ότι για μια ακόμη φορά όλα αυτά δεν είναι ευθύνη της ελληνικής κυβέρνησης. Όλα αυτά τα δάνεια ως γνωστόν δίνονται με, την, με τον ορισμό της αιρεσιμότητας. Θα κάνεις αυτά για να πάρεις τα δάνεια. Δεν τα κάνεις, δεν μπαίνει τα δάνεια. Και αυτός που επιβλέπει αυτά είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Για το δούνο του δεν έχουν από τίποτα, είναι η δουλειά τους, αυτή η δουλειά κάνουν. Δίνουν δάνεια με όρους. Δυστυχώ όμως και η Τρόικα που προέρχεται από την ρωσική λέξη ε, κάρο που το σέρνουν τρία άλογα, ε, ουσιαστικά σέρνει την Ελλάδα και τα κοινωνικά δικαιώματα στον κρεμό. Αυτή είναι η πικρή πραγματικότητα. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας, ε, σας ευχαριστώ. Αλλά τώρα από δύο μέρες έχετε καινούργια κυβέρνηση. Τώρα θα δούμε τι θα κάνουν. Ναι, αυτό και, και ευχαριστώ μου δίνετε την ευκαιρία να χαιρετήσω <laughs> και την ε, σε ελληνική κυβέρνηση, δικοματική και λοιπόν, ελπίζω, λοιπόν, ελπίζω να γίνει κάτι καλύτερο. Τώρα. Ελπίζω. And let's move to the next petition, which is Πάμε τώρα στην επόμενη αναφορά που είναι κάτι παρόμοιο. Είναι αυτή που αφορά τη Συμφωνία Διενειοδότησης των ε, Διεθνών Φορέων με την Ελλάδα. Είναι εδώ ο αναφέρον ή αναφέρος. Είναι η αναφερον ειναι η κυρια Μη πήγε ο κύριος Πεδικάρης. Ε, θα δώσω στον καθένα σας από δύο λεπτά. Έχετε το λόγο. Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, αναφορικά με τα νομικά επιχειρήματα της Επιτροπή έχουμε καταθέσει αναλυτικό υπόμνημα με τη θέση. Προσέρχομαι σήμερα εδώ στην έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με την ιδιότητα του Ευρωπαίου πολίτη. Εδώ πιστεύω ότι λειτουργούν οι θεσμοί, η δημοκρατία και ο δίκαιος νόμος. Είμαι Ελληνίδα αγρότησα, γεννημένη το 1948, λίγο μετά την καταστροφή της Ευρώπης από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και από μια χώρα που προσπαθούσε να ανασυγκροτηθεί μετά την κατοχή από τους Ναζί και από την άλλη ζούσε μέσα στο δράμα του εμφυλίου σπαραγμού. Τα παιδικά μας χρόνια ήταν εξαιρετικά δύσκολα σε ηλικία κάτω των 10 ετών αναγκαζόμασταν να προσφέρουμε εργασία αμέσως μετά το τελευταίο μάθημα του σχολείου μέχρι να πέσει ο ήλιος πηγαίναμε στα χωράφια για να βοηθήσουμε στον βιοπορισμό της οικογένειάς μας αλλά και ως εργάτες, παιδιά εργάτες σε άλλους εργοδότες για ένα πενιχρό μεροκάματο 2,5 δραχμών την ημέρα. Δεν μπορέσαμε να μάθουμε πολλά γράμματα Λίγοι άνθρωποι της δικής μας γενιάς κατόρθωσαν να τελειώσουν ένα δημοτικό σχολείο. Αλλά μάθαμε στη σκληρή δουλειά και την οικονομία. Μέσα από στερήσεις και πολλή δουλειά καταφέραμε να αγοράσουμε δικά μας μικρά αγροκτήματα. Χωρίς σύγχρονα εργαλεία και μηχανήματα. Μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 70. Με υπόδειες εργαλεία οργώναμε τα χωράφια μας, για τη σκορά. Κουβαλούσαμε τα βαριά φορτία, νερό για άδρευση στους λόφους των ελαιοδέντρων, τα στάχια των σιδηρών, τον καρπό της ελιάς για τα λετριβία, οι άνδρες στην πλάτη τους, οι γυναίκες στο κεφάλι. Άλλωστε οι καλλιέργειες στον τόπο μας, στο νησί μου, δεν σταματούν ποτέ. Το επάγγελμα του αγρότη απαιτεί να βρίσκεται στο χωράφι κανείς με κάθε καιρό. Δεν έχει καμιά σημασία αν είναι ο κάψανος του καλοκαιριού ή η βροχή και το κρύο του χειμώνα. Ο αγρότης της δικής μου γενιάς ήταν αναγκασμένος να είναι στο χωράφι του. Δουλεύοντα από το πρωί μέχρι το βράδυ, κερδίζαμε έντοιμα ένα εισόδημα για να ζήσει η οικογένειά μα. Πολλοί πιστεύουν ότι δεχτήκαμε μεγάλη βοήθεια μέσα από τι επιδοτήσει τη πολιτι... ελληνική πολιτεία και τη ΟΚ. Αλλά όπω ίσω γνωρίζετε, αυτό δεν αφορά τους μικρούς αγρούς, αφού οι επιδοτήσεις μέχρι και πρόσφατα ήταν αναλογικές και στην Ελλάδα το 10% των αγροτών κατέχει το 70% της καλλιεργήσιμης γης. Το 1988 η ελληνική πολιτεία δημιούργησε τον αγαρισμό γεωργικών ασφαλίσεων, που έναντι ασφαλιστικών εισφορών από τους αγρότες ανέλαβε τη συμβατική υποχρέωση να παρέχει σύνταξη στο 65ο έτος της ηλικίας μας. Ο κάθε αγρότης είχε τη δυνατότητα να επιλέξει την κλίμακα, το μηνιαίο ασφάλιστο, που ανταποκρινόταν στην οικονομική δυνατότητα του καθενός μας και στις προσδοκίες μας για το ύψος της σύνταξής μας. Το 2002 οι αγρότες επιτέλους αποκτήσαμε ένα σχεδόν ολοκληρωμένο οργανισμό κοινωνικής ασφάλειας αφού μας δόθηκε πρόταση μέσω του ΟΓΑ και σε ιατροφαρμακευτική περίδαλψη. Όμως δεν υπήρχε καμία άλλη παροχή για τους αγρότες της δικής μας γενιάς. Συνεχής δουλειά και κανένα είδους επίδομα χωρίς να έχουμε δυνατότητα να σταματήσουμε την εργασία μας παρά μόνο για ελάχιστες μέρες μετά τον δοκετό των παιδιών μας. Μάλιστα ήταν σύνηθε την εποχή μας πολλές γυναίκες να γεννούν ακόμα και στα χωράφια. Παρά τι ανοιξότητε, παραμείναμε συνεπεί στι υποχρεώσει μα απέναντι στο ασφαλιστικό μα φορέα. Με τη βεβαιότητα ότι έτσι θα εξασφαλίσουμε έστω μια αξιοπρεπή σύνταξη για τα ύστερα μα χρόνια. Όμω, ξαφνικά λίγε μέρε πριν μα ταλούν οι προσκλήσει για να υποβάλουμε τι αιτήσει μα για συνταξιοδότηση, χωρί καμία διαβούλευση, η ελληνική κυβέρνηση, εκτελώντα τα προαπαιτούμενα του μηχανισμού χρηματοπιστωτική σταθερότητα που βρισκόταν σε πλήρη συνοδισμό με τις κατευθύνσεις που είχε δώσει τόσο ο Επίτροπος για την Νομισματική Πολιτική όσο και το ΕΚΟΦΙΤ, ψηφίστηκε νόμος που μετέφερε το όριο ηλικίας συνταξιοδότηση στα 67 χρόνια, προσαυξάνοντας και τις εισφορέ. Μάλιστα, η αλλαγή αυτή έγινε χωρί να ληφθεί υπόψη το μειωμένο προσδόκιμο των αγροτών που οφείλεται τόσο στη σκληρή φύση της εργασίας μας, αλλά και στο γεγονός ότι για χρόνια χρησιμοποιούσαμε φάρμακα και στεβάρματα που αργότερα η ΕΟΚ και μετά η Ευρωπαϊκή Ένωση απαγόρευσαν καθώς αποδείχθηκαν κακινογόνα ή και προκαλούσαν νομονικές ανομαλίες και εγγένει μεγάλη ζημιά στην υγεία μας. Ειλικρινά δεν πιστεύω πως η οικονομία της Ευρώπης μέρει να σωθεί από μια χούφτα ζαρωμένων και κουρασμένων ανθρώπων που η δουλειά και η υγρασία έχει διαβρώσει τα χέρια μας και τα πόδια μας και υποφέρουμε τα βράδια από πόνους καθώς ζούμε αναγκαστικά ακόμα κοντά στους αγρούς. Όμως, αντίθετα με τα όσα ισχυρίζεται η Επιτροπή, όχι μόνο δεν περιορίστηκα, δεν περισσώθηκε το ασφαλιστικό σύστημα από τις θυσίες που ζήτησε η Επιτροπή και το ΙΣΜΗ, αλλά τα πράγματα έγιναν πολύ χειρότερα το κούρεμα των αποθεμάτων των ταμείων που έγινε παρά τη διαβεβαίωση της ομάδας των κρατών που συμμετέχουν στο ευρώ και στο μηχανισμό σταθερότητας ότι δεν θα πειραχτούν τα ομόλογα του επίσημου τομέα, οδήγησε το ταμείο μας στο να χάσει 600 εκατομμύρια ευρώ. Σήμερα, τρία χρόνια μετά, ακόμη λιγότεροι άνθρωποι ακολουθούν το επάγγελμα του διεργού και ακόμη λιγότεροι μπορούν να καταβάλουν εισφορές στον ΟΓΑ καθιστώντας ακόμη πιο ανασφαλή το μέλλον των συντάξεων στη χώρα μας και ειδικά στον αγροτικό τομέα. Ειδικά μάλιστα όταν έχει διαρριχθεί η σχέση εμπιστοσύνη πολιτών και πολιτείας. Έτσι, τόσο από τη μεριά των αριθμών, αλλά και με βάση τις πανανθρώπινες αξίες, αυτές του σεβασμού και της αξιοπρέπειας του ανθρώπου και της προστασίας του μόχτου που μετεσιώνεται σε περιουσία η συγκεκριμένη ρύθμιση είναι και άδικη και παράνομη, χωρίς να φέρνει κανένα θετικό αποτέλεσμα για την βιωσιμότητα των συντάξεων ή την αύξηση των ευκαιριών στην εργασία στον αγροτικό τομέα. Πόσο μάλλον σήμερα, όταν γενικά τα κόστη είναι μεγάλα, η ανεργία, ναι. ενέργεια, σπορά, ενεργεια σπορα φορολογια κτλ. Συνεπώ, λοιπόν, όπω γενικά έχει αποδεχτεί, έχει αποδεχθεί το ΕΔΑΤ. Το μέρος της σύνταξης που είναι αποτέλεσμα εισφορών αποτελεί περιουσιακό στοιχείο και δεν είναι δυνατό να απαλωτριωθεί. Πάντα θα πρέπει να υπάρχουν μια ισορροπία ανάμεσα στις ανάγκες του ατόμου και στις απαιτήσει του γενικότερου καλού. Όμω, η αύξηση του χρόνου συνταξιοδότηση σε συνδυασμό με τη μείωση του προσδόκιμου ζωή στη χώρα μου την καθιστά ιδιαίτερα επαχθή και άδικη τη συγκεκριμένη ρύθμιση. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Now. Και τώρα έχουμε εδώ όλο αυτό το υλικό στη διάθεσή μας, το ξαναδιαβάσατε, αλλά το έχουμε και εμείς το κείμενο. Να είστε βέβαιοι ότι το έχουμε το κείμενο και θα το μελετήσουμε ε, σε μεγάλο βάθος και με μεγάλη προσοχή. Ε, θα ήθελα τώρα να παρακαλέσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρουσιάσει τις θέσεις για την αναφορά αυτή. Δυστυχώς, θα δω καταλαβαίνεις. Ναι. Η μητέρα σου ε, ήταν εκτενέστατη. Δεν μπορείς να προσθέσεις πάρα πολλά σε αυτά. Οπότε θα προτιμούσα να δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να μην αναφερθώ ξανά σε στοιχεία που κάλυψε η προηγούμενη αναφορά. Έχουμε να κάνουμε με ατομικά αγαθά και ατομικά δικαιώματα, τα οποία έχουν συλλεχθεί κατά την παράδοση των ετών. Το πρόβλημα είναι ότι υπήρχαν πάρα πολλές προσδοκίες που είχε η χώρα και την μη δυνατότητά της να τις ε, εκπληρώσει. Υπήρχε κίνδυνος άτακτης χρεοκοπίας, ενώ αυτή ήταν συντεταγμένη προσπάθεια ε, και αλλιώς τα δεινά θα ήταν πολύ περισσότερα και οι δυσκολίες πολύ μεγαλύτερες. Ε, σε ό,τι αφορά λοιπόν τα επιδόματα, τους μισθούς, ε, τα συνταξιωτικά δικαιώματα ε, και τα λοιπά, ήταν σημαντικό τμήμα αυτό της προσαρμογής. δεν ήταν από ευχαρίστηση που επιβάλλει τη λιτότητα κανείς, αλλά ήταν ανάγκη έτσι ώστε η χώρα να γίνει ελκυστική για επενδυτές, να υπάρχει επαρκής αίσθηση σταθερότητα ότι η ε, οικονομία θα έμπαινε σε μια ισορροπία και θα δημιουργούσαμε νέες θέσεις εργασίας. Από όλων αυτών το κράτος δεν δύναται να χρηματοδοτεί πολλά πράγματα. Οπότε αυτό που είπατε και θα απαντήσω τώρα είναι ότι ε, τα επιδόματα ναι. ε, που σας είχαν υποσχεθεί δεν συνδέονται με τη δυνατότητα που έχει το κράτος να τα πληρώσει, να τιμήσει αυτές τις υποσχέσεις. Και ήταν πολύ μεγάλος ο κίνδυνος αυτός, εξού και το χρέος. Και πρέπει τώρα να εξυπηρετεί και το χρέος και τις υποχρεώσεις στο ιστορικό της χώρας. Αυτή ήταν η πραγματικότητα και αυτό θα έπρεπε να αντιμετωπίσει η χώρα. Γι' αυτό προσπαθήσαμε να εξασφαλίσουμε ότι θα υπήρχε μια ισορροπία ανάμεσα στο ατομικό και το γενικό καλό και μοιραία ε, επλήγησαν ε, ατομικά κάποιοι πολίτες. Είναι δύσκολο σε τέτοιες επίγουσες καταστάσεις να εξασφαλίζεται η αναδιανομή. Ε, ο καθένας επιλέγει ή ελπίζει την καλύτερη δυνατή ανάλυση. Ήταν πολύ μεγάλη η ανάγκη σε εκείνη τη στιγμή και η κυβέρνηση προσπάθησε και σε συνεννόηση μαζί μας να αντιμετωπίσει τα μεγάλα προβλήματα και κοίταξε πρώτα το γενικό ε, καλό, τις γενικές ανάγκες της οικονομίας και αυτό οδήγησε κάποιες προσαρμογές για τον καθένα ξεχωριστά πολίτη, ατομικά δηλαδή. Σε ό,τι αφορά το ρόλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τώρα γενικά και τη θέση μας για το πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις σε επίπεδο κυβέρνησης, θέλω να επανέλθω στην προηγούμενη συζήτηση για να ξεκαθαρίσω το εξής. Έχουμε την απόφαση Pringle. Εκεί ξεκαθαρίσει ότι δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων. Και επομένω με αυτό το προηγούμενο, αυτό το δεδικασμένο τώρα μπορούμε να καλύψουμε τα συμφέροντα των ελληνικών αρχών επί τη βάση της εντολής που έχουμε λάβει από το Eurogroup αλλά βέβαια και ως εκπρόσωποι του Θεσμικού Οργάνου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το 12 εξεδόθη αυτή η απόφαση, ε, οπότε δεν είμαι ενημερωμένο για αυτό στο οποίο αναφέρεται το βιβλίο σε σχέση με τις εξελίξεις, αλλά πάντως θα ήθελα να σας υπενθυμίζω ότι έχουμε και άλλες εξελίξεις σε σχέση με την Τρόικα. Όλα αυτά τα γνωρίζει το Κοινοβούλιο. Αυτά τα έχει αναγνωρίσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στα ψηφίσματά του αξιολόγηση από το Κοινοβούλιο στον αυτό το ρόλο και τη λειτουργία της Τρόικα. Ε, όπως επίσης και τη συμμετοχή της Τρόικας σε συναντήσεις, ε, σε εκδηλώσεις επίσημες ή ανεπίσημες. Φυσικά όλα αυτά θα κρυθούν και θα συνεχιστούν εκεί που πρέπει. Να μην επαναλαμβάνουμε τα ίδια, αλλά πάντως θεωρούμε ότι δεν έχουμε παραβεί την των δικαιωμάτων. Δυστυχώς υποφέρει ο κόσμος. Έχει δυσκολίες ο καθένας. Είναι τόσο περιπλοκή η κατάσταση που απαιτούνται δύσκολες αποφάσεις. Οπότε και εμείς προσδοκάμε από όλες τις ελληνικές κυβέρνησεις να κάνουν κάτι. Έγιναν προσπάθειες να συνεχιστούν και στο μέλλον. Και να δούμε τι θα γίνει το πρόγραμμα, τι θα γίνει για το μέλλον της χώρας. Η Πρόεδρος, σας ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, πρώτος θα λάβει το λόγο κύριος Μαριάς. Παρακαλώ κύριε Μαριά, δύο λεπτά. Η αναφορά έχει σχέση με συνταξιοδοτικά δικαιώματα. Δηλαδή, είχαν δικαιώματα στον ΟΓΑ οι αναφέροντες και εκτιμά ότι όλα αυτά χάθηκαν από τη συμπεριφορά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και από το μνημόνιο. Σύντομα. Πρώτον, το πρώτο μνημόνιο αναφέρει αναλυτικά ότι πρέπει να γίνει μείωση των συντάξεων συμπεριλαμβανομένου και του ΟΓΑ. Βεβαίω λέει η Επιτροπή, μα αυτό είναι εκτός κοινοτικού δικαίου, διότι δεν έχει καμία σχέση το κοινοτικό δίκαιο. Να σας διαβάσω λοιπόν ότι το πρώτο μνημόνιο ενσωματώθηκε στο κοινοτικό δίκαιο με την απόφαση 2010 κάθετος 320 κάθετος Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι στην Official Journal L145 11 έκτου 2010. Εκεί είναι η απόφαση του ΕΚΟΦΗΝ η οποία περιλαμβάνει όλο το μνημόνιο όπου εκεί αναφέρεται και η μείωση των συντάξεων. Άρα εδώ είναι κοινοτικό δίκαιο και είναι ευθύνη της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το κακό αποτέλεσμα που υπάρχει. Τέτοιες αποφάσεις του ΕΚΟΦΗΝ είναι πολλές και έχουν σχέση με τα μνημόνια. Άρα εδώ έχουμε κοινοτικό δίκαιο για να σταματήσει αυτό που λέει αβάσιμα η Επιτροπή. Δεύτερο, λέει η petitioner. Μα έχασε τα δικαιώματά της επειδή ο ΟΓΑ είχε ομόλογα του ελληνικού δημοσίου και με το PSI το οποίο συμφωνήθηκε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης μειώθηκαν κατά 40% ή 53% τα ποσά. Και προσέξτε, όλα τα ομόλογα συμπεριλαμβανομένου του δημόσιου τομέα, του ΟΓΑ των Πανεπιστημίων κουρεύτηκαν, εκτός από τα ομόλογα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Αυτά δεν πειράχτηκαν καθόλου. Λέει λοιπόν η αναφέρουσα, έχασε τα δικαιώματά της, γιατί ενώ θα έπαιρνε σύνταξη στα 65 πήγε στα 67. Γιατί, γιατί πρώτον η ιδιοκτησία του ασφαλιστικού ταμείου που ήταν τα ομόλογα του ελληνικού δημοσίου κουρεύτηκαν με το PSI. Δεύτερον, επιβλήθηκαν τα μέτρα ενάντια στα ασφαλιστικά της δικαιώματα από το μνημόνιο και επικροτήθηκαν αυτά και εγκρίθηκαν από το ΕΚΟΦΗΝ και τώρα λέει κάποιος πρέπει να αποφασίσει και να τη δικαιώσει. Είναι ξεκάθαρη παραβίαση από πλευρά και Επιτροπή, με βάση αυτά που είπα πριν και ξαναλέω, και Κεντρική Τράπεζα και επομένω πρέπει να μείνει ανοιχτή η συγκεκριμένη ε, αναφορά. Πρέπει να κληθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μα πει επίση τι απόψει τη και έχουμε μια σοβαρή υπόθεση πολύ συγκεκριμένη απώλειας δικαιωμάτων με ευθύνη και του προγράμματος στη σύλληψή του. Διότι όταν έχεις περιοριστική πολιτική, περιορισμό της ζήτησης, αύξηση της ανεργίας, τότε έχεις λιγότερες εισφορές, άρα πρόβλημα στα ασφαλιστικά ταμεία. Ευχαριστώ. Thank you very much. Nobody else has thought... Ευχαριστώ πολύ. Θέλει κανείς άλλο το λόγο. Ξέρετε τι θα κάνω τώρα. Θα δώσω το λόγο στον Θεόδωρο, το γιο της αναφέρουσας, και εάν είμαστε τυχεροί θα μιλήσω ειδικά, γιατί αν κατάλαβα καλά σπουδάζει στη Σουηδία κοντά στο μέρος που γεννήθηκα σχεδόν. Έχετε λοιπόν λίγο χρόνο για να ολοκληρώσετε. Είχα την ευκαιρία να σπουδάσω στα αγγλικά, γιατί τα αγγλικά στη χώρα σας είναι σε πολύ ψηλό επίπεδο και χρησιμοποιούνται πολύ. Μπόρεσα λοιπόν να σπουδάσω σε Πανεπιστήμιο τη Σουηδίας στα αγγλικά. Σας ευχαριστώ πολύ μου για την ευκαιρία που μου δώσατε να μιλήσω σουηδικά. Δύο πράγματα θα ήθελα να πω. Διότι οι λεπτομέρειε βρίσκονται στην αναφορά μας. Καταρχάς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρει ότι η συμφωνία ήταν ελεύθερη, διότι νόμος είναι κάτι μόνο κατόπιν συνένεσης. Όμως αυτό δεν ισχύει, γιατί ξέρουμε ότι όταν ο κύριος Παπανδρέου ζήτησε δημοψήφισμα, υπήρξε αντίδραση από την κυβέρνηση και από τις ε, ευρωπαϊκές δυνάμεις και στη συνέχεια αποχώρησε. Υπήρξαν επίσης κινδυνολογίες ότι θα αδειάσουν τα ATM κτλ. Φυσικά όλα αυτά ήταν απειλές και οι απειλές δεν συνιστούν κανένα νόμο και καμία συμφωνία. Όμως, όπως λέει και ο Κικέρονας, Ο πιο σημαντικός νόμος, ο ανώτατος νόμος, είναι εκείνος ο οποίος είναι προς όφελος του λαού. Αλλά και στην Αντιγόνη αναφέρεται κάτι τέτοιο. Βέβαια, πιστεύω ότι η αναφορά συμφωνεί με το πνεύμα του νόμου. Και Και τον 20ο αιώνα η Ευρώπη κατάφερε να προοδεύσει. Ζήσαμε εκτός από τους δύο παγκόσμιους πολέμους μια εποχή διαφωτισμού αν θέλετε. Και είναι κρίμα αυτό να χαθεί. Σας ευχαριστώ πολύ. Πιστεύω πως ε, η αναφορά θα πρέπει να κλείσει, διότι έχουμε και μια άλλη αναφορά ανοιχτή, για την οποία περιμένουμε μια απάντηση. Επίσης θα πρότεινα τη μελέτη που έγινε για αυτήν την αναφορά να τη στείλουμε ε, στις ε, αναφορές που παρέμειναν ανοιχτές. Ο κύριος Μαριάς θέλει το λόγο. Σε κάθαρη αναφορά σε ατομικό επίπεδο. Δηλαδή, εξήγησε η αναφέρουσα την βλάβη που έπαθε η ίδια στο συγκεκριμένο θέμα. Η απάντηση που δόθηκε από την Επιτροπή δεν είναι ικανοποιητική, δεν της δίνει καμιά απάντηση. Ουσιαστικά της λέει δεν φταίει η Επιτροπή να κόψει το λαιμό της, να πάει να βρει το δίκιο της. Δεν νομίζω ότι πρέπει να κλείσει η αναφορά αυτή, πρέπει να μείνει ανοιχτή, πρέπει κατά τη γνώμη μου να κληθεί να έρθει εδώ η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ή να στείλει τις απόψεις της και πρέπει να βρούμε τρόπο με τον οποίο θα δικαιωθεί η αναφέρουσα, επομένως πρέπει να εμπλέξουμε στην αναφορά και την Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων, διότι αυτό είναι ένα σοβαρό ζήτημα. Peter. Ο Πέτερ Γιάρ. Χωρίς μικρόφωνο δυστυχώς δεν είναι αναμένο το μικρόφωνο. Ναι, τώρα το άναψα. Ε, λοιπόν, να συμπληρώσω μόνο κάτι. Τα θέματα που θέτει η αναφέρουσα με βάση τη συνθήκη είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών και στα πλαίσια της οικονομικής κρίσης, της δημοσιονομικής κρίσης, σταθεροποίησης του ευρώ, έγιναν κάποιες διαπραγματεύσεις και αυτές οι διαπραγματεύσεις έγιναν στο Συμβούλιο. Δηλαδή θα πρέπει να απευθυνθούν στο κράτος μέλος του, στην Ελλάδα. Δεν, επειδή εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με την Ελλάδα. Δεν έχω πρόβλημα να παραμείνει ανοιχτή η αναφορά και να ε, ρωτήσουμε τι γίνεται και τι ε, ε, πρέπει να αποφασιστεί. Είναι εσωτερικό το θέμα αυτό, τώρα έχει αλλάξει η κυβέρνηση, αλλά θα πρέπει κάπως να υπερασπιστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εδώ στο συγκεκριμένο η Κομισιόν τι να κάνει, τι να πει. Αν ε, έχει κάποιο αποφασίσει, αυτό είναι το Συμβούλιο ή τα κράτη-μέλη αποφάσισαν ή τα μέλη τη Ευρωζώνη, σε πάση περιπτώσει. Απευθυνθείτε σε αυτού που πήραν αυτή την απόφαση. Γιατί αλλιώ πραγματικά φρούδε ελπίδε και ψεύτικες δημιουργούμε. Ωραία. Αν κατάλαβα καλά λοιπόν Πέτερ, αυτό που προτείνει τώρα εσύ είναι να στείλουμε την αναφορά αυτή και όλο το υλικό που μπορούμε να έχουμε, την μελέτη κτλ και μετά να την κλείσουμε την αναφορά ή όχι. Γιατί είναι εθνική υπόθεση, είναι εθνική αρμοδιότητα. Ωραία. Κοιτάξτε, αν δεν κάνω λάθος, έχουμε στο μυαλό μας το εξή. Ταυτόχρονα, όταν η Ελλάδα ζητούσε δάνεια, δεν ήταν η Ευρωπαϊκή Ένωση εκείνη που την κυνηγούσε να της δώσει λεφτά. Η Ελλάδα ζητούσε δάνεια. Και ταυτόχρονα αρνήθηκαν να μειώσουν τις δαπάνες ε, για τις, ε, τους εξοπλισμούς και για την Ορθόδοξη Εκκλησία ταυτόχρονα. Ε, οπότε να το συζητήσουμε και αυτό μια στιγμούλα. Ή να μην το συζητήσουμε, δεν ξέρω. Ο κύριος Μαριάς, δεν θα σας ξαναδώσω το λόγο. Θα κάνουμε το εξή μισό λεπτό. Θα αφήσουμε ανοιχτή την αναφορά αυτή, γιατί ξέρω ότι θα επιμείνετε γι' αυτό. Οπότε και μετά θα στείλουμε όλες τις προφορίες που έχουμε στις ελληνικές αρχές τη νέα ολοκένουργια κυβέρνηση ε, με τις καλύτερες ευχές μας για το μέλλον. Συμφωνείτε? Ωραία. Οκ. Okay. Like Μαριάς, θα ήθελα για μισό λεπτάκι να μου δώσετε το λόγο, να σας τα πω στα αγγλικά, ούτως ώστε να μην υπάρξει καμία παρεξήγηση εδώ με τον φίλο Πίτερ Όταν προηγουμένως έλαβα το λόγο, σας εξήγησα ότι η απόφαση όσον αφορά το πρώτο μνημόνιο το βιολοποιήσε αποφάσεις που αφορούν τα δικαιώματα των ε, συνταξίχων ήταν κάτι το οποίο ενσωματώθηκε σε απόφαση του ΕΚΟΦΗΝ με αριθμό 2010 και δημοσιεύθηκε στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 11 έκτου του 10. Επομένως πρόκειται για θέμα το οποίο αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί πρόκειται για απόφαση του Συμβουλίου Υπουργών Οικονομικών. Πρόκειται για απόφαση που υλοποιεί το μνημόνιο και το καθιστά κοινοτικό δίκαιο κινούμαστε επομένω στα πλαίσια του κοινωτικού δικαίου, επομένω θα πρέπει να μείνει ανοιχτή αυτή η αναφορά. Και επίση να ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα. Να ζητήσουμε το Συμβούλιο να προσέλθει. Επίση το ίδιο και η Κεντρική Τράπεζα. Κύριε Μαριά, έχω κουραστεί κάπω. Και εγώ, και εγώ, γιατί είμαι εδώ από το πρωί, λέει ο κύριο Μαριά. Έχω κάτσει για όλε τι συζητήσει. Πρόεδρο, αυτό που θέλω να σα πω είναι το εξή. Ότι ακριβώ αυτό και προτείναμε να μην ανοιχτεί η αναφορά. Είπατε ότι είναι εκτό ε, αρμοδιότητα, αρμοδιότητας, λέει ο κ. Μαριά. Α θα μείνει ανοιχτή επομένω. Ε, μην ξαναρχίσουμε την ε, κουβέντα επί τη ουσία τότε, λέει ο πρόεδρο, αλλά ας κάνουμε ακριβώ αυτό που σα προείπα. Α μην ανοιχτή η αναφορά, ούτω ώστε όλοι να είναι ικανοποιημένοι και α ενημερωθεί αυτή η όλο καινούργια ελληνική κυβέρνηση ε, και με τι ευχέ μα να τα καταφέρει. Μαριά, θα πρέπει να τοποθετούμε επί του θέματο γιατί αφορά το PSI, τη, τη, τη, τη συνεισφορά του ιδιωτικού τομέα όσον αφορά την εξαγορά αυτών των ομολόγων, γιατί η Ευρωπαϊκή Κοινή Τράπεζα ε, δεν έλαβε μέρο. Και εδώ πέρα αυτή η κυρία εκπροσωπεί συγγνώμη, φορέα συνταξιούχων, των οποίων το Ταμείο επέστη αυτό το κούρεμα. Πρόεδρος, να κάνουμε αυτό που σας είπα. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε εδώ και κάνετε όλο αυτό το ταξίδι ούτω ώστε να παραστείτε ε, σε αυτή την πολυτάρχη συνεδρίαση και πρέπει να εξασφαλίσω ότι δεν θα είναι και όλε οι συνεδριάσεις τόσο πολυτάραχες. Τώρα για να δούμε. έχουμε την επόμενη αναφορά, την επόμενη αναφορά που προέρχεται από τον κύριο Ζων Ζανελά όσον αφορά το σύμφωνο σταθερότητα και αφορά και την παραβίαση την ενδεχόμενη των, των δικαιωμάτων του κόσμου για τα εθνικά δικαιώματα και θα δώσουμε τώρα το λόγο τέλος πάντων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Λουίς Ζορσό, ευχαριστώ Πρόεδρε. Η αναφέρουσα ισχυρίζεται ότι η συνθήκη για τη σταθερότητα και τη διακυβέρνηση της ΟΝΕ επιβάλλει γενική λιτότητα στις χώρες της Ευρωζώνης και αυτό με τρόπο δυσανάλογο επηρεάζει τους ευάλωτους πληθυσμούς. Μιλάω πολύ γρήγορα, μάλιστα. Σε βαθμό που να επηρεάζει και να θίγει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και άλλα ε, δικαιώματα θεμελιώδη και τα δικαιώματα των παιδιών καθώς επίσης και των ηλικιωμένων. Και ζητάει απλούστατα να ε, καταργηθεί αυτό το σύμφωνο. Ε, τι λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά κάποιες διευκρινήσεις για την εμβέλεια, το πεδίο εφαρμογή και το είδος της συνθήκης. Είναι μια συνθήκη διακυβερνητική. Την έχουν υπογράψει αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων και δεν είναι ευθύνη των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων να εγκαταληφθεί ή να καταργηθεί. Από την άλλη, δεν υπάρχει όρος της δημοσιονομικής πειθαρχία. Από το 1997 έχει ε, θεσπιστεί, δεν είναι καινούριο και υπάρχουν κείμενα που ενισχύουν κάποια στοιχεία του Συμφώνου Σταθερότητας και επιμένει στην ανάγκη για τα κράτη-μέλη που προσυπογράφουν να ενθανιστούν, να κάνουν κτήμα τους ε, και να μεταφέρουν στο εθνικό δίκαιο αυτή την νομοθεσία για να υπάρξει ε, δημοσιονομική πειθαρχία. Τώρα, οι δυσκολίες που υφίστανται οι ευάλωτοι ε, ε, στις διάφορες κοινωνίες. Στη Γαλλία είναι οι αναφέροντες, που η Γαλλία δεν είναι σε πρόγραμμα, δεν είναι σε μνημόνιο. Ε, είναι πραγματικά λυπηρό το γεγονός, αλλά οι ρίζες είναι πολλές. Δεν είναι μόνο η δημοσιονομική προσαρμογή, είναι απόρρια κρίσης μεγάλης εμβέλειας που διανύει η Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ και καιρό και έχει και πολλές αιτίες ακριβώς για να αντιμετωπίσουμε την κρίση έχει σφίξει το πλαίσιο αυτό, το δημοσιονομικό και ε, της διακυβέρνησης και μία από τις απαντήσεις που έχει φέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αυτή για να ε, μην έχουμε νέα κρίση, για να ε, συμμαζευτούν κάπως τα δημόσια οικονομικά. Επίσης γίνεται λόγος και για ένα ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 18 Ιανουαρίου του 2012 και χαρακτηρίζουν, λέει, τη συνθήκη αυτή, τη σύμβαση, το σύμφωνο, άχρηστο. Δεν λέει κάτι τέτοιο το ψήφισμα, απλώς εκφράζει κάποιες επιφυλάξεις εάν ε, ήταν σκόπιμη αυτή η συνθήκη ή χρειάζεται κάτι διαφορετικό. Ούτε αμφισβητεί τους στόχους. Ίσα ίσα το ψήφισμα θυμίζει ότι η δημοσιονομική πειθαρχία είναι θεμέλιο για την βιώσιμη ανάπτυξη. Τούν το η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γνωρίζει τις ανετικές συνέπειες που έχει η δημοσιονομική προσαρμογή και έχει λάβει μέτρα για να υποστηρίξει την ανάπτυξη. Πέρα από τα μέτρα που περιγράφονται στη γραπτή ε, απάντησή μας του 2013-28 Ιουνίου, ε, έχουν γίνει κάποια βήματα, έχουν ληφθεί μέτρα πριν από 15 μέρες, 13 πρώτου, έγινε μια ανακοίνωση για την ευελιξία για να μπορεί ο καθής να χρησιμοποιεί όλες τις δυνατότητες, οικονομική κύκλη, δημόσιες επενδύσεις, διαστατικές μεταρρυθμίσεις ε, στην δημοσιονομική εποπτεία. Η ανακοίνωση αυτή γενικότερα εγγράφεται στο πλαίσιο του σχεδίου Juncker που προβλέπει επενδυτικό σχέσιο μαζί με ε, δημοσιονομική ευθύνη και προσαρμογή για να επανέλθει η ανάπτυξη. Δεν θα εγκαταλειφθεί κάθε είδους ε, δημοσιονομική εποπτεία, αλλά θα πρέπει να συνοδεύεται με διαρθρωτικά μέτρα, επενδυτικά μέτρα, με υποστήριξη της ανάπτυξης και καλύτερη εκτίμηση των κοινωνικών επιπτώσεων στις μεταρρυθμίσεις. Αυτό άλλωστε προτίθεται να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα επόμενα έτη. Συμπέρασμα. Κατόπιν των ανωτέρων η Επιτροπή δεν μπορεί να δώσει συνέχεια στο αίτημα της αναφέρουσας, η οποία ζητεί απλούστατα την κατάργηση και την εγκατάλειψη της συνθήκης για τη σταθερότητα, το συντονισμό και τη διακυβέρνηση. Ευχαριστώ. Ανοίγει η συζήτηση, ε, με σύντομη συζήτηση από αυτού. Όχι, όχι με αναφέροντες, τα μέλη της Επιτροπής έχουν το δικαίωμα να μιλήσουν. Δεν θέλει κανείς το λόγο. Λοιπόν, προτείνω να κλείσουμε αυτή την αναφορά. Την κλείνει. Είναι, είναι καλή ενδιαφέρουσα αναφορά, μάθαμε ε, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε πολύ καλά τη δουλειά της και προχωρούμε στην επόμενη. Συμφωνείτε, μπορούμε να προχωρήσουμε ωραία. Επόμενη αναφορά. Η Ισάκ η Ισπανική Ιθαγένεια, σχετικά με το πρόγραμμα μεταρρύθμιση που ζητεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εφαρμοστεί στην Ισπανία. Αυτή είναι μια αναφορά που ήταν στον κατάλογο Β και ζήτησαν δύο μέλη της Επιτροπής να μεταφερθεί στον κατάλογο Α. Η κυρία Βαλίνα και η κυρία Αλβιόλ. Χαίρομαι που παρευρίσκεται η κυρία Αλβιόλ. Θα σας δώσω το λόγο μόλις ακούσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την απάντησή της. Σύντομα, παρακαλώ. Λουίς Γκαρθία Λομπαρντέρο, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο αναφέρον διατύπωσε δύο ερωτήματα. Πρώτα, ποιο είναι το, το νομικό καθεστώς για τη συστάσεις αναχώρα και συγκεκριμένα για την Ισπανία που τις έγιναν το 2013. Και αυτές οι συστάσεις είναι νομικά δεσμευτικές ή όχι. Δεύτερη ερώτηση. Εάν οι απόψεις πολιτικών από άλλα κράτη-μέλη σχετικά με τις πολιτικές φορολογίας και αγοράς θα έπρεπε να θεωρούνται άμεση παρέμβαση στα εσωτερικά της χώρας. Η απάντηση έχει ως εξής. Στην πρώτη ερώτηση έχω να πω ότι οι συστάσεις αναχώρα δεν είναι νομικά δεσμευτικές. Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιστεύει ότι είναι προς το συμφέρον των κρατών μελών να εφαρμόσουν τις ε, συστάσεις αναχώρα που τους γίνονται, διότι η εφαρμογή τους θα βοηθήσει να αυξηθεί η ανάπτυξη, να διατηρηθούν υγιή δημόσια οικονομικά και να διορθωθεί το υπερβολικό ε, κρατικό έλλειμμα και οι μακροοικονομικές ανισορροπίες μέσω των ε, οποίων θα οδηγούνταν σε κυρώσεις το συγκεκριμένο κράτος απόψεις ενός κράτους, να πω, για τα οικονομικά ενός άλλου κράτους μέλους δεν ε, υπόκειται σε κάποια σχετική ευρωπαϊκή νομοθεσία. Είναι ε, μια ενέργεια που μπορεί να γίνει από κά, οποιοδήποτε κράτος μέλος. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ο λόγος τώρα στην κυρία Αλβιόλ. Υποθέτω πως θα θέλετε να μιλήσετε. Ναι, ευχαριστώ. Απίστευτα μου φαίνονται αυτά τα πράγματα που ακούμε. Αυτοί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τολμούν, έχουν το θράσος να λένε ότι αυτά τα μέτρα που μας συνέστησαν, βλέπε μας επέβαλαν, ε, θα βοηθήσουν για να διατηρήσουμε, λέει, και την ανάπτυξη και την απασχόληση και ε, υγιή δημόσια οικονομικά. Άκουσαν, άκουσαν τέτοια ώρα, τέτοια λόγια. Τι ακούμε εδώ πέρα μέσα και τι γράφουν σε χαρτί. Ε, ε, λόγω αυτών των συστάσεων για τις μεταρρυθμίσεις που έπρεπε να κάνει η Ισπανία το 2013, χάρη σε τέτοιες συστάσεις και άλλες προηγούμενες, οι, οι κυβερνήσεις μας ε, που είναι υπόδουλες, πρώτα ο Σαπατέρο και μετά ο Ραχώη, έκαναν διάφορες μεταρρυθμίσεις, στις συντάξεις, στην εργασία, αύξησαν το ΦΠΑ, ε, περικοπή στην υγεία, στην παιδεία, ε, στους φόρους, μέχρι και το Σύνταγμα τροποποίησαν ε, για να είναι πρώτος στόχος η αποπληρωμή του χρέους. Το βάλαμε στο Σύνταγμα. Και ε, αυτή τη στιγμή στο Ισπανικό κράτος έχουμε 24% ανεργία, 53% και μισό στους νέους. Έχουμε πάνω από ένα εκατομμύριο οικογένειες με παιδιά, όπου όλοι οι ενήλικες είναι στην ανεργία, 30% του πληθυσμού κινδυνεύει από τη φτώχεια 2.600.000 παιδιά κάτω από το κατόφλι της φτώχειας, 7 εκατομμύρια άνθρωποι ενεργειακή φτώχεια και δημόσιο χρέος που έχει ξεπεράσει το 14, 98 του ΟΕΠ και το 15 είναι 101,2% του ΟΕΠ. Ωραία όλα αυτά. Και έρχεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μας λέει ότι τα μέτρα αυτά ήταν για να αυξηθεί η ανάπτυξη και η απασχόληση. Όπως σας είπα προηγουμένως, δεν πιστεύω στα αυτιά μου αυτά που ακούω και αυτά που συνεχίζουν να ισχυρίζονται από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν ήθελα να τα πω γιατί διαβάζοντας την απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν πίστευα στα μάτια μου. Θα συνεχίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ακολουθεί αυτή τη γραμμή της λιτότητας που μας οδήγησε σε αυτά τα δραματικά στοιχεία ε, φτώχειας ε, μιζέριας και ανεργίας. Και για τη συγκεκριμένη αναφορά έχουμε συζητήσει πολλές αναφορές απόψε για τη λιτότητα και για τέτοιου είδους συστάσεις και θα ήταν θετικό τουλάχιστον να γίνει μια έκθεση από πλευράς Επιτροπής μας ή με κάποιο τρόπο να δούμε πώς οι πολιτικές της Τρόικα έχουν επηρεάσει την κατάσταση στο Ισπανικό κράτος. Και τι σημαίνει αυτό από πλευράς, ε, από τη σκοπιά της ανισότητας και της φτώχειας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Πείτε, ζήτησε το λόγο. Ναι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δίκιο όσο περίεργο και αν ακούγεται αυτό. Πολλές φορές είναι έτσι τα πράγματα συγκεντρώνονται οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, όπως έγινε και αποφάσισαν για ένα κοινό νόμισμα, το ευρώ στην προκειμένη περίπτωση. Και ανέφεραν ορισμένα βασικά κριτήρια στα οποία, τα οποία πρέπει να τηρούνται από όλους τους συμμετέχοντες σε αυτό το κοινό νόμισμα. Και όταν καμιά φορά τα πράγματα δεν πάνε καλά, συνήθως έχουν συμφωνηθεί από πριν οι λύσεις και οι επόμενες ενέργειες. Και αυτό ίσως πολλοί το ξεχνάνε. Και η Γερμανία έτσι και ήταν και η πρώτη που παραβίασε τις ε, συμφωνίες αυτές. Και πολλές φορές υπήρξαν χρήματα τα οποία δόθηκαν για λάθος ε, σκοπούς και πάλι δεν αντέδρασε κανένας. Αυτό όμως που χρειάζεται είναι διάλογος. Ο διάλογος είναι ε, πιο σημαντικός από ποτέ. Διότι πρέπει να δούμε μέσω του διαλόγου πώς θα συνεχίσουμε και πώς θα διορθώσουμε τα λάθη μας και στον χώρο της υπαίθρου και τι θα γίνει στην περίπτωση της χρηματοδότησης για την Ελλάδα, τι έγινε σε αυτή την περίπτωση, γιατί η κυβέρνηση της Ελλάδας δεν ήταν σε θέση να παρουσιάσει ένα ε, ολοκληρωμένο πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της, ε, του προβλήματος ανάπτυξης και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Πρέπει να υποχρεώσουμε τα κράτη να διεξάγουν αυτό το διάλογο. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη και επίσης να πω ότι για μένα η αναφορά αυτή θα έπρεπε να κλείσει και να διοργανώσουμε ενδεχομένω μία εκδήλωση στην οποία θα συζητήσουμε το θέμα. Πρέπει να προσέξουμε γενικά, να μην πετάξουμε το μωρό μαζί με τα νερά της σκάφης. Και φυσικά ο κόσμος δεν μπορεί να αλλάξει από μόνος του και να γίνουν ξαφνικά όλα καλά. Φυσικά πρέπει να λυθούν τα προβλήματα, αυτό όμως δεν θα γίνει με κατηγορίες. Και πάλι πιστεύω πως αρμοδιότητα εδώ έχουν τα κράτη-μέλη και το Συμβούλιο και όχι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ. Σολεδάδ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ θέλω να πω το εξής. Εν μέρη συμφωνώ με τα όσα είπε ε, η συνάδελφος Αλμπιόλ. Είναι πολιτική αυτή η συζήτηση που κάνουμε. Είμαστε στην πολιτική αναφορών όμως και θα πρέπει να ξέρουμε μέχρι που φτάνει ε, μία συζήτηση και που αρχίζει η άλλη. Δεν συμφωνούμε όλοι με τον τρόπο που αντιμετωπίζεται και επιβάλλεται η λιτότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά θέλω να πω το εξή εγώ. Αυτή η συζήτηση που αρχίσαμε τώρα, που ανοίξαμε, είναι πολιτική. Εγώ δεν πρόκειται να υπερασπιστώ τις πολιτικές που έχουν υιοθετηθεί σε καμία περίπτωση, αλλά η αναφορά από μόνη της θα πρέπει να επικεντρώνεται ε, σε συγκεκριμένα πράγματα. Εγώ θα ρωτούσα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κάνει ερώτηση, επηρεάζεται η πολιτική ε, που ακολουθούν τα κράτη-μέλη τα ανθρώπινα δικαιώματα και αν υπάρχει κάτι που μπορεί να θεωρείται ότι είναι εις βάρος κατά των συνθήκων και τις παραβιάζει ε, στο σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης να το πούμε και αυτό. Τι εννοώ. Αυτό που χρειάζεται τώρα είναι να δείξουμε τι ζητάμε, πού θέλουμε να πάμε και ε, για ποιο θέμα θέλουμε να κάνουμε έκθεση. Γιατί δεν μπορούμε τώρα ο ένας να τα ρίχνει στον άλλον, ποιος φταίει, οι σοσιαλιστές, το ΕΛΚ, τα κάνανε όλα ε, άσχημα και οι αναφερόμενοι καλοί και άγιοι. Και... Τελικά θεωρώ ότι είναι σημαντικό να μιλούμε για την διαφάνεια όσον αφορά τις αποφάσεις της Τρόικας και του Συμβουλίου γι' αυτό. Οπότε θέλουμε ένα εργαλείο για να μπορέσουμε να αλλάξουμε την ε, πολιτική για αυτή την πλειοψηφία στη που επέβαλε την λιτότητα θέλουμε κάποιες μεταρρυθμίσεις σε αυτές τις χώρες γιατί η πολιτική αυτή ήταν άστοχη. Άρα θα πρέπει εδώ να επικεντρωθεί η συζήτηση. Δούμε πώς μπορεί να γίνει κάποια έκθεση όσον αφορά πώς παραβλάφτηκαν τα ανθρώπινα δικαιώματα από αυτή την πολιτική για το Σύμφωνο Σταθερότητας που δεν έχει τηρηθεί κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό όσον αφορά την και σοβαρό όσον αφορά τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ρώσα, ευχαριστώ. Ε, οπότε θα πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε σε σχέση με τις εκλογές του Μαρτίου, του Μαΐου, του Σεπτεμβρίου, του Οκτωβρίου. Όλες αυτές οι εκλογές ε, γιατί ήταν πάρα πολύ άδικη αυτή η κυβέρνηση ή πάρα πολύ άδικη αυτή η επίθεση σε Θαπατέρο και σε Ραχώρη. Αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να μην ε, συζητήσουμε αυτά τα θέματα, να σεβαστούμε την Επιτροπή των Αναφορών, μειωθεί η απεργία, να μειωθεί το έλλειμμα. Κυρία Ολμπιόλ. Αυτά μπορεί να τα λέτε σε οποιοδήποτε παράθυρο της τηλεόρασης. Να μην κάνουμε τη συζήτηση της αναφοράς προεκλογική συγκέντρωση. Ζητήθηκαν μεταρρυθμίσεις. Και ζητήθηκαν επίσης πάρα πολλές θυσίες από τον κόσμο αυτό έχει σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η Επιτροπή προέβησε κάποιε συστάσεις. Για μένα ήταν θετικέ. Και όπω είπε και ο Πίτερ, πήρε με τη σειρά του Συμβούλιο κάποιες αποφάσεις. Άρα εδώ δεν έχουμε κάποια αρμοδιότητα για το θέμα. Άρα να κλείσει και αναφορά και να αφήσουμε τι ε, πολιτικέ κουβέντε για την προεδρική εκστρατεία. Η Πρόεδρος, κυρία Αλμπιόλ. Sí, gracias. No, simplemente es porque... Ευχαριστώ. Κοιτάξτε. Δύο μέρες εδώ πέρα στην Επιτροπή Αναφορών, κάθε φορά που παίρνω το λόγο, απαντάει η κυρία, ε, οι διάφοροι συνάδελφοι, λέγοντας ότι εδώ δεν είναι ο χώρος να συζητήσουμε πολιτική. Μα είναι ένα δημόσιο βήμα και μπορούμε να κάνουμε και πολιτικές συζητήσεις. Η πολιτική έχει να κάνει με τα δημόσια πράγματα. Γιατί κάθε φορά που παίρνω το λόγο μου λέτε να μην μιλάω για πολιτική. Εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην Επιτροπή Αναφορών και παντού ε, ήρθαμε για να μιλάμε για τα δημόσια πράγματα που είναι πολιτική, που είναι η δουλειά μας να ασχολούμαστε με αυτά. Μιλάω για τη φτώχεια, για την ανεργία, για την ένδια, την απόλυτη. Αυτό επηρεάζει τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών και η αφορά περί αυτού αν, ε, κατετέθη για τις συστάσεις που έκανε το Συμβούλιο προς την Ισπανία και που δύο κυβερνήσεις ήρθαν να εφαρμόσουν και οδήγησαν σε δράματα, τραγωδίες κανονικές στην κοινωνία μας. Ε, και γι' αυτό θα πρέπει να συζητήσουμε. Είναι αυτό πολιτική, ε, είναι βεβαίως. Και για εδώ ερχόμαστε να κάνουμε πολιτική, να συζητήσουμε και να ε, κάνουμε προτάσεις, πρωτοβουλίες. Αυτά, ευχαριστώ. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Έχει απολύτω δίκιο. Βεβαίω θα πρέπει να το συζητούμε, αλλά τώρα δεν μπορούμε πια να συζητήσουμε γιατί τελείωσε η ώρα μα. Ε, έληξε ο χρόνο και θα πρέπει να κλείσουμε. Οπότε και πρέπει να στραφώ ει όλου του διερμηνεί και να σα ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ήταν πολύ μακρά η συνεδρίαση και τα πήγατε πάρα πολύ καλά όπω πάντα. Αλλά πρώτα πρώτα αυτό το οποίο σα προτείνω από όσα άκουσα είναι να κλείσουμε σύμφωνα με τη σχετική πρόταση αυτήν την αναφορά. Αυτό και εγώ προτιθέμουν να κάνω. Δεν άκουσα κανεί να θέλει να παραμείνει αναφορά, επομένω ε, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να πάει από την λίστα Β στη λίστα Α. Δύο συνάδελφοι πρότειναν να κλείσει και εγώ αυτό θέλω να κάνω, εκτός αν κάποιος άλλος έχει ένσταση. Όχι, καλώς σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τώρα τελειώσαμε αυτή την τόσο τόσο μακρά ημέρα συνεδρίασης. Ευτυχώς. Ελπίζω να υπάρχουν κάποιες ε, συμπαθητικές ε, ομιλίες ε, γιατί έχουμε ε, κάτι το πάρα πάρα πολύ θλιβερό. Αναχωρεί, αποχωρεί ο Ντέιβιτ. Παρ' όλα αυτά όμως θα του εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας και ε, θα γίνει μεγάλη πλάκα. Σε δύο λεφτά θα τα πούμε έξω.